Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren. Αξιότιμοι συνάδελφοι, αγαπητοί κυρίε και κύριοι, άρχεται η ακρόαση για τη Λευκή Βίβλο για τις μεταφορές. Το συζητήσαμε το πρωί στην πρώτη συνεδρίαση. Ο Πιμ Βαντανκάπ είναι εισηγητής, επίσης παρόν. Δυστυχώς πιέζει πολύ ο χρόνος. Γι' αυτό θα ήθελα να παρακαλέσω και να θυμίσω σε όλους τους ομιλητές ότι Έχουμε μόλις έξι λεπτά για την παρουσίαση με μία εξαίρεση τον κύριο Γκρός που είναι σήμερα ο κύριος ομιλητής γιατί ε, το 2011 ήταν ο κύριος συγητής για τη Λευκή Βίβλο. Είναι πάρα πολύ φορτωμένο το πρόγραμμα άρα και ε, πολύ πιεστικός ο χρόνος. Παρακαλώ να τηρείτε όλο το χρόνο σας να προχωρήσει και η συζήτηση όμως. Αυτά... Μετά από κάθε παρουσίαση θα παίρνουν το λόγο οι σκιώδεις για δύο λεπτά και στη συνέχεια ε, όσοι άλλοι το επιθυμούν για ένα λεπτό. Βέβαια όλα αυτά θα εξαρτηθούν από τον αριθμό των ομιλητών που θα ε, ζητήσουν το λόγο. Αυτά ήταν τα διαδικαστικά μου και πάμε αμέσως στον πρώτο μας ομιλητή που είναι ο κύριος Ματιέ Γκρός γνωριζόμαστε 10 χρόνια και χαιρόμαστε πάντα όταν ξαναβρισκόμαστε. Ο κύριος Γκρός που ήταν βουλευτής παλιά και εισηγητής το 2011. Έχει το λόγο Ματιό Γκρός. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε, αγαπητέ Μιχαήλ. Γνωριζόμαστε ε, από παλιά, δεν συμφωνούσαμε πάντα, αλλά συχνά συμφωνούσαμε. Ε, σε ευχαριστώ θα προσπαθήσω να τηρήσω το χρόνο μου, το πλαίσιο και το περιθώριο που μου δίνεται και που αναλογεί και ε, ξέρω και τις παραδόσεις, αν τυχόν μακρηγορήσω υπάρχει και το σφυράκι. Τι να πεις μέσα σε 10 λεπτά. Ε, όλα τα κέντρα βάρους και όλες τις συζητήσεις να περιγράψω που είχαμε για τη Λευκή Βίβλο δεν γίνεται. Η πρόκληση είναι και παραμένει η ίδια ε, στις μεταφορές οι μεταφορές κυριαρχούν οικονομικά. Είτε πρόκειται για την απασχόληση, για το ΑΕΠ μιας χώρας, αλλά γνωρίζουμε επίσης ότι ε, το επόμενο διάστημα θα αυξηθούν ε, οι ανάγκες για μεταφορές είτε είναι επιβατικές είτε ε, αυτές είναι εμπορευματικέ μεταφορές. Ήδη φαίνεται από τώρα πόσο μεγάλη είναι η σημασία θα σας δοθούν οι διαφάνειες στη συνέχεια. Κοιτάξτε γενικά πώς έχει η ζήτηση και σε σχέση με τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Είναι σαφέστατη η, διαψήφωση, η διαπίστωση συγγνώμη, ότι είναι ε, πολύ επιβαρεμένη. Έχει μειωθεί από το 90 ε, η κατανάλωση σε άλλους τομείς, ενώ στις μεταφορές έχει αυξηθεί και συνεχίζει να αυξάνεται. Το 2011 λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτό θέλησε να το διορθώσει. Επίσης έχουν αλλάξει και τα μέσα μεταφοράς. Έχουμε μια κατανομή στα διάφορα μέσα πολύ διαφορετική. Κοιτάξτε τις εμπορευματικές μεταφορές. Οδικές 45, θαλάσσιες 36. Γνωρίζουμε, για να το πω απλά, όταν φτάσει ένα λιμάνι το εμπόρευμα, μετά ε, συνεχίζει η προώθηση οδικός. Στις επιβατικές μεταφορές είναι πιο υψηλά, 73, σχεδόν 80% δίκες. Αυτή είναι η επόμενη πρόκληση αν θέλουμε μια διαφορετική ή καλύτερη κατανομή, φιλικότερη προς το περιβάλλον. Άλλη πρόκληση που είχαμε στην τελευταία Λευκή Βίβλο κυρίως είναι αυτό ε, που λέμε κοινωνικές συνθήκες, εργασιακές συνθήκες. Έχω βρει μια μελέτη ενδιαφέρουσα από την Ιταλία που βγήκε τις τελευταίες εβδομάδες και είναι πάρα πολύ εύγλωτη. Έχει αυξηθεί η ζήτηση, αλλά αν δείτε σε ποιες χώρες αυτό έχει επιπτώσεις ε, στην απασχόληση, καταλαβαίνετε σαφέστατα ότι έχουμε να κάνουμε με ένα τομέα όπου ήταν πολύ σημαντική η δημιουργία θέσεων εργασίας, αλλά κυριαρχεί το κοινωνικό ντάμπινγκ και οι κοινωνικές συνθήκες εργασίας. Το είδαμε αυτό στις διαπιστώσεις, καθώς επίσης και τα θέματα οδικής ασφάλειας, δικαιώματα επιβατών. Ε, την επόμενη περίοδο θα ε, έχουμε τα αποτελέσματα διαφόρων εκθέσεων και συζητήσεων. Πώς φανταστήκαμε τον Ευρωπαϊκό Χώρο Μεταφορών. Και το διαπιστώσαμε εκ των υστέρων. Ένα δίκτυο των τριών μέσων μεταφοράς, μια, ένας ενιαίος ένα αέριος χώρος, ε, ξέρετε τις παλιές εκθέσεις και τις δυσκολίες Θέλουμε μεγαλύτερη επιστηποποίηση της τεχνολογίας και της επικοινωνίας, βελτίωση των υποδομών. Σύμφωνα με εκτιμήσεις μέχρι το 2030 θα μας χρειαστούν 500 δισεκατομμύρια. Ε, η διάνοιξη των αγορών ήταν κάτι που μας ενδιέφερε πάρα πολύ. Θα έρθω στη συνέχεια λαμβάνοντας υπόψη ορισμένα στοιχεία και βεβαίως οι νησιωτικές περιοχές οι ιδιαίτερα απομακρυσμένες και η έρευνα και η παραγωγή. Να δια... Έτσι στα γρήγορα να κάνουμε μια αξιολόγηση που βγήκε από τις συζητήσεις. Να δούμε από πλευράς αποτελεσματικότητας, αηφορίας, βιωσιμότητας, κοινωνικές και ασφάλεια. Βλέπουμε τι διαφορές έχουν τα διάφορα μέσα μεταφοράς. Ε, αυτό είναι μια χονδρική εκτίμηση, δεν είναι συζητήσεις σε λεπτομέρειες. Ε, αυτό όμως που μπορέσαμε να διαπιστώσουμε είναι το εξή, ότι γνωρίζουμε πόσο αποτελεσματικές είναι οι οδικές μεταφορές, αλλά εκεί είναι το συν, αλλά τα μείον είναι το περιβάλλον, οι κοινωνικές συνθήκες και η ασφάλεια. Όλα αυτά είναι αρνητικά, παρόλο που έχουμε κάνει ε, καλά έργα. Ε, στο σιδηρόδρομο έχουμε περίπου το αντίστροφο από το δρόμο. Ε, στις ε, πλωτές μεταφορές της θαλάσσιας, μάλλον έχουμε από τη μια της θαλάσσιας και από τις άλλες εσωτερικές ποτάμιες πλωτές μεταφορές, αλλά και η διαφορά είναι πάνω κάτω σαν το σιδηρόδρομο και στην και κυκλοφορία έχουμε αντιστοιχεία με τις οδικές. Τι προτάσεις κάναμε και συζητήσαμε εδώ στο Κοινοβούλιο βάσει του εγγράφου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συμφωνήσαμε ε, να υπάρχει μια αποτελεσματική ε, συνδυασμένη μεταφορά. Ξέρει ο ο πρόεδρος ότι ο κάθε εισηγητής θέλει να βάλει ένα προσωπικό τόνο στη συζήτηση και στην έκθεση. Εγώ είπα λοιπόν ότι χρειαζόμαστε όλα τα μέσα μεταφορών, δεν είναι ανταγωνιστικά, αλλά θα πρέπει να αναγνωρίσουμε τις αδυναμίες τους για να τις βελτιώσουμε και να τα χρησιμοποιούμε πιο αποδοτικά και πιο αποτελεσματικά. και μιλούσαμε για όλα τα μέσα μεταφορών και για το ποδήλατο, για τις δημόσιες συγκοινωνίες και στα ευρωπαϊκά δίκτυα το φέραμε. Είναι ένα θέμα ιδιαίτερα προσφυλές στον Πρόεδρο. Ε, βλέπετε τι προτείνουμε για το περιβάλλον. Ποια είναι η διαφορά με την πρόταση ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τα εξής δύο σημεία. Πρώτον, συμπεριλαμβάνουμε όλα ε, με ενισχυμένη προσοχή για το ποδήλατο και τις δημόσιες συγκοινωνίες και μιλήσα, τα μέσα μαζικής μεταφοράς δηλαδή και μιλήσαμε για μια ενιαία ε, κινητικότητα, ε, ασφάλεια των επιβατών και δικαιώματα αυτών είναι θέματα που απασχόλησαν και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πολύ στο παρελθόν και ακόμα και σήμερα έχουμε κάποιες προσδοκίες, ε, ας πούμε χάρτης δικαιωμάτων των επιβατών για όλα τα μέσα μεταφοράς και βεβαίως ε, να είναι και ενιαία ε, η προσφορά, τα εισιτήρια. Εγώ προέρχομαι από μία μεθόριο στο ένα τριεθνές Λουξεμβούργο, Βέλγιο, Γερμανία και έχουμε προβλήματα γιατί δεν μπορούμε διασυνοριακά και σε όλα τα μέσα μεταφοράς να έχουμε μια ενιαία αντιμετώπιση. Η απάντηση ποια είναι, να υπάρχει ένα γνήσιο δίκτυο στην Ευρώπη, το ξέραμε και από πριν αυτό, έτσι ώστε να ε, υπάρχει ένα δίκτυο μεταφορών με ε, διαδρόμους που να είναι σημαντικοί άξονες, αλλά και να υπάρχει και ένα δευτερεύον δίκτυο συμπληρωματικό με το κεντρικό δίκτυο. Αυτά που μας ενδιέφεραν ιδιαίτερα στη Λευκή Βίβλο ε, ενδιαφέρουν και τα διευρωπαϊκά δικτύα και τη χρηματοδότηση. Βλέπετε εδώ ε, τα σημαντικότερα γιατί διαπιστώσαμε ότι δεν λειτουργεί το δίκτυο διασυνοριακά, ήταν πολύ δύσκολο. Ε, υπάρχουν κάποιες στενοποί bottlenecks, δεν συνδέονται πάντα τα λιμάνια με την ενδοχώρα, ε, επίσης ε, η διαλειτουργικότητα θα πρέπει να ευνοήσει ε, το σιδηρόδρομο, τις εσωτερικές πλωτές οδούς, να φύγουν από τους αυτοκινδυνοδρόμους τα πορεύματα, όλα αυτά βέβαια σκεπτόμενοι τη μείωση του διοξιδίου του άνθρακα. Και εκτός ευρωπαϊκών δικτύων είναι τα λειτουργικά διαστήματα, τα εναέρια, FABs για τους ενιαίους εθέρες, βρισκόμαστε ακόμα σε ένα πλήρη κατακαιρματισμό του ευρωπαϊκού εναέριου χώρου που ε, απαρτίζεται από ένα άθροισμα 28 μονάδων. Επίσης θελήσαμε ένα σωστό χρηματοδοτικό μέσο και θέλω να τονίσω ότι μια χρηματοδότηση της τάξης των 30% του 100 είναι ο μέσος όρος για τις μεταφορές και είναι δύσκολο να βρεθούν κονδύλια από αλλού. Ήταν γνωστό ήδη το μέσο χρηματοδότησης διασυνδέοντας την Ευρώπη, Connecting Europe ε, Facility και 14 ε, δις για ε, το, τις μεταφορές από εκεί και 11 από το Ταμείο Συνοχής. Είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι χρειάζεται μια χρηματοδότηση από 20 μέχρι 80%. Ε, αυτά είναι από τα σημαντικότερα στοιχεία που μας ενδιέφεραν σε αυτό το τομέα. Διάνοιξη αγορών. Το είχαμε συζητήσει, αλλά με τρία συνοδευτικά μέτρα. Ποιότητα των υπηρεσιών της εκπαίδευσης και της απασχόλησης στο περιβάλλον. Δηλαδή, δεν θέλουμε να ανοίξουν οι αγορές ως αυτός σκοπός, αλλά θέλουμε να οδηγήσει σε αύξηση της ποιότητας. Ιδιαίτερα οι σιδηρόδρομοι πρέπει να ανοίξουν στην έκθεση μου θυμάμαι πάρα πολύ καλά είχα αναφέρει και τις λιμενικές υπηρεσίες, αλλά το Κοινοβούλιο, η Επιτροπή Μεταφορών, μου το έβγαλε στην ψηφοφορία και τελικά δεν υπήρχε στην έκθεση. Και φαντάζομαι ότι και η σημερινή Επιτροπή Μεταφορών έχει πρόβλημα με τις ε, λιμενικές υπηρεσίες ή το άνοιγμα των αγόρων. Μιλήσαμε για την εφηφοδιαστική, τα logistics, πώς βελτιώνεται και είναι πολύ σημαντική η χώρη αποθήκευση η ε, εκπαίδευση, μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα η την εκπαίδευση των ναυτικών, γιατί ιδιαίτερα στι οδικε μεταφορές είναι πολύ μεγάλη η προσφορά. Ε, χρόνος οδήγησης και χρόνος ανάπαυσης ε, σε σχέση με τη λευκή βίβλο. Αυτό είναι καλός τρόπος να διορθωθούν πολλά στρεβλά που επικρατούν εκεί, αλλά και στο παρελθόν ήταν πάρα πολύ καθόδηση αυτή η συζήτηση και αντιφατική. Και δεν φαντάζομαι θα ανοίξει πολύ γρήγορα. Ε, αποτελεσματική διαλειτουργικότητα, συνδυασμένε μεταφορές και χρηματοδότησή του χρειάζεται μια αντικειμενική συζήτηση για την εσωτερήκευση, τη λεγόμενη του κόστου, Που αυτό τι σημαίνει, για να το ξεκαθαρίσουμε, ότι αύριο όλα τα μέσα μεταφοράς θα μπορούν να ε, χρηματοδοτούνται όχι μόνο άμεσα, αλλά και από εσωτερήκευση, με ΣΔΙΤ ας πούμε, ε, συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Έχουμε όλα τα πρότυπα, τα ξέρουν όσοι ασχολούνται με το σιδηροδομικό πακέτο, να υπάρχει μια τυποποίηση των προτύπων και προδιαγραφών σε όλη την Ένωση. Ε, τονίζουμε τα θέματα του σιδηροδρόμου γιατί είναι αδυναμία σήμερα. 27 χώρες τα μοιράζονται αυτά, 28 σε πολλούς τομείς διασυνοριακά, δεν εννοώ μόνο τις υποδομές αλλά και την έγκριση των διαφόρων τύπων και αυτό είναι εις βάρος του σιδηροδρόμου. Αλλά αυτό το λέω ειλικρινά και προσωπικά θα πρέπει και ο ίδιος ο σιδηρόδρομος να το καθορίζει αυτό και να πείσει ο κλάδος τα κράτη-μέλη να ακολουθήσουν αυτό το δρόμο. Δεν μπορεί μόνο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έχουμε στόχους, έχουμε ημερομηνίε. Εδώ σας έχω σε αυτή τη διαφάνεια ορισμένες σημαντικές, γιατί είναι σημαντικό να μην αναλωνόμαστε σε θεωρητικές συζητήσεις. Έχουμε και προσδοκίες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Θα τα δείτε στη συνέχεια στις διαφάνειες που θα σας δοθούν και θα καταλάβετε. Και έρχομαι στις τελικές παρατηρήσεις. Είπαμε, για ποιο λόγο να έχουμε θεωρητική συζήτηση για το μέλλον ε, του, των μεταφορών πρέπει να μετράμε την πρόοδο. Ζητήσαμε λοιπόν ετήσια έκθεση πρόοδου για να δούμε ποιοι είναι οι στόχοι και πώς υλοποιούνται και να το ελέγχουμε. Επίσης, Είχαμε πει ότι για μας ε, είναι και παραμένει σημαντικό ε, πώς ελέγχεται η εφαρμογή στα κράτη-μέλη, η υλοποίηση και ενδεχομένως να πείπτει και ράβδος, κυρώσεις. Δεν θέλω να μπω σε συγκεκριμένα παραδείγματα, αλλά σήμερα βρισκόμαστε στο τέταρτο σιδηροδρομικό πακέτο. Αυτό έχει να κάνει μεταξύ άλλων το γεγονό ότι η υλοποίηση των όσων έχουν προτείνει τα τρία θεσμικά όργανα σε κάποιε χώρε είναι τόσο περιοριστική στην εκτέλεση και τόσο διαφοροποιημένη που κάθε φορά χρειάζονται νέες νομοθετικές πρωτοβουλίες για να βελτιωθούν όλα αυτά. Τα έχουμε συζητήσει και αυτά τα θέματα στο Κοινοβούλιο. Μια τελευταία μόνο παρατήρηση το Κοινοβούλιο θα πρέπει να ασχοληθεί όχι μόνο με τη δουλειά στο Συμβούλιο, αλλά και με την ίδια τη δική του. Δηλαδή με την επιτροπολογία και τις κατεξουδότηση πράξης. Γιατί σε πάρα πολλές προτάσεις γίνεται λόγος και παρένθεση. Θυμάστε όλα αυτά που συζητήσαμε για τους χρόνους ε, πτήσεις, τις ώρες πτήσεων για τους ε, κυβερνήτες των αεροσκαφών, κλείνει παρένθεση, θα πρέπει στο Κοινοβούλιο αυτά να συζητώνται με τρόπο πιο έντονο και πιο ουσιαστικό. Τέλος, εδώ κλείνει αυτός ο κύκλος, γιατί εμείς τι πρέπει, να κάνει η Επιτροπή Μεταφορών. Αύξηση της αποδοτικότητας για να μπορέσουν να αξιοποιηθούν όλα αυτά που περιμένουν οι χώρες και οι περιφέρειες στις μεταφορές επιβατών και εμπορευμάτων. Και το περιβάλλον, κάθε ε, ένα που ασχολείται με τις μεταφορές ε, τι σημαίνει αυτό και το κοινωνικό dumping και οι συνθήκες ε, απασχόλησης και ε, εργασιακές. Και για να επανέλθουμε σε αυτή τη διαφάνεια, ήταν μία από τις τελευταίες συζητήσεις που κάναμε στο Κοινοβούλιο. Για μένα η Ευρώπη δεν θα πρέπει να γίνει στη φτηνότερη τιμή, αλλά στην καλύτερη τιμή. Το τίμημα δηλαδή. Ευχαριστώ πολύ, Ματιό Εγκρός. Ε, έχει φύγει από το Κοινοβούλιο 9 μήνες, αλλά ε, δεν βλέπω διαφορά. Ο ενθουσιασμό του παραμένει εντονότατος. Ευχαριστώ που μας ήρθες και μας μίλησες. Και τώρα ακολουθούν οι παρουσιάσεις. Ε, θα δώσω το λόγο στο Μίχελ Νίλζεν από την Ένωση Διεθνών Οδικών Μεταφορών για 6 λεπτά. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε και ευχαριστώ που μας καλέσατε στην ακρόαση αυτή. Νομίζω ότι γνωρίζετε την ένωσή μας. Είναι η Διεθνής Ένωση Οδικών Μεταφορών σε πάνω από 100 χώρες στον κόσμο, 28 και από τις 28 βέβαια χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πολύ μεγάλη σημασία έχουν για την ανάπτυξη και την απασχόληση οδικές μεταφορές. 5 εκατομμύρια άνθρωποι απασχολούνται στον τομέα αυτό, 75% του όγκου μεταφέρεται οδικά, 90% της αξίας και οι άνθρωποι χρησιμοποιούν τους σιδηρόδρομους, τα τράμα, λεωφορεία κλπ. Θέλουμε να συνεχίσουμε να μπορούμε να έχουμε ανάπτυξη, οικονομική ανάπτυξη και ένα από τα πράγματα που κάναμε παλιότερα ήταν να διορθώσουμε ό,τι έλειπε. Και πολλοί ευρωβουλευτές θελήσαν να συμπεριληφθούν και τα λεωφορεία και τα πούλμαν στα μέτρα τα οποία είχαν προταθεί. Και κατέληξαν με αυτό που είναι δικιά σας η δουλειά προκειμένου να δημιουργηθεί ένα πρόγραμμα δράσης Ένωση Ένωσης 2015-2025 για να διπλασιαστεί η χρήση της συλλογική ε, γης όπου μπορούν να κυκλοφορούν επιβάτες. Χρειάζονται καινοτομίες βέβαια και σε άλλες περιπτώσεις. Πρέπει να βελτιώσουμε το περιβάλλον, την αποτελεσματικότητα και πρέπει να βγούμε από τα κλειστά πλαίσια μέσα στα οποία σκεφτόμαστε. Πρέπει να γίνουν σημαντικές αλλαγές και να δούμε συνολικά το σύστημα μεταφορών. Για μας είναι ζωτική σημασία σε αυτό, γιατί δεν μπορεί να έχουμε μια αλλαγή μόνο στα επόμενα 12 χρόνια για να περάσουμε από το ένα στο άλλο μέρος. Δεν είναι κάτι καλό για την Ευρώπη, πρέπει να τα δούμε όλα. Και για τις εμπορικές μεταφορές πρέπει να εγκαταλείψουμε την ιδέα μικρών αλλαγών κάθε τόσο, αλλά να υπάρξει ένας νέος ορισμός των εμπορικών μεταφορών. Και πρέπει να σκεφτούμε και ακόμα παραπέρα για την καινοτομία. Και για μας αυτό που έχει σημασία είναι να χρησιμοποιούμε τις ε, τεχνολογίες εχμής πιο αποτελεσματικά από ό,τι μέχρι τώρα. Να χρησιμοποιήσουμε τα κατάλληλα οχήματα και να έχουμε τις κατάλληλες υποδομές. Χρειάζεται να μπορούμε να έχουμε πληροφορίες ηλεκτρονικά μέσα από το όχημά μας που μπορούμε να παρκάρουμε, που μπορούμε να πληρώσουμε ηλεκτρονικά πάντα. Και για να σκεφτούμε και εκτός πλαισίων πρέπει να δούμε τι θα γίνει το 2030. Θα οδηγούμε τα ίδια χήματα. Μα το μόνο δεν είναι το πώς θα μεταφέρουμε ε, τις ροές μεταφορών από το ένα μέσο στο άλλο. Αυτό το είχαμε κάνει και το 1991. Αποφασίσαμε για τα ηλεκτρικά τρένα. Τώρα ίσως θα έπρεπε να σκεφτούμε κάτι διαφορετικό. Την ε, ε, διευκόλυνση συνδέοντας την Ευρώπη. Ίσως αυτό θα μπορούσε να γίνει πιο αποτελεσματικό. καινοτομία χρειάζεται σε όλες τις μορφές μεταφορών. Και να υπάρχει σύνδεση με ταξί των διαφόρων τρόπων μεταφορές. Σε αυτό θέλουμε να καταλήξουμε. Υποδομές, πρώτα απ' όλα, και χρηματοδότηση των μεταφορών για μας είναι ζωτική σημασίας και για όλα τα είδη μεταφορών. Τα κύρια μέσα χρηματοδότηση πρέπει να χρησιμοποιηθούν και για τις οδικές μεταφορές, για τα κομμάτια των δρόμων που δεν έχουν ολοκληρωθεί και συνδέουν δύο σημεία και να ληφθούν υπόψη και υποδομές για εναλλακτικέ μορφές καυσίμων που χρησιμοποιούμε. Και αυτό χρειάζεται και δεν έχει νόημα να έχουμε άλλα είδη ενέργειας αλλά να μην έχουμε τις υποδομές για να τα χρησιμοποιήσουμε έχουμε, θα έχουμε χρήματα στο μέλλον για τις υποδομές αυτές. Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα που θέτουμε όλοι στους αυτούς μας. Όλοι έχουμε πει ότι θέλουμε να συνεισφέρουμε σε κάποια πληρωμή. Θα το κάνουμε. Χρειάζεται μια μελέτη που να δείχνει τι πληρώνουμε ήδη σε σχέση με αυτά που θα έπρεπε να πληρώσουμε, δηλαδή ανάλογα με αυτά που καταναλώνουμε. Οπότε θέλουμε ένα σύστημα χρέωσης με αυτό να διέπεται από διαφάνεια. Δεν θέλουμε διπλές χρεώσεις και φυσικά πρέπει να έχουν νόημα. Να πηγαίνουν δηλαδή τα χρήματα για να εξυπηρετήσουν τα μέσα μεταφοράς από τα οποία προέρχονται. Αν θέλετε να το κάνετε αυτό με ευθύ τρόπο πρέπει να έχετε ένα σύστημα ηλεκτρονικής χρέωσης και να υπάρχουν συμβατά συστήματα μεταξύ τους. Όλα αυτά μπορούμε να τα κάνουμε στο μέλλον. Βέβαια, δεν θα γίνουν πραγματικότητα αν δεν λειτουργεί ικανοποιητικά εσωτερική αγορά. Και ο κύριο Κρό το είπε ότι δεν λειτουργεί αρκετά καλά σήμερα. Έχουμε πολλούς και διαφορετικούς κανόνες, έχουμε διαφορετικούς φορούς, φορείς, έχουμε κυρίαρχους φορείς, έχουμε διάμεσους, οι οποίοι ίσως να μην είναι καταλληλότεροι και να μην δρουν υπεύθυνα Έχουμε σαφείς κανόνες που πλήττουν τον ανταγωνισμό και σημαίνει επίσης ότι έχουμε και αθέμητο ανταγωνισμό. Ας δούμε τα ταξί. Όλοι έχετε ακούσει παραδείγματα τέτοια στα ταξί όσον αφορά τον αθέμητο ανταγωνισμό. Λένε ότι είναι καινοτομία. Δεν είναι καινοτομία. Τα ταξί έχουν κάνει διάφορες εφαρμογές, τοπικά και γενικότερες. Υπάρχουν. Το πρόβλημα με τα ταξί σήμερα θα εξακολουθούν ε, να υπάρχουν τα ταξί για να ε, βοηθούν τις υπόλοιπες μεταφορές. Αυτό πρέπει να το έχουμε υπόψη μας. Στην οργάνωσή μας πιστεύουμε ότι πρέπει να υπάρχουν οι ε, ίδιοι κανόνες για όλους. Οι κανόνες υπάρχουν για να τηρούνται και όλοι πρέπει να συμμορφώνονται. Πιστεύουμε ότι για τον τομέα των ταξί πρέπει να υπάρχει πρόσβαση για όλα τα οχήματα και τους οδηγούς. Συγχρόνως όμως ο κλάδος πρέπει να προσφέρει υπηρεσίες που να ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές των υπηρεσιών που προσφέρονται και σήμερα. Δεν πρέπει να πέσει η ποιότητα. Η πρόσβαση στην αγορά ξέρουμε ότι είναι μεγάλη. Υπάρχει το θέμα της πρόσβασης στην αγορά, των κατώτατων μισθών, κλπ. κλπ. Όλα αυτά τα θέματα ανταγωνισμού πρέπει να διορθωθούν. Θέλουμε κανόνες σαφείς και ίδιους για όλους. Θέλουμε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον όπου οι κανόνες να ισχύουν εξίσου για όλους. Και θέλουμε να υπάρχει αλυσίδα ευθύνης ανάμεσα στην ε, προμήθεια και την αλυσίδα κινητικότητας. Ό,τι καινοτομία και αν εφαρμόσουμε δεν θα αποδώσει αν δεν φροντίσουμε να ανταποκρινόμαστε κατάλληλα στις ανάγκες. Όλοι λοιπόν πρέπει να δουλέψουμε για να δημιουργήσουμε ένα αποτελεσματικό σύστημα μεταφορών για το μέλλον. Ευχαριστώ πολύ Μιχάλη Νίλσον. Επόμενος, Ζαρ Χουσέιν Χάν από την Ένωση Ευρωπαϊκών Αερομεταφορέων. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Με τα χαράς να μοιραστώ μαζί σας κάποιες από τις δικές μας παρατηρήσεις και να ευχαριστήσω και τον εισηγητή, πρώην εισηγητή. Πολύ γρήγορα πάνω αυτές τις διαφανείς, εντάξει. Εδώ είμαστε. Το προηγούμενο εισηγητή και τον τρέχοντα εισηγητή για τη δουλειά τους για τη Λευκή Βιβλό. Ήταν πολύ επικοδομητικέ οι παρατηρήσεις του για την αεροπορία την αεροπλοεία και μπορούμε να τι αξιοποιήσουμε και εδώ, στο Κοινοβούλιο, αλλά και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώ προχωρούμε. Εδώ βλέπετε για λόγου διαφάνεια ποιοι συμμετέχοντε στην ε, Ένωση των Ευρωπαϊκών Αερογραμμών. Βλέπετε του ε, μεγάλου μεταφορεί που περνάνε από τα μεγάλα κομπικά σημεία στην Ευρώπη στις μεγάλες πόλεις, αλλά έχουμε και κάποιους επιπλέον, ε, κάποιες επιπλέον εταιρείες, καθώς και μερικές περιφερειακές αντιθέτως με αυτό που κάποιοι πιστεύουν, είναι πολύ ποικιλόμορφη η συνολική εικόνα. Ανέφεραν ο κύριος Γκρός, ανέφερε ο κύριος Γκρός νωρίτερα, ότι έχουμε 9,6 εκατομμύρια πτήσεις στον ενέργο χώρο της Ευρώπης κάθε χρόνο και 7,5 εκατομμύρια επιβάτες μετακινούνται στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο, μάλιστα με ευρωπαϊκές αερογραμμές ένα πολύ μεγάλο μέρος τους. Αυτό δείχνει πολλά για την ε, διασύνδεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, Έχουμε 7,5 εκατομμύρια τόνου ε, εμπορευμάτων που μεταφέρονται από ευρωπαϊκές αερογραμμές παγκοσμίω, 25% από το σύνολο του τι συμβαίνει διεθνώ και 120 χώρες συνδέονται με την Ευρώπη μέσω των ευρωπαϊκών οργανών. Έτσι δημιουργούμε και αξία, το ανέφεραν και οι προηγούμενοι μιλητές για τις μεταφορές, 1,2 δις ημερησίως ε, προσφέρονται στο ευρωπαϊκό ΑΕΠ, ετησίως μάλλον, 1,2 την ημέρα. Ένα ε, Μία στις 40 θέσεις εργασίας στην Ευρώπη δημιουργούνται χάρη στις αερομεταφορές. Και εάν δείτε ότι το περιθώριο δυστυχώς του καθαρού κέρδους των αερο... Ε, κέρδους, του καθαρού κέρδους της αερομεταφορές δεν είναι τεράστιο, είναι 1,3 σε 1,4% όμως είναι πολλές, πολλοί κλάδοι παγκοσμίω που ξεπερνούν πολύ αυτά τα ποσοστά. Ουσιαστικά έχουμε κέρδος 2,4 ευρώ ανά επιβάτη μέσα στη χρονιά. Κάποιοι μου είπαν με τρόπο κοινικό ότι δεν είναι απλώς η τιμή ενός καφέ, αλλά σε κάποιες περιπτώσεις είναι και το 1 τρίτο της τιμής ε, ενός καφέ σε κάποια ευρωπαϊκά κράτη. Ελπίζουμε φέτος να τα πάμε καλύτερα από πέρσι, αλλά να σας πω και κάτι που μας κάνει πολύ περήφανος ως ε, κλάδο ότι έχουμε όλες αυτές τις επιτυχίες. Μιας και μιλάμε για καινοτομίες και επενδύσεις. Οι αερογραμμές που εκπροσωπούμε θα αγοράσουν 745 νέα αεροσκάφη στο προσεχές μέλλον. Η επένδυση αυτή εκπροσωπεί 73 δις ε, δολάρια, περίπου 75 δις ευρώ με τις σημερινές οτιμίες, και δεν είναι η επένδυση σημαντική αυτή καθεαυτή. Απλώ τα μισά από αυτά τα σκάφη έχουν φτιαχτεί στην Ευρώπη. Έχουν κατασκευαστεί στην Ευρώπη. Οπότε αυτό σημαίνει καινοτομία, έρευνα και επένδυση στην ευρωπαϊκή γνώση και τι θέσει εργασία και το μέλλον μα. Επίση, κάθε οικογένεια, κάθε στόλο αεροσκαφών που ε, αντικαθιστά μια προηγούμενη είναι ε, στο επίπεδο του 15 για την ηχορύπανση και την ατμοσφαιρική ρύπανση αλλά και την βιωσιμότητα και την ασφάλεια. Δεν είναι απλώ λοιπόν το χρήμα, αλλά είναι και το πλαίσιο τη βιωσιμότητα που γίνεται σεβαστό από τι αερογραμμέ. Αυτό για μα ε, παίζει καθοριστικό ρόλο. Αν δούμε τώρα το μέλλον της Ευρώπης και την ανταγωνιστικότητα των ε, αερομεταφορών, αυτό θέλουμε να συζητήσουμε εδώ μαζί. Ας ε, πάρουμε λίγο απόσταση από το δίκτυο των αερομεταφορών και ας σκεφτούμε τι γίνεται γενικότερα στην διασύνδεση των αερομεταφορών στην Ευρώπη. Οι προηγούμενοι ομιλητές το επενήχθησαν. Νομίζω ότι συμβαδίζουμε πλήρως, εάν δείτε ποιες είναι απαιτήσει του κλάδου μας με τον προηγούμενο ομιλητή. Δηλαδή, εφόσον εκπροσωπούμε αερομεταφορέ σε διεθνέ επίπεδο, πρέπει να καταλάβουμε ότι η Ευρώπη δεν θα μπορεί πλέον να κάνει τα πράγματα μόνη τη απομονωμένα. Είμαστε μέρο ενό διεθνού δικτύου και έτσι θα πρέπει να σκεφτόμαστε. Υπάρχουν κάποια παραδείγματα στο Ευρωπαϊκό ευρωπαϊκό νομοθετικό πρόσφατο παρελθόν που μας δυσκολεύουν κάπως. Χρειάζεται λοιπόν ευφιέστερη ε, νομοθεσία. Και νομίζω όλοι σήμερα το απόγευμα θα πούμε ότι χρειαζόμαστε λιγότερο άχθος και πιο αποτελεσματική νομοθεσία με σωστή υλοποίηση. Ας υλοποιήσουμε πρώτα την νομοθεσία που ήδη έχουμε εγκρίνει για να έχουμε ισότιμους κανόνες ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά. Πρέπει να μειωθούν ε, το άχθος για, την, ε, για τους φόρου τους φόρους, για όλες τις Διαστάσει του θέματο. Αυτό το λέω και βγαίνω των μεταφορών γενικότερα, αλλά και ιδίω εκ των αερομεταφορών. Ω προ του ίσους κανόνε του παιχνιδιού, λοιπόν, είναι σημαντικό να γίνει αυτή η συζήτηση για τα μέσα μεταφοράς που χρησιμοποιούμε, γιατί αν δούμε τι γίνεται στο παγκόσμιο σκηνικό, ένα από τα πλεονεκτήματα τη Ευρώπη είναι ότι ω προ την ανταγωνιστικότητα Έχουμε το πιο έγκριθμο σύστημα μεταφορών παγκοσμίω. Είμαστε πολύ καλύτεροι από τι ΗΠΑ, από τη Μέση Ανατολή και από την Απανατολή. Δεν είμαστε πάρα πολύ καλοί στην βελτιστοποίηση του συστήματο. Πρέπει να βρούμε λοιπόν τρόπου να μεγιστοποιήσουμε ε, αυτά τα μεμονωμένα συστήματα που έχουμε για να είμαστε πιο ανταγωνιστικοί. Με κοιτάζει ο Προεδρο και με το δίκιο του. Έχω περάσει τα 6 λεπτά κατά 29 δευτερόλεπτα. Κλείνω εδώ. Ευχαριστώ. Thank you very much as well. Ευχαριστώ πολύ. Λίμπορ Λόχμαν, ο επόμενος, από πλευράς σιδηροδρόμων. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Controller. Thank you. Okay. Thank you very much. So... Σχετικά με τη Λευκή Βίβλο, πού βρισκόμαστε και πού θα έπρεπε να βρισκόμαστε και πώς εφαρμόζουμε τα μέσα τα οποία προβλέπονται στη Λευκή Βίβλο. Από πλευρά σιδηροδρόμων, λοιπόν, έχουμε σωστές πολιτικές προτεραιότητες. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να πετύχουμε τις προτεραιότητες αυτές. Λαμβάνοντας υπόψη μας την μείωση ε, των ε, αερίων του θερμοκηπίου, σε σχέση με το 1990. Πρόταση λοιπόν για δεσμευτικούς στόχους όσον αφορά την μείωση των εκπομπών αυτών διοξιδίου του άνθρακα. Δεσμευτικό. Δεύτερον, όσον αφορά πάντα τα αέρια του θερμοκηπίου, έχουν προταθεί λύσεις, το είπε και ο κύριος Γκρός. Έχουμε το μέσον λοιπόν για να το πετύχουμε, για να κάνουμε αυτό που θέλουμε. Και μετά από αυτό που εξήγησε ο κύριος Γκρός πριν από λίγο, όσον αφορά την απόδοση των σιδηροδρόμων, ναι, μπορούμε να βελτιωθούμε περισσότερο και όχι μόνο με το πακέτο αλλά και με την καινοτομία, αλλά πρώτα απ' όλα πρέπει να δούμε τις στατιστικές και την εξέλιξη η οποία θα μας οδηγήσει να έχουμε σιδηροδρόμους που είναι όλο και περισσότερο φιλικοί προς το περιβάλλον και που θα λάβουν υπόψη τους και τον συνδυασμό της πολυτροπικές μεταφορές δηλαδή. Η σειρόδρομοι λοιπόν είναι μέρος της λύσης και είναι μέρος της λύσης και για την μείωση κατανάλωσης πετρελαίου. Άρα ας κάνουμε αυτό που πρέπει για να το πετύχουμε. Να χρησιμοποιήσουμε ηλεκτρικά οχήματα. Η λύση είναι πως οι δημόσιες μεταφορές θα είναι ηλεκτρικές. Όχι να μειώσουμε την κατανάλωση μόνο, αλλά να αλλάξουμε και την ενέργεια που χρησιμοποιούμε. Απασχόληση τώρα. Οι σιδηρόδρομοι προσφέρουν, ε, είναι από τους κλάδους που προσφέρει τις περισσότερες θέσεις απασχόλησης και άμεσα και έμεσα. 1,1% του Ευρωπαϊκού ΕΠ είναι η σιδηρόδρομοι. Αυτό πρέπει να το αντιληφθούμε και να το συνδυάσουμε και με τα υπόλοιπα είδη μεταφοράς, σε πολυτροπικές μεταφορές. Η πρόταση λοιπόν είναι, αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε περισσότερο την εξέλιξη αυτή, πρέπει να έχουμε και τις κατάλληλες κοινωνικές συνθήκες. Νομίζω ότι συμφωνούμε εδώ με τους συναδέλφους ότι πρέπει όντως να ισχύουν οι ίδιοι κανόνες για όλους. Επιπλέον αυτό το οποίο πρέπει να πετύχουμε για να έχουμε αυτούς τους ίδιους κανόνες είναι το θέμα των τιμών και της πολιτικής που ισχύει. Ας δούμε τα νούμερα. Ας τα λάβουμε υπόψη μας και ας τα βάλουμε πάνω στο τραπέζι. Οι σιδηρόδρομοι είναι οι μόνοι που είναι υποχρεωμένοι να πληρώνουν βάσει της απόστασης. Και δεν είναι μόνο η χρέωση βάση της ε, απόστασης, είναι και θέμα κόστους. Να εσωτερικεύσουμε λοιπόν το εξωτερικό κόστος. Συμφωνούμε λοιπόν απόλυτα ότι πρέπει να εντοπίσουμε τις δυσκολίες και αυτά που μπορούμε να κάνουμε για να αποφασίσουμε ότι τα χρήματα τα οποία θα εισπραχτούν να χρησιμοποιηθούν για την ανανέωση του τομέα. Και αν θέλουμε πιο αποτελεσματικές μεταφορές στο μέλλον, μεταφορές που να καταστρέφουν λιγότερο το περιβάλλον και να είναι φιλικές και προς την κοινωνία, πρέπει να αναπτύξουμε τις υποδομές. Και οι υποδομές πρέπει να αναπτυχθούν για εκείνα τα είδη μεταφοράς που είναι πιο βιώσιμα. Δεν πρόκειται μόνο να αλλάξουμε, που εμείς του σιδηρόδρομο το θέλουμε να περάσουμε τις οδικέ ας πούμε στις ε, σιδηροδρομικές μεταφορές, αλλά θέλουμε να υπάρχει χρηματοδότηση επαρκής για τις υποδομές εκείνες που εξυπηρετούν καλύτερα το κοινό. Λαμβάνοντα υπόψη ω κριτήριο βέβαια το περιβάλλον σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό για να χρηματοδοτηθούν κατάλληλα προγράμματα. Συνεπώς, πώς θα χρηματοδοτήσουμε καλύτερα τις υποδομές, πώς θα ακολουθήσουμε μια ρυθμιστική πολιτική η οποία θα προσφέρει τους ίδιους κανόνες για όλα τα είδη μεταφορών και πώς θα έχουμε μια καλύτερη πολιτική που θα βελτιώνει την κατάσταση για την κοινωνία. Πώς θα χρησιμοποιήσουμε περισσότερο τον ηλεκτρισμό για τις ε, δημόσιες μεταφορές. Έχουμε το 80% αλλά πρέπει να το βελτιώσουμε ακόμα περισσότερο. Και να έχουμε και δεσμευτικούς στόχους όσον αφορά την μείωση των αερίων του θερμοκηπίου. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Το επόμενο διαμιλήτρια κάνει τη ΣΥΕΠΑ, για, ε, ε, είναι Διευθύντρια των Εσωτερικών Πλωτών Μεταφορών στην Ευρώπη. Ευχαριστώ κύριε Κράμερ και ευχαριστώ κύριε Φαντεγκάμπ που οργανώσατε αυτή την ακρόαση. Θέλουμε να μοιραστούμε μαζί σας τις δικές μας παρατηρήσεις. Είμαστε μια πλατφόρμα για την διαχείριση των ιστορικών πλωτών μεταφορών και την προώθηση του σχετικού δικτύου. Όταν δούμε ποιοι είναι οι βασικοί στόχοι που μας αφορούν, βλέπουμε ότι είναι κυρίως η ένταση χρήσης άνθρακα του μεταφορές. Αυτό πρέπει να πάψει. Υπάρχει και άλλο ένα θέμα που είναι εξίσου σημαντικό και νομίζουμε ότι θα πρέπει να μας οδηγήσει σε έναν ευθύ συνδυασμό, δηλαδή οι μεταφορές να γίνουν ένα μέσο ώστε να ενισχυθούν η βιομηχανία και το εμπόριο. Όπως έχουν διαμορφωθεί τα πράγματα με τις κυκλοφοριακές συμφορήσεις, το κόστος είναι τεράστιο και αυξάνεται διαρκώς. Αν δείτε τι γίνεται με, τα, με τους λιμένες, τους θαλάσσιους λιμένες, 90% ε, του εμπορίου μας θα μπορούσε να περνάει όλα από εκεί και να τετραπλασιαστεί το σημερινό ποσοστό. τα αστικά κέντρα όμως δεν είναι έτοιμα για αυτού του είδους την αύξηση. Εάν δείτε τη Λευκή, Βίβλος, τη Λευκή Βίβλο του 2011 υπάρχει ο στόχος της βελτίωσης αποδοτικότητας του κάθε μέσου μεταφοράς, αυτό είναι πολύ σημαντικό και καλούμε το Κοινοβούλιο να στηρίξει με την γοργή υλοποίηση του Ναϊάδες, των Ναϊάδων δηλαδή, το ε, όλο πρόγραμμα, τον στόχο αυτό. Θέλουμε να υπάρξει καλή υλοποίηση, αλλά δεν θα αρκέσει αυτό. Χρειάζεται να αποφύγουμε και την συμφόρηση που διαρκώς αυξάνεται. Μπορεί να εκπλαγείτε εάν δείτε αυτό το τεχνητό όριο των 300 χιλιόμετρων αλλά πραγματικά θα πρέπει να περάσουμε στο σιδηρόδρομο και τις πλωτές οδούς για τις αποστάσεις άνω των 300 χιλιόμετρων. Συμφόρηση υπάρχει και στους λιμένες λοιπόν και στις αστικές περιοχές. Εάν θέλουμε να να μπορούν να χρησιμοποιήσουν ε, τις οδικές μεταφορές όσοι δεν μπορούν να τις σταματήσουν θα πρέπει να απαλλάξουμε τους αυτοκινητοδρόμους από τη συμφόρηση και να υπάρχει δυνατότητα χρήσης πολλών μέσων μεταφοράς όπου αυτό είναι απαραίτητο. Επίσης, με μεγάλη θλίψη βλέπουμε ότι όπου έχουμε μια ε, πολιτική για τον συνδυασμό μέσων, όπως το Connecting Group Facility, με τρία χρόνια διαπραγματεύσεις στην πλάτη του, εδώ έχουμε τουλάχιστον 20% περικοπές, δυστυχώς, ε, προς το ΕΦΣΥ, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στατικών Επενδύσεων. Δεν είμαστε κατά του ΕΦΣΥ βεβαίως, αλλά πιστεύουμε ότι υπάρχουν και άλλοι ευθύς τρόποι χρηματοδότηση του ΕΦΣΥ. Αυτό που τώρα έχουμε είναι ένας, ένα κατακαιρματισμένο σύστημα μεταφορών και ουσιαστικά πίεση ασκείται στη βάση του συστήματος με μεγάλο κόστος λόγω της συμφόρησης και της χρήσης του άνθρακα. Αυτό που χρειαζόμαστε, δεν θα σας εκπλήξει, είναι ε, χαμηλότερα επίπεδα συμφόρησης, με χαμηλότερη χρήση άνθρακα και με ανταγωνιστικό κόστος προφανώς. Για να το πετύχουμε αυτό χρειάζεται να προωθηθεί η ψηφιακή ατζέντα μας, και όχι μόνο να έχουμε το συνδυασμό των πολλών διαφορετικών μέσων μεταφοράς, αυτό μας απασχολεί τώρα, με ευθύ τρόπο, αλλά να είναι πραγματικά η ποικιλία των μέσων το σύστημα που θα επικρατήσει, ώστε να μπορέσει και η κινητικότητα να τονωθεί. Το ίδιο και για τα εμπορεύματα. Αυτά τα εμπορεύματα πρέπει να προωθηθούν με πολλούς ε, διαφορετικούς τρόπους, με άλλα μέσα ε, μεταφοράς. Το Ρότερνταμ, η Αμβέρσα, ε, η Μασαλία, η Κωνσταντζα είναι τα λιμάνια από τα οποία θα πρέπει να έχουμε συνδυασμό μέσων με οδικό τρόπο λόγου χάρη και να, προωθηθεί και το, να προωθηθούν έτσι και οι όγκοι των εμπορευμάτων. Τότε μειώνεται το κόστος της μεταφοράς και μπορούμε να περάσουμε σε ένα συνεργατικό ε, μοντέλο ε, κατανομής των δυνατοτήτων. Κάτι που για την ώρα δεν το έχουμε με το κατακαιρματισμένο σύστημα μεταφορών. Εδώ μπορεί να μας βοηθήσουν οι νομοθέτες ώστε να ευθογραμμιστούν οι προτεγραφές των διαφόρων ε, ε, λειτουργόντων στην αγορά και να υπάρξει και προστασία του περιβάλλοντος με τις κατάλληλες υποδομές βεβαίως και αυτό είναι πολύ σημαντικό για τον πυλώνα της ανάπτυξης του, της ποικιλία των μέσων μεταφοράς. Το ίδιο και για τους λιμένες, τους θαλάσσιους ή τους εσωτερικούς. Εκεί θα πρέπει να υπάρχει άμεση πρόσβαση για τους μεταφορείς, ε, για τα πολλά διαφορετικά μέσα και βεβαίως ο συνδυασμός, το bundling είναι πολύ σημαντικό για να μπορέσει να τονωθεί η οικονομία γύρω από τους λιμένες μας. Δεν θέλουμε λιμένες μόνο για την διέλευση. Δεν θέλουμε να είναι γκαράζ και χωρίς τάθμευσης για το εμπόρευμα. Θέλουμε να υπάρχει προστεθέμενη αξία και αυτή να ε, δημιουργείται διαρκώς ώστε να έχουμε και θέσεις εργασίας. Βιωσιμότητα λοιπόν θέλουμε στην ενίσχυση των λιμένων για να πάυσουν οι δυσκολίε. Και για την καινοτομία που είναι το τελευταίο αλλά όχι το λιγότερο σημαντικό. Δεν είναι απλό να έχουμε καινοτομία στι μεταφορέ, ιδίω ένα σύστημα με χαμηλέ τιμέ και μικρή διάρκεια συμβάσει. Αν θέλουμε έντονη καινοτομία, στην πρασίνισμα λόγου χάρη ή την ε, διοργάνωση της ποικιλία των μέσων, θα πρέπει να είμαστε πολύ καινοτόμοι και να αναλάβει κάποιο το επιπλέον κόστος. Ε, θα πρέπει να σταματήσουμε όμως να τιμωρούμε όσους ακριβώς προσπαθούν να παράγουν περισσότερη καινοτομία στο πρασίνισμα και την διοργάνωση της ποικιλία των μέσων μεταφοράς. Κάτι που για την ώρα δεν ισχύει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Επόμενος ομιλητής και τελευταίος για αυτό το πάνελ, Χέρμα Μάγε ε, είναι CEO της ΕΡΤΙΚΟ για ευφυή e συστήματα μεταφορών στην Ευρώπη. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Κράμερ, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση σε αυτή τη σημαντική ακρόαση. Μου δίνετε ένα τηλεχειριστήριο παρακαλώ. That's Πρώτα χρειάζεται τη τεχνολογία, μετά ο χρήστης και αν ε, συνδυάζονται καλά και κάποιο αποτέλεσμα. Ε, θα σας πω τι είναι τα FEE συστήματα μεταφορών. Ε, ε, για να υπάρχει μια ουσιαστική ολοκλήρωση των διαφόρων μέσων μεταφορών για να ε, έχουμε ένα ολοκληρωμένο σύστημα που να εξυπηρετεί και τους επιβάτες και τις εταιρείες οδιαστικής. Βλέπετε εμείς πόσους εταίρους έχουμε. Πάνω από 100 είναι οι διάφορες εταιρείες από τους διάφορους κλάδους που είναι απαραίτητοι για να γίνουν ε, οι έξυπνες μεταφορές στην Ευρώπη πραγματικότητα. Εδώ ε, πραγματικά η εστίαση είναι στη συνεργασία για να αναπτυχθεί το σύστημα και να εξελιχθεί. 19 ευρωπαϊκά κράτη-μέλη συμμετέχουν διότι οι υποδομές ε, είναι ένα κεκτημένο που πρέπει να έχουν τα κράτη-μέλη για να συμμετέχουν. Τι είναι λοιπόν τα ΕΦΗ συστήματα μεταφορών. Με δύο λόγια, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η συλλογή, η ανταλλαγή, η διαχείριση στοιχείων και δεδομένων έτσι ώστε να παρέχονται υπηρεσίες και να είναι μεταφορές πιο ασφαλείς, πιο αποτελεσματικές και τελικά πιο άνετες. Τριών ειδών υπηρεσίες ε, παρέχουμε. Το ένα είναι ενημέρωση, ας πούμε τι ώρα περνάει το επόμενο λεωφορείο. Ε, είναι διευκόλυνση, δηλαδή να μπορείτε αν θέλετε να κλείσετε το εισιτήριό σας, να κάνετε και ηλεκτρονική πληρωμή αγοράζοντας το εισιτήριο και αυτοματοποίηση. Δηλαδή χρησιμοποιούμε ήδη την πληροφορία για να αυτοματοποιήσουμε την ε, οδήγηση ας πούμε οχημάτων. θα αλλάξει πραγματικά την κατάσταση και το παιχνίδι αυτή ε, η ε, πρόοδος με πολλούς τρόπους. Πρώτον, στη διαχείριση των μεταφορών, γιατί στοιχεία υπάρχουν και δεδομένα, τα οποία όμως δεν ανταλλάσσουμε, δεν μοιραζόμαστε και να είναι καλύτερη η διαχείριση έτσι των μεταφορών ε, μέσω της γνώσης. Η πληροφορία και η γνώση είναι πολύτιμη για να παρέχεις καλύτερες ε, υπηρεσίες στον κόσμο. Το ίδιο ισχύει και για τα ηλεκτροκίνητα οχήματα, διότι αυτό μπορεί να βοηθήσει τον οδηγό ενός τέτοιου οχήματος να δει πού είναι ο επόμενος σταθμός για να ε, φορτίσει το αυτοκίνητο, ε, να κάνει ε, όλες τις πληρωμές του ηλεκτρονικά. Γι' αυτό χρειάζεται μια πανευρωπαϊκή λύση, αλλιώς δεν πρόκειται να προχωρήσει αυτή η υπόθεση των ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων. Τα ίδια ισχύουν και για την εφοδιαστική, για την αυτοματοποίηση και τις υπηρεσίες μπορεί αυτό να βοηθήσει σε πιο αποτελεσματική οδήγηση, πιο άνετη και πιο ασφαλή. Ήδη από σήμερα τα οχήματα που έχουν και κάμερες μέσα συλλέγουν τόσο πολλά στοιχεία και δεδομένα και αν μπορεί κανείς αυτό να τα ε, μοιραστεί με άλλους οδηγούς είναι πιο ασφαλής η οδήγηση ε, και αυτό μπορεί να μεταφερθεί με αυτοματοποιημένο τρόπο για να βοηθήσει να ε, αυξηθεί η οδική ασφάλεια. Αυτό αφορά και τις συνδυασμένε μεταφορές, τις πολυτροπικές και πιο αποτελεσματική εφοδιαστική. Γιατί έχουν σημασία όλα αυτά. Ξέρετε ότι θα αυξηθούν οι προκλήσεις για την κινητικότητα. είναι ε, πιο ε, αποτελεσματική, χρειάζεται ε, να έχουμε μεγαλύτερη χρήση των ήπιων τρόπων μεταφορών για να βεβαιωθούμε ότι και στο μέλλον η κινητικότητα θα είναι και αποτελεσματική και ασφαλής για να μην πω ασφαλέστερη και αποτελεσματικότερη από ό,τι μέχρι σήμερα. Τώρα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε από μια ομάδα εμπειρογνωμόνων να δώσουν μια εκτίμηση ως προς το δυναμικό για τα εφή συστήματα μεταφορών και πώς μπορούν να βελτιώσουν την κατάσταση. Εδώ σας έχω μερικά αριθμητικά στοιχεία. Για το 2020 οι εκτιμήσεις λέγουν ότι τα θανατηφόρα τροχιά μπορούν να μειωθούν κατά 30% και η συμφόρηση κατά 15%. Ε, για το 2020 επίσης αυτά μπορεί να σημαίνουν 13 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό είναι μια τεράστια ε, ευκαιρία για την Ευρώπη. Η Λευκή Βίβλος για τις μεταφορές έχει ήδη μια ισχύ, δηλαδή ζητάει ε, να αναπτυχθούν ευφυή συστήματα μεταφορών. Και βλέπετε εδώ το πιο σημαντικό για μένα εδάφιο, ότι η υποδομή ε, ε, καθορίζει την κινητικότητα και την διαμορφώνει. για να μην γίνει καμία μεγάλη αλλαγή που δεν θα μπορεί να γίνει δυνατή χωρίς τις ε, ευφυείς μεταφορές και ένα αποτελεσματικό δίκαιο. δίκτυο. Συγγνώμη. Τι χρειάζεται τώρα από πλευρά σας. Η διαλειτουργικότητα είναι σημαντική. Χρειάζεται μια διαλειτουργικότητα ασύνδεση και για το χρήστη αλλά και για τις εταιρείε του κλάδου. Χρειάζονται επενδύσεις στις ψηφιακές υποδομές. Τώρα προχωρούμε στην επικοινωνία της τέταρτης γενεάς. 4G και πέμπτη η γενεά στο μέλλον. Εκεί θα πρέπει να ε, κινούμαστε. Ε, και επίση, πρόσβαση σε δεδομένα. Χρειάζεται ένα σωστό πλαίσιο κατάλληλο για ανταλλαγή δεδομένων. Όλα αυτά σεβόμενοι την ιδιωτική ζωή και σφαίρα που είναι πραγματικά αποφασιστική και πρέπει να διασφαλίζεται. Χρειαζόμαστε ένα νέο νομικό πλαίσιο επίσης ε, για να ε, βγουν στους αυτοκινητοδρόμους στο δημόσιο δρόμο αυτόματα αυτοκίνητα. Αν δεν μπορείς ένα πρόγραμμα να το βγάλεις στην αγορά, να το αναπτύξεις, δεν έρχονται ούτε επενδύσεις ούτε εξελίξεις. Χρειαζόμαστε επίσης ασφαλείς ε, επικοινωνίες ασυρμάτου ε, με 5,9 GHz και τις αντίστοιχες προδιαγραφές για τις ε, έξυπνες μεταφορές. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας και τελικά ελπίζουμε η κινητικότητα να γίνει υπηρεσία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ερωτήσεις και απαντήσεις. Ο Βιν Φαντεκάμπ δεν είναι μόνο συντονιστής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος αλλά και εισηγητής του θέματος. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Έχουμε αυτή την ακρόαση και την έχουμε χωρίσει σε τρία τμήματα. Αυτό ήταν το πρώτο τμήμα. Πρόκειται για το οικονομικό πιο πολύ. Πώς θα έχουμε χρήματα για να μπορέσουμε να πληρώσουμε τα δύο επόμενα μέρη που θα ακούσουμε. Που έχουν να κάνουν με την βιωσιμότητα τη κινητικότητας, είναι το δεύτερο και το τρίτο είναι οι πελάτες. Αυτοί που θα μεταφερθούν Υπάρχουν πάρα πολλές ερωτήσεις βέβαια που τίθενται, δεν είμαι μόνο εγώ, υπάρχουν και άλλοι συνάδελφοι που θέλουν να ρωτήσουν, οπότε θα προσπαθήσω να είμαι σύντομο. Κύριε Κάν, ποιες είναι οι τρεις προϋποθέσεις για να υπάρχουν ίσες συνθήκες και να έχουμε θεμητό ανταγωνισμό. Συζητάμε πολύ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για ανταγωνισμό που έχουμε εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κύριε Νίλσον, λέτε ότι δεν είσαστε κατά του EPS, διότι πρόκειται για εξυγχρονισμό των ταξί, αλλά είσαστε κατά, ε, ας μην αναφέρω το όνομα τώρα, ξέρετε ποιανού. Πώς γίνεται αυτό εδώ, υπάρχουν δύο, όλοι βασικά εδώ είμαστε υπέρ των ε, εφαρμογών αυτών για τα ταξί. Πιστεύουμε ότι είναι μια μεγάλη πρόκληση στην Ευρώπη ολόκληρη. Έπειτα κύριε Λόχμαν και κυρία Τεσχέπερ πείτε μας, ποιες είναι οι τρεις προδιαγραφές θα έλεγα που στην μεσοπρόθεσμη αναθεώρηση, όχι την ολοκληρωμένη αναθεώρηση, τη μεσοπρόθεσμη, ποιες είναι οι τρεις προϋποθέσεις που πρέπει να έχουμε για να αλλάξει το είδος μεταφοράς. Ο κύριος Λόχμαν λέει να υπάρχουν δεσμευτικοί στόχοι για τη μείωση εκπομπών εξουδίου του άνθρακα. Ποια κριτήρια πιστεύετε εσείς ότι πρέπει να υπάρχουν για να γίνει πραγματικότητα αυτή η πολυτροπικότητα στις μεταφορές. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Σμέλερ του επόμενος. Α, ζητώ συγγνώμη, όχι. Η Κλάουδια Ταβαρδέλ που είναι και σκιώδης συζητήτρια. Μετά εσύ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θέλω κι εγώ να ευχαριστήσω τους εμπειρογνώμονες που ακούσαμε και που μας παρουσίασαν πώς εκείνοι βλέπουν τις εξελίξεις και την εφαρμογή της Λευκής Βίβλου όσον αφορά τις μεταφορές. Εγώ στηρίζω την ιδέα μιας ενιαίας αγοράς μεταφορών όπου να αναπτυχθούν εξίσου όλα τα είδη μεταφοράς, όλοι οι τρόποι μεταφοράς και να υπάρξουν εξίσου επενδύσεις σε όλες αυτές τις μορφές μεταφορών για να έχουμε μία ενιαία αγορά μεταφορών. Και άρα όλοι οι παίκτες πρέπει να είναι στο ίδιο επίπεδο για όλα τα είδη μεταφορών. Δεν έχουμε πολύ χρόνο βέβαια και υπάρχουν και άλλοι συνάδελφοι που θέλουν να υποβάλουν ερωτήσεις, οπότε μία ερώτηση θα υποβάλω εγώ σε όλους τους ομιλητές μας. Η λευκή αυτή βίβλος πρέπει να είναι ρεαλιστική, πραγματιστική, να εφαρμόζεται εύκολα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θέλω λοιπόν ο καθένας από εσά να μου πει Πέρα από τα προβλήματα τα οποία υπογραμμίσατε, να μου μιλήσετε για ένα στόχο, για μία λύση που θέλετε να συμπεριληφθεί στη λευκή αυτή βίβλο και που θα οδηγήσει σε καλύτερη εφαρμογή του εγγράφου το οποίο συζητάμε σήμερα. Τι θα έπρεπε να συμπεριληφθεί δηλαδή στην νομοθεσία η οποία θα μας βοηθήσει να δημιουργήσουμε αυτόν τον ενιαίο χώρο μεταφορών στην Ευρώπη ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τους διάφορους ε, ομιλητές για τις ε, παρουσιάσεις τους. Εδώ και καιρό ασχολούμαστε με διάφορες πτυχές των μεταφορών, αλλά είναι καλό να ακούμε τον κάθε κλάδο. Βέβαια, ο καθένας από εσά το δικό του κλάδο υπερασπίστηκε και είπε ότι θα πρέπει να μπει ε, στη Λευκή Βιβλό. Έχει φύγει ο Ματιό Κρόσπου, εδώ είναι. Α, εδώ είσαι, νόμιζα ότι είχες φύγει το ακούμε στη συζήτηση, έχουμε τη Λευκή Βίβλο το 2011, χρειάζεται ενημέρωση, επικυροποίηση που υπάρχουν ελλείμματα και πώς θα προχωρήσουμε. Να ρωτήσουμε και τον Ματιό Γκρός, γιατί μου έκανε εντύπωση στην ομιλία του όταν αναφέρθηκε στις θαλάσσιες μεταφορές, έβαλε ένα αρνητικό πρόσημο για τη κατά πόσο σέβονται το περιβάλλον. Αυτό αφορά τα πολύ μεγάλα δεξαμενόπλια ή κάποια πολύ μεγάλα καράβια που χρησιμοποιούν καύσιμα που ρηπαίνουν το περιβάλλον. Γιατί έχει βάλει αρνητικό πρόσημο. Εγώ θεωρούσα ότι είναι φιλικές οι θαλάσσιες μεταφορές. Για τον κύριο Νίλσεν ήμουνα σε μια τέτοια ομάδα υψηλού επίπεδου ε, ζητάτε να διπλασιαστεί η κυκλοφορία στους δρόμους. Ε, και εγώ συμφωνώ γενικά γιατί αλλιώς δεν γίνεται. Είμαι και υπέρ των πιο μεγάλων φορτηγών σε διαστάσεις, αλλά δεν είναι το θέμα μας αυτό. Το συζητήσαμε στην ομάδα υψηλού επίπεδου, αλλά από εμά τι ζητάτε, τι μπορούμε να κάνουμε για σας. Για τον κύριο Χάν, είμαι πάρα πολύ δίκαιη, βλέπετε, έχω μια ερώτηση για τον καθένα. Είπατε κανονικά ότι είμαστε καλύτεροι από τους αερομεταφορείς άλλων ε, περιοχών του κόσμου. Για ποιο λόγο. Και ε, εδώ όμως υπάρχει και μεγάλος ανταγωνισμός σε σχέση ας πούμε με αερομεταφορείς από τις χώρες του Περσικού κόλπου. Ε, και η Επίτροπος διαπραγματεύεται αυτό το καιρό με τις χώρες αυτές. Ε, τι περιμένετε από μας να κάνουμε για να βελτιωθεί η θέση μας προς τον κύριο Λόχμαν. Έχω μια συνήθιστη ερώτηση, θα δείτε, γιατί μιλήσατε για εξηλεκτρισμό, ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για το σιδηρόδρομο. Συμφωνώ απολύτως αλλά και κάτι που θα μπορούσα να ρωτήσει και από πριν, ε, τώρα το σκέφτηκα. Στον εξηλεκτρισμό είναι λιγότερες εκπομπές και το επιθυμούμε όλοι βεβαίως, αλλά ο σιδηρόδρομος πανευρωπαϊκά εξασφαλίζει, δηλαδή είναι και αηφόρος και βιώσιμη η, παροχή, η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, γιατί δεν είναι πάντα αηφόρος και βιώσιμη και σεβόμενη το περιβάλλον η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτό θα με ενδιέφερε. Πού θα το βρείτε το ρεύμα και πώς θα παράγεται. Ε, για την κυρία Τεσχέπερ. Αναφέρατε κάτι με το οποίο συμφωνώ κι εγώ. Ε, για να υπάρχουν εσωτερικές πλωτές μεταφορές, να μην είναι πάνω από 300 χιλιόμετρα η απόσταση. Συμφωνώ, αλλά θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο. Υπάρχει ένα πακέτο για την καθαρή ενέργεια στις μεταφορές. Clean Power of Transport. Δεν ήταν και τόσο λαμπρά τα αποτελέσματα. Στις εσωτερικές πλωτές ε, οδούς και αλλού ε, δεν ε, προχωράει πολύ το θέμα της εγκατάστασης θυμάτων αερίου για την κίνησή τους. Και έχω και μια ερώτηση. Μ' αρέσουν όλα αυτά για τις έξυπνες μεταφορές. Ο γαμπρός μου και αυτός είναι εφευρέτης και βρίσκει διάφορα οχήματα χωρίς οδηγό, με αυτόματη οδήγηση κτλ. Αλλά ενδιαφέρομαι πάρα πολύ ε, για ε, την προστασία των δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής. Με όλα αυτά τα σούπερ δίκτυα και τα καινούργια, ε, πώς εξασφαλίζετε την προστασία των δεδομένων. Η Μαρία Κίλων. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ όλους τους ομιλητές. Έχω μια ερώτηση στην οποία μπορεί να απαντήσει οποιοδήποτε εφόσον έχουμε χρόνο. Πώς μπορούμε να δεδοθούμε ότι τα συστήματα μεταφορών μας, όλα τα μέσα και όλοι οι τρόποι μεταφοράς θα διασυνδεθούν σωστά ώστε οι χρήστες να έχουν τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες. Για την ώρα επικεντρωνόμαστε στο κάθε τρόπο και στο κάθε μέσο μεταφοράς ξεχωριστά. Φαίνεται να υπάρχει ανταγωνισμός μεταξύ των διαφόρων δικτύων για να προσελκύσουν ξεχωριστά όλο ο δυνατόν περισσότερους επιβάτες. Σκέφτομαι προς τον κύριο Μάγερ λοιπόν, διότι από τη σκοπιά της οδικής ασφάλειας μπορούμε να φανταστούμε να δημιουργείται ένα σύστημα παρόμοιο με τα τραπεζικά. Εσείς έχετε βάσεις δεδομένων που έχετε όλες αυτές τις πληροφορίες. Μπορούμε να σκεφτούμε κάτι τέτοιο. Κυρία Κλούν, ευχαριστώ όλους τους ομιλητές για τον κύριο Καν των Ευρωπαϊκών Αερομεταφορών. Βεβαίως μας απασχολεί ο αντίκτυπος ε, της λειτουργίας των αερογραμμών εκτός Ευρώπης και είπατε ότι το σύστημα είναι παγκόσμιο πλέον. Εντός αυτού λειτουργούν και οι ευρωπαϊκές αερογραμμές και θα πρέπει αυτό να το λαμβάνουν υπόψη. Το ίδιο και για την τιμή που επιβάλλουν. Βεβαίω για του επιβάτε τα νέα δεν είναι πάρα πολύ καλά γιατί η κατάσταση δεν φαίνεται να είναι βιώσιμη όσο έχει σήμερα. Πώ θα αντιμετωπίσετε λοιπόν τι προκλήσει για να υπάρχουν ίσοι κανόνε ανταγωνισμού, διότι όλοι συζητάμε την ε, διέλευση εκατομμυρίων επιβατών από τα αεροδρόμια μας, όμως η κυκλοφορία επιβατών στις ΗΠΑ είναι συγκρίσιμη. Πώς θα τους πάρουμε πίσω. Και μας ενδιαφέρει πώς αυτό θα μπορούσαμε να το αντιμετωπίσουμε. Ακόμη και για τις μικρές περιφερειακές αερογραμμές. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ ο Δίτερ Κόχ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θέλω να ρωτήσω κάτι τον εκπρόσωπο της Έρτικο. Κύριε Μάιε, για το πολυτροπικό εισιτήριο και τη τιμολόγηση, ε, πραγματικά είναι κάτι που σας γοητεύει πάρα πολύ. Εγώ συζητώ με εταιρείε που κανονικά θα πρέπει να συμμετείχαν σε ένα τέτοιο σύστημα. Αυτοί φοβούνται τι υπερβολικέ ρυθμίσει περισσότερο, τρομάζουν. Και σου λέει, κάτω τα χέρια η πολιτική από αυτό, θα τα ρυθμίσει η αγορά. Εσεί πώ το βλέπετε, χρειάζεται πολιτική ρύθμιση, κίνητρα, νομοθεσία ή θα τα ρυθμίσει η αγορά από μόνη τη. Ευχαριστώ. Αυτέ ήταν οι ερωτήσει. Δύο λεπτά για τι απαντήσει. Αρχίζουμε. Ήθελα να σα αφήσω για τελευταίο, Ματιό, να σου δώσω το λόγο στο τέλος, με την αντίστροφη σειρά δηλαδή, να απαντήσεις. Ευχαριστώ πολύ για τις ερωτήσεις σας, λέει ο κύριος Νίλσεν. Ναι, για τις εφαρμογές ευχαριστώ, να τις αναφέρω. Για ποιον λέτε, για την Ούρβα, για ποιον λέτε, που δίνει τόσα λεφτά για να γίνει γνωστή. Ευχαριστώ. Μία μόνη υπηρεσία έχουν από τις διάφορες. Οι άλλες είναι παράνομες. Το πλάκα είναι μια άλλη περίπτωση. Εμείς θέλουμε οι κανόνες να τηρούνται. Αυτό είναι το πρώτο που θέλουμε. Και έπειτα, όπως είπα, θέλουμε πρόσβαση σε κανόνες επαγγελματικούς που να ισχύουν και για αυτές τις εφαρμογές και για αυτές τις εταιρείες που λένε ότι είναι καινοτόμες εταιρείες Υπήρχε μια ερώτηση που κάνατε για την ενιαία αγορά μεταφορών και τι θέλουμε να συμπεριληφθεί. Πιστεύουμε ότι αυτό που πρέπει να γίνει είναι να υπάρξει καινοτομία σε όλους τους τρόπους μεταφοράς. Να μην υπάρχει προστατευτισμός και κάποια είδη μεταφορών εμποδίζουν την καινοτομία σε άλλα είδη μεταφορών. Αυτό είναι πολύ σημαντικό πιστεύω. Ευχαριστώ όλους και την κυρία Μάισνερ αλλά και τους άλλους συναδέλφους. Ναι, είμαστε υπέρ των μεγαλύτερων φορτηγών, ναι, βεβαίως. Εδώ είχαμε εννέα που συμμετείχαν. 25 δευτερόλεπτα έχω ακόμα. Αυτοί οι εννέα λοιπόν είναι από ρυθμιστές, καινοτόμοι κλπ. Δύο θα αναφέρω. Η μία περίπτωση έχει να κάνει με τις υποδομές. Πρέπει να υπάρχουν υποδομές. Στη Σουηδία υπάρχει ένα πάρα πολύ καλό σχέδιο για το πώς να γίνει τα λεωφορεία, τα πούλμαν λοιπά έχουν πρόσβαση σε σταθμούς, αεροδρόμια κλπ. πολύ εύκολα. Δικτύωση. Και εδώ είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει δικτύωση και στα αεροδρόμια, στους σταθμούς κτλ. αλλά και μεταξύ των διαφόρων ειδών μεταφοράς να υπάρχει σύνδεση. Αν είχαμε ένα καλό πολυτροπικό σύστημα θα έπρεπε όντω να υπάρχει σύνδεση με τα δεδομένα είτε πρόκειται για τα λιμάνια στα, στην εδωχώρα, στις εσωτερικές πλωτές δηλαδή μεταφορές, θα έπρεπε να υπάρχει σύνδεση και με τα αεροδρόμια και με τους σταθμούς, τα τρένα κτλ. Αυτή η διασύνδεση, τα δίκτυα είναι κάτι πολύ σημαντικό. Ευχαριστώ πολύ ο κύριος Χάν. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ενδιαφέρον που οι περισσότερες ερωτήσεις από διάφορους βουλευτές ασχολούνται όλοι με το ίδιο θέμα. Ας προσπαθήσω να τις ομαδοποιήσω. Τι θα πρέπει να κάνουμε. Σε αυτά που είπε ο κύριος Βαντεκάμπτ. Πρώτο, να είμαστε πολύ σαφείς και πολύ ρεαλιστές. Θα πρέπει να βάλουμε τον οίκο μας σε τάξη στην Ευρώπη και δεν διακρινόμαστε σε αυτό. Έχουμε νομοθεσία για τη βελτιστοποίηση, ό,τι θέλετε, ε, αξιοποίηση, καλύτερη βελτιστοποίηση στην ε, ευρωπαϊκή αγορά. Δεν το εφαρμόζουμε δεν είμαστε πάρα πολύ καλοί στο κόστος ωφέλεια, δεν αποδίδουν τα μέσα μεταφοράς. 5 δισεκατομμύρια άχρηστα ε, κοστίζει ε, το σύστημα των ε, εθέρων και 11 εκατομμύρια, ε, ε, με μάλιστα διάφοροι τόνοι εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα το χρόνο και ε, άσκοπη ταλαιπωρία και καθυστέρηση για τους επιβάτες. Χρειάζεται μεγαλύτερη αποκλειστικότητα, αποτελεσματικότητα. Σε ό,τι αφορά τις αεροπορικές εταιρείες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς θεωρούμε ότι η εσωτερική αγορά ήταν πάρα πολύ επιτυχής με Οφέλη και προσφορές για ε, τους επιβάτες θα έπρεπε να το έχουμε κάνει πριν από 15 χρόνια. Είναι καλοδεχούμενο οποιαδήποτε εξωτερική εταιρεία υπό τον όρο ότι θα παίζουν με τους ίδιους κανόνες, γιατί έτσι δημιουργήθηκε η ενιαία αγορά στην Ευρώπη των αερομεταφορών. Και ποιο θα ήταν το κλειδί, κύριε Βανταγκάμπ, ε, η σύγκληση στις ρυθμίσεις και μάλλον η διαφάνεια. Είναι τα βασικά ζητήματα που μας ενδιαφέρουν και εκτιμούμε πάρα πολύ στην Ευρώπη και που θα ζητούσα εγώ από τους άλλους. Για την κυρία Κλούν, για τις περιφερειακές αγορές, ε, οι περιφερειακές εταιρείε ή την ειδικιά σας ή άλλες χώρες περιφέρειας είναι απαραίτητες για τη διασύνδεση στην Ευρώπη και την προστιθέμενη αξία. Η Διατλαντική Συμφωνία τι λέει, η Ευρωπαϊκή Ένωση και ε, οι Ηνωμένε Πολιτείε θα πρέπει να έχουν κάπως το ίδιο πλαίσιο ιδεών για τον ανταγωνισμό, για ε, την ε, λειτουργία της αγοράς και να το χρησιμοποιούν ως ένα προσχέδιο που θα μπορούσε να εξαχθεί και σε άλλες χώρες. Ο Λίμπορ Λόχμαν και πάλι τώρα. I was asked Για τρία πράγματα με ρωτήσατε για τις υποδομές οι ηλεκτρικές υποδομές, υποδε... υποδομές που να στηρίζουν τις πολυτροπικές μεταφορές. Αυτό είναι το ένα. Δεύτερον, οι ίδιες συνθήκες ανταγωνισμού. Αρχή, ο χρήστης πληρώνει, ο ρηπαίνων πληρώνει. Και εσωτερήκευση του εξωτερικού κόστους. Πιστεύω ότι έτσι καλύπτω. Τρίτον, έρευνα και καινοτομία για να βοηθηθούν όλοι οι τομείς. Περιμένουμε όμως χρόνια για το πρόγραμμα Shift Rail και ακόμα περιμένουμε. Αυτό είναι το τρίτο λοιπόν. Όσον αφορά τώρα τον ηλεκτρισμό για του σιδηροδρόμου εξαρτάται φυσικά από το ενεργειακό μείγμα, το γνωρίζουμε. Ξέρουμε όμως επίσης ότι υπάρχει και μετακίνηση για το φιλτράρισμα του διοξιδίου του άνθρακα μεταφορά προς καθαρές ενέργειες, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αν το λάβουμε αυτό υπόψη μας και την ηλεκτρική ενέργεια, όντως η ηλεκτρική ενέργεια θα μπορούσε να είναι η λύση για το μέλλον. Ηλεκτρισμός λοιπόν για τους υδροδρόμους και για όλους τους τρόπους μεταφοράς. Και αυτό το λαμβάνουμε υπόψη μας όταν προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε τις εκπομπές και ξέρετε ότι και στην ε, Ελβετία και στη Σουηδία έχουμε 1% χωρίς ρήπανση. Το cross ticketing, ναι, βάσει εμπορικών συμφωνιών, ώστε να επωφεληθεί ο πελάτης, αλλά για να γίνουν και πιο ελκυστικές οι υπηρεσίες που προσφέρουν επιχειρηματίες. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Thank you, Chairman. Ευχαριστώ. Τρία πράγματα ε, ε, του Βιν Καμπ και εγώ. Ήδη στην Ευρώπη η χημική βιομηχανία και άλλοι κλάδοι ακριβώς λόγω της λειτουργίας τους εξαρτώνται από τις εσωτερικές πλωτές οδούς. Το χρειάζονται. Είναι ένα πλεονέκτημα ανταγωνιστικό που διαπερνά όλη την αλυσίδα και ε, ε, τους ενδιαφέρει ο κλάδος μας. Και με φρίκη διαπιστώνουν ότι τα κράτη δεν συντηρούν και δεν αναβαθμίζουν τις εσωτερικές πλωτές οδούς και τα συστήματα. Ε, θα πρέπει αλλιώς να βρουν μια εναλλακτική λύση, να αλλάξουν τρόπο μεταφοράς και θα το ζήσουμε στις τιμές και θα το αισθανθούμε εμείς. Μετά, όταν έχουμε τη δυνατότητα για πλήρως συνδυασμένες μεταφορές, θα πρέπει να έχουμε πραγματικό συνδυασμό, πραγματικά ε, πολυτροπικές μεταφορές στους τερματικούς σταθμούς, στους λιμένες, θα πρέπει να υπάρχουν όλες οι δυνατότητες και όταν υπάρχουν προβλήματα να μπορούν να επιλέγουν οι φορείς της αγοράς έναν άλλο τρόπο μεταφοράς και επίσης να εξασφαλίσουμε την ανταλλαγή δεδομένων για να υπάρξει αυτή η σύνδεση, ο συνδυασμός, το bundling. Είναι και άλλα, αλλά ε, θα μπορούσα να φερθώ σε περισσότερα, συνοψίζω. Για την καθαρή ενέργεια για τις μεταφορές, την κυρία Μάισνερ, θέλω να πω ότι ο κλάδος με τη βοήθεια και των ιδιωτών και του δημοσίου πάρα πολύ γρήγορα έχει περάσει στην ανάπτυξη με το σχέδιο το ρυθμιστικό για το υγροποιημένο φυσικό αέριο. Και έχει σημασία να συνεχιστεί η υποστήριξη, διότι υπάρχει ε, Ρήνος, Μάιν, Δούναβης, αυτός ο άξονας ε, για ε, νέα ε, μορφή ε, παροχής αυτού του καυσίμου να εξοπλιστούν τα πρώτα σκάφη, τα πρώτα ποταμόπλια με αυτή την ενέργεια ε, και είναι πολύ σημαντικό γιατί κάποιοι εργάζονται και για υδρογονοκίνητα σκάφη όταν γίνεται λόγος για τέτοιες μεταφορές όλοι χειροκροτούν, αλλά μετά το θέμα είναι τι γίνεται στην εφαρμογή, την ουσιαστική. Ο κύριος Μάιερ θα αρχίσω από το αυτονόητο, η προστασία των δεδομένων. Σίγουρα είναι πολύ σημαντικό αυτό το θέμα στα ευφύ συστήματα μεταφορών και την ανταλλαγή δεδομένων. Πολλή δουλειά γίνεται έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε ε, ότι θα λαμβάνονται αυτά υπόψη, βέβαια με ανώνυμο τρόπο χρήσης των δεδομένων, με μειωμένη αποθήκευση χρονικά με ενημέρωση του χρήστη, τι γίνονται τα δεδομένα και υπάρχει μια δυνατότητα ε, για κάποιο χρήστη να καταλήψει αυτή τη δυνατότητα, να τη σβήσει, να πει δεν με ενδιαφέρει αυτή η παροχή υπηρεσιών γιατί ανησυχώ. Υπάρχουν όμως περιπτώσεις που έχει πολύ μεγάλη σημασία η ανταλλαγή δεδομένων και σώζει και ζωές. Και εκεί χρειάζεται συζήτηση, εάν σε αυτό το πλαίσιο επιτρέπεται ή αν επιτρέπεται κάποιος να σβήσει ε, το σύστημα και να βγει στις μεταφορές. Ένας οδηγός ας πούμε. Και αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη. Αλλά χρειαζόμαστε περισσότερες συζητήσεις και τη δική σας υποστήριξη πάντα σε αυτή τη συζήτηση. Τώρα, για το ενιαίο εισιτήριο, για διάφορους τρόπους μεταφοράς. Εγώ δεν ζητάω εύκολα νομοθεσία. Και σε αυτό το θέμα πάλι νομίζω δεν βρισκόμαστε σε ένα στάδιο ή σε μια φάση που να ζητούμε νομοθεσία. Υπάρχουν μεγάλες δυνατότητες σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Τούτων όμως λεχθέντων θα πρέπει να πούμε ότι και εδώ χρειαζόμαστε ευρωπαϊκές λύσεις. Για ποιο λόγο ευρωπαϊκές λύσεις. Διότι αυτό είναι προς όφελος και των χρηστών αλλά και επειδή είναι υπέρ και ωφελούν τη βιομηχανία γιατί δημιουργείται μεγάλη κλίμακα και ε, συμφέρει η παροχή αυτών των υπηρεσιών. Θα πρέπει να κινηθούμε προς τα εκεί, ευρωπαϊκές λύσεις, αλλά το πρώτο βήμα πάντα είναι η εθελοντική συμμετοχή. Για να βρούμε το σωστό τρόπο ώστε να παρέχονται υπηρεσίες, να ανταλλάσσονται πληροφορίες και δεδομένα και να διευκολύνονται. Σε ό,τι αφορά την πρόταση για το τραπεζικό λογαριασμό, Ενδιαφέρον είναι αυτό, δεν ξέρω, πρέπει να δούμε και με την ασφάλεια δεδομένων τι γίνεται, ας το σκεφτούμε. Και ό,τι αφορά τη χρήση ευφυών συστημάτων μεταφορών για να ολοκληρωθούν διάφορα μέσα και τρόποι μεταφοράς, μα ακριβώς περί αυτού πρόκειται. Αυτό θέλουμε, να έχουμε ολοκληρωμένες μεταφορές στα διάφορα μέσα υπέρ ε, των ε, επιβατών, των ταξιδιωτών και των εμπορευματικών μεταφορών. Και εκεί πρέπει να κινηθούν οι σχεδιασμοί για τις μετρονητικές πολιτικές. Ευχαριστώ. Τελευταίος, χωρίς να είναι λιγότερο σημαντικός, ο Ματιό Εγκρός. Ευχαριστώ για το ενδιαφέρον και για τις ερωτήσεις. Γκεζίνε, εσύ απάντησες μόνη σου την ερώτηση. Είναι μόνο 3% των εσωτερικών πλωτών μεταφορών. Εγώ ξεκίνησα από τους μεγάλους, αλλά χρειάζονται και στις αλλάσεις μεταφορές προσπάθειες. Αν δούμε τι γίνεται αλλού, ε, ανάμεσα στο ε, ευρώ 1 και το ευρώ 6 για τους κινητήρες των αυτοκινήτων, ας πούμε, ε, υπάρχει περιθώριο. Και πάντα ο πρόεδρος μας ανέφερε ένα παράδειγμα κάποιων εγκαταστάσεων καύσης που ήταν εξωφρενικά πράγματα. Τώρα για την νομοθεσία. Κάτι που ε, ρυθμίζει μόνη της η αγορά, δεν χρειάζεται νομοθεσία. Αλλά εάν η αγορά δεν μπορεί να ρυθμίσει τα κοινωνικά, τα περιβαλλοντικά ή κάποια θέματα ασφαλείας ή ακόμα και του χώρου που λέγεται Ευρώπη, ας πούμε αν δεν κάνουμε προσπάθειες, αύριο θα έρθουν προδιαγραφές και πρότυπα από την Κίνα και από αλλού που θα μας ξεπεράσουν γιατί εμείς δεν θα έχουμε βάλει τη βάση, τα θεμέλια. Γι' αυτό η νομοθεσία στις μεταφορές είναι για μένα απαραίτητη και αναγκαία, συνοδευτικά για κάτι που ήδη κάνει αγορά. Πάντως έχουμε διαπιστώσει το εξής. Στα ΙΧ για τις εκπομπές ε, διοξιδίου του άνθρακα και αερίων Είχαμε αφήσει την αγορά να το ρυθμίζει και ε, δεν έκανε τίποτα. Και όταν κάναμε νομοθεσία, μετά από δύο χρόνια είχαν έρθει όλα αυτά που ζητούσαμε δέκα χρόνια και δεν γινόντουσαν. Και κάτι άλλο που είπα και προηγουμένως, για μένα είναι πάντα κακό και αρνητικό να αποφασίζουμε κάτι εδώ και να μην το επιλούν τα κράτη-μέλη. Εκεί είμαστε, πρέπει να είμαστε πιο αποτελεσματικοί για να εξηγήσουμε στους πολίτες. Έχουμε λάβει σε τρία ε, φόρα αποφάσεις τα λειτουργικά διαστήματα ε, στον αέρα θα πρέπει να λειτουργούν για τον έλεγχο της ενέργειας κυκλοφορίας. Έξι είναι τον αριθμό. Σήμερα έχουμε ακόμα 27 διαφορετικές δομές που είναι και πιο ακριβές και πιο εχθρικές για το περιβάλλον και πιο επιβαρυντικές και από πλευράς αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας είναι χειρότερα ουδής κατανοεί για ποιο λόγο δεν προχωράει αυτή η υπόθεση. Και ένα τελευταίο ερώτημα για τις συνδυασμένες μεταφορές. Είναι πολλά τα υπέρ. Για μένα το σημαντικό είναι ο σωστός και θεμητός ανταγωνισμός μεταξύ των διαφόρων μέσων μεταφοράς. Η εσωτερήκευση του κόστους ξέρω ότι είναι δύσκολο, αλλά θα πρέπει αύριο να το τολμήσουμε το κόστος που δημιουργεί ή προκαλεί ένα μέσο μεταφοράς ή οι επιβάτες θα πρέπει να το επομίζονται και αυτοί. Για να λειτουργήσουν αύριο συνδυασμένες μεταφορές χρειάζονται πολύ ε, πιο ενιαίες ε, προδιαγραφέ και πρότυπα για του χώρους αποθήκευση, γιατί διαφέρουν τόσο πολύ ανάλογα ε, με το μέσο μεταφοράς που έχουμε ε, πραγματικά πρόβλημα. Θυμάστε την έκθεση Στόκμαν πριν από 8 χρόνια ακόμα είναι στα σερτάρια του Συμβουλίου, για να μην πω στο ψυγείο του Συμβουλίου. Έχει παγώσει. Ε, αν έχει κανείς και θέλει να έχει σωστή εφοδιαστική, υπάρχουν σήμερα οι δυνατότητες και μπορούμε να βρούμε ε, ένα τρόπο, χωρίς να απεμπολίσουμε τον έλεγχο, να διευκολύνουμε πάρα πολύ τις διοικητικές δομές. Εκεί παίζει ρόλο η καλύτερη συνεργασία διαφόρων ε, τρόπων μεταφοράς και μεταφόρτωσης και εκεί μπορούν να βοηθήσουν κάποιοι νόμοι. Ευχαριστώ πολύ ο Πρόεδρος, τον Ματιό Εγκρός και όλους ε, τους ε, ομιλητές του πρώτου πάνελ. Ενδιαφέρουσες και η παρουσιάση και η συζήτηση. Παρακαλώ καθίστε για να έρθουν οι ομιλητές για το δεύτερο πάνελ. Because we are short in time. Επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο, ας αρχίσουμε με το δεύτερο πάνελ. Okay, das zweite Panel, das beschäftigt sich. Δεύτερο πάνελ το δεύτερο πάνελ έλεγα ασχολείται με την αηφόρο και βιώσιμη κινητικότητα. Ο πρώτος ομιλητής μας είναι ο Γιος Ντίνξ, ε, Διευθυντής της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Μεταφορών και Περιβάλλοντος. Έχετε το λόγο για έξι λεπτά, παρακαλώ. Uh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Για τη διοργάνωση αυτής της επίκαιρης εκδήλωσης και για την ευκαιρία να εκφράσω τις απόψεις μου. Είμαι ε, ο πρόσωπος του Ευρωπαϊκού, της Ευρωπαϊκής Νομοσπονδίας για τις μεταφορές και το περιβάλλον και εκπροσωπούμε ένα σωρό ενώσει σαν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για τις μεταφορές ξέρω ότι η πρόοδος ακόμη δεν είναι αρκετή, αλλά κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βρούμε λύσεις. Η Ευρώπη οι μεταφορέ είναι υπεύθυνε για το 1 τρίτο των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα και ουσιαστικά οι μεταφορές ε, το ίδιο και για την καύση άνθρακα και τη χρήση πετρελαίου μάλλον. Εδώ πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να καλύψουμε το κόστος των περιβαλλοντικών ε, πολιτικών και των πολιτικών μας ασφάλειας διότι πρέπει να αποδώσουμε κέρδος στην καινοτομία και στην αποτελεσματικότητα για να μειώσουμε και τις εισαγωγές πετρελαίου που είναι τουλάχιστον αντιπαραγωγικός τρόπος για να δαπανούμε τα χρήματά μας. Ελπίζω να συμφωνούμε όλοι σε αυτό. Έχουμε όμως και καλές ειδήσει. Έχουν εγκριθεί νόμοι για τα οχήματα και τα κάψιμα που φαίνεται να, να έχουν κάποια θετικά αποτελέσματα όπως ο αέρας μας που γίνεται λίγο καθαρότερος και η χρήση ενέργειας λίγο αποτελεσματικότερη. Βλέπουμε τα ηλεκτρονικά αυτοκίνητα που αρχίζουν να χρησιμοποιούνται στην Δυτική Ευρώπη. Αυτό είναι καλή ε, είδηση, διότι σημαίνει ότι θα χρειαστεί να κατασκευάσουμε λιγότερου δρόμους. Η οροφή ε, για τα ηλεκτρονικά ποδήλατα όλο ένα και αυξάνεται. Έχει φτάσει στα 2 εκατομμύρια ε, στην Ευρώπη, που έχει και κατανομή των τιμών. Ε, η κατανομή μάλλον των διαδρομών στα αυτοκίνητα. Πολλοί μοιράζονται τα αυτοκίνητα κάτι που έχει, ήταν σε μηδενικά επίπεδα πριν από 10 χρόνια. Λόγω αυτών των εξελίξεων βλέπουμε για πρώτη φορά ότι η χρήση του πατρελαίου και τη βενζίνη, οι εκπομπέ του δεξιού του άνθρακα μειώνονται κάπω για πρώτη φορά. Αλλά δεν μειώνονται αρκετά δραστικά. Μόνο 1% το χρόνο συνολικά. Ε, αυτό δεν οφείλεται βέβαια Αυστρία και μόνο στην κρίση. Ε, τι σημαίνουν όλα αυτά για τη Λευκή Βίβλο και την αναθεώρησή της. Να ε, κάνω πέντε παρατηρήσεις. Πρώτον, νομίζω σημαντικό είναι να θέσουμε στόχους για τις εκπομπές αερίου αερίων του θερμοκηπίου μέχρι το 2030 και οι πολιτικοί μας ευθύνοντες έχουν ήδη θέσει ένα πλαίσιο για τους τομείς για τους τομείς του συστήματος ανταλλαγής ε, δικαιωμάτων και όχι. 60% ε, μέχρι το 2050. Αυτές είναι σωστές κατευθυντήριες γραμμές και είναι ένας καλός τρόπος για να ε, έχουμε ένα πλαίσιο για το τι να επιδιώκουμε στις μεταφορές. Η στόχη είναι ένα πράγμα, το να του επιτύχουμε είναι κάτι άλλο βέβαια. Πώς θα το επιδιώξουμε. Η ε, ανακοίνωση για την Ενεργειακή Ένωση σωστά θέτει πρώτο στόχο την αποδοτικότητα. Εκεί έχουμε κάποια εμπειρία με του στόχου αποδοτικότητα για ορισμένα οχήματα. Θα πρέπει να το επεκτείνουμε παντού, στα φορτηγά, τα πλοία, τα αεροσκάφη. Θα πρέπει να προβλέψουμε τα επόμενα βήματα για τα φορτηγάκια και τα ε, αυτοκίνητα. Πολύ σύντομα, διότι χρειάζεται πολλή χρόνο μέχρι όλα αυτά τα οχήματα να ε, εξοπλιστούν σωστά και να περάσουν στον στόλο που χρησιμοποιείται. Είναι σπαζοκεφαλιά. Επίση, ε, η νέα ανακοίνωση μιλά για την ηλεκτροκίνηση ως νέα ε, λύση, κάτι που μας βρίσκει σύμφωνους. Ε, είμαι ακόμη πολύ ακριβή η βενζίνη και είναι και βρώμικη και εισάγεται. Ε, για τα βιοκαύσιμα δεν έχω δει ακόμη ένα μεγάλο φιλόδοξο πρόγραμμα για την ευρεία διάδοσή τους. Έτσι λοιπόν, ε, με όλα τα άλλα να, τα, ε, να μην μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε παρκώς, ο ηλεκτρισμός γίνεται το καλύτερη λύση. Η... Έχει μειωθεί και κατά 10 η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από την αιωλική τα τελευταία 10 χρόνια. Είμαστε κοντά στα, σε μια πραγματική επανάσταση τα τελευταία χρόνια και το 70% των νέων δυνατοτήτων για την παραγωγή ενέργειας, ε, ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη γίνεται πλέον από ανανεώσιμες πηγές. Αυτό είναι πολύ καλή είδηση, άρα ο τομέας αυτός βρίσκεται σε πολύ καλή πορεία, πολύ καλύτερη από την μηχανία λόγου χάρη. Όμως η ηλεκτρική ε, Διαφέρει πολύ από το να αλλάξουμε τους κινητήρες σε ένα όχημα και να κάνουμε ηλεκτρικούς. Ε, δεν είναι αυτό το μόνο πρόβλημα. Είναι πολύ ευρύ ε, το θέμα. Αφορά και τους υδροδρόμους, τα ποδήλατα, τα μικρότερα οχήματα και την μετακίνηση εμπορευμάτων. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε πολύ ελκυστικότερο τομέα ενέργεια ώστε το μέλλον τα ηλεκτροκίνητα οχήματα να καλύπτουν την πρόσβαση στην ανανεώσιμη ηλεκτρική ενέργεια εφόσον υπάρχει αρκετή ζήτηση και ε, προσφορά, και να φροντίσουμε τα σημεία φόρτιση των ηλεκτροκινητών οχημάτων, αλλά και το θέμα των εισιτηρίων, κάτι που συζητήθηκε προηγουμένω για τι δημόσιε μεταφορέ. Θα πρέπει να μεγιστοποιήσουμε την ε, κατανεμημένη χρήση, δηλαδή τα ηλεκτροκίνητα οχήματα να χρησιμοποιούνται συλλογικά, είναι πολύ ακριβά να να αγοράσει κανεί, αλλά πολύ φτηνά στη χρήση. Είναι πολύ καλό λοιπόν το επιχειρηματικό μοντέλο τη πολλαπλή χρήση ε, για να ξεφύγει κανεί από την ιδιωτική χρήση, τα γεωταχή, ένα άλλο μεγάλο θέμα που απασχολεί πλέον την κοινωνία μα και πρέπει να επικεντρωθούμε στι αστικέ περιοχέ, τι μεγάλε αποστάσει και όχι μόνο τα μεγάλα αστικά κέντρα, αλλά και τι διεθνεί μα προτεραιότητε. Μιλάμε για μια μεγάλη μετάβαση με μεγάλε ευκαιρίε και πιστεύουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να καταστρώσει μια ευρεία στρατηγική για να καλύψετε τι ανάγκε. Αυτή την έκκληση σα απευθύνουμε και ελπίζουμε να μην αφήσουμε τι ΗΠΑ να μα περάσουν. Εάν όλα αυτά θέλουμε να γίνουν πραγματικότητα, πρέπει να εργαστούμε ώστε οι τιμέ να είναι σωστέ για τι μεταφορέ. Οι τιμέ αυτή τη στιγμή δεν είναι οι καταλληλότερε. Ε, φορολογούμε πάρα πολύ την εργατική δύναμη και μετά μας εκπλήσει γιατί υπάρχει τόση ενεργεία. Οι βρώμικες μεταφορές από την άλλη είναι πολύ ε, χαμηλής φορολόγησης. Γι' αυτό μας απασχολεί μετά περιέργως πώς έχουμε τόση ρήπανση. Πρέπει λοιπόν να βιαστούμε και να επιβάλλουμε τέλη και στην ε, μετακίνηση εμπορευμάτων και ε, στην κυκλοφορία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να διευκολύνει στην επιβολή ε, τελών. Για την ε, η να πω δύο λόγια, η η ΚΑΟ ε, εργάζεται για τα διεθνή πρότυπα και σας είπα προηγουμένως για το σύστημα εμπορία δικαιωμάτων αέριων θερμοκηπίου. Ο λόγος που έχουμε διεθνείς προτεραιότητες είναι επειδή και σε περιφερειακό επίπεδο πρέπει να συνεχίσουμε τις προσπάθειες. Θα μπορούσαμε βέβαια να συζητήσουμε το τι γίνεται με τον ε, έξωθεν ανταγωνισμό. Ε, με το υπόλοιπο ίσως πάνελ, δεν θα προλάβω να το θίξω. Και μετά για την για, τα, για τις θαλάσσιες μεταφορές, εδώ δεν έχουμε στόχους σε σχέση με το κλίμα, θα πρέπει λοιπόν να θέσουμε και εδώ κάποιες προτεραιότητες στόχους και πρότυπα για να, μειωθεί, για να μειωθούν και σε αυτό το τομέα εκπομπές. Μόλις άρχισαμε να τις παρακολουθούμε, έχετε μια έκθεση της πρωτοβουλίας για το θέμα, είναι η στιγμή να μειωθούν και αυτές οι εκπομπές. Χρειαζόμαστε στόχοι λοιπόν, στόχους, προδιαγραφές αποδυτικότητας, ηλεκτροκίνηση, σωστή τιμαρρύθμιση και τιμολόγηση μάλλον και για την αεροπλοεία και σωστή φορολόγηση των εκπομπών ε, των ε, θαλάσσιων μεταφορών. Με 7,5 λεπτά συγχωρείτε. Ευχαριστώ, Σίχ Ρούπερτ ε, από την ε, εταιρεία Consultants. Ευχαριστώ. Έχω μια παρουσίαση, ελπίζω να εμφανιστεί στην οθόνη. Τι είναι η Transforum. Είχαμε 7 προγράμματα σε δύο χρόνια και το σημαντικό που πρέπει να θυμάται κανείς για τα προγράμματα αυτά είναι ότι είχαμε συστηματικά διαβούλευση με όλους τους κλάδους μεταφορών από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. 127 εμπειρογνώμονες συμβουλευτήκαμε, είχαμε διάφορα εργαστήρια και στόχος μας ήταν να καταλάβουμε οι άνθρωποι επιτόπου πώς βλέπουν την εφαρμογή της Λευκής Βίβλου για τις μεταφορές ή εν πάση περιπτώσει τους στόχους της. Το κάναμε αυτό για δύο χρόνια λοιπόν όσον αφορά την καθαρή αστική κινητικότητα, τις ε, μεταφορές, ε, τις μεγάλες ε, εμπορευμάτων και τις συνδυασμένε μεταφορές, πώς γίνεται η διαχείρισή τους και η πληρωμή τους. Όπως επίσης ασχοληθήκαμε και με τα τρένα υψηλής ταχύτητας. Πρώτα απ' όλα λοιπόν πρέπει να δούμε πώς θα βελτιωθεί ο συντονισμός. Δεύτερον πρέπει να ε, βελτιώσουμε την αποτελεσματικότητα και τρίτον να δούμε την υποδομή. Για όλους τους μικρούς τομείς προσπαθήσαμε να δούμε σε ποιον από αυτούς τους τομείς πρέπει να επικεντρωθούμε περισσότερο. Δεν θα αναφερθώ σε αυτήν την διαφάνεια, έτσι καλώς δεν μπορείτε να τη διαβάσετε. Θα επικεντρωθώ περισσότερο σε δύο τομείς και επειδή έχουμε τόσο λίγα για τις αστικές συγκοινωνίες, εγώ θα επικεντρωθώ στις αστικές ε, συγκοινωνίες. Πώς μπορούμε να έχουμε καθαρές μεταφορές χωρίς διοξίδιο του άνθρακα στις πόλεις μας λοιπόν. Το πρώτο και σημαντικό πράγμα που πρέπει να έχουμε υπόψη μας ε, για τις ε, αστικές συγκοινωνίες και τους στόχους τους είναι ότι δεν Πρόκειται για τεχνολογική λύση, γιατί οι πόλεις διαφέρουν πολύ μεταξύ τους στην Ευρώπη και το πιο σημαντικό είναι οι τοπικοί παράγοντες να εγκρίνουν όποια πολιτική θεωρούν ότι μπορεί να προσαρμοστεί στις συγκεκριμένες τοπικές προϋποθέσεις που ισχύουν. Το πρώτο μήνυμα κλειδί λοιπόν για του αστικούς στόχου είναι ότι πρέπει να υπάρχει μια ανοιχτή προσέγγιση η οποία να επιτρέπει οι ευρωπαϊκοί στόχοι να ευθυγραμμίζονται με τα τοπικά ωφέλη. Έπειτα, αντικατάσταση οχημάτων και καυσίμων σίγουρα είναι σημαντικός στόχος, έτσι το βλέπουν ε, οι διάφοροι παράγοντες, δεν φτάνουν όμως. Χρειάζονται τοπικές λύσεις που να μπορούν οι πολίτες να εφαρμόσουν και αυτές είναι καλύτερη διασύνδεση και ολοκλήρωση των μεταφορών, να συνδυαστεί ο σχεδιασμός των μεταφορών με τη χρήση γης, να βελτιωθεί, ε, βελτιωθούν οι ηλεκτρικές δημόσιες μεταφορές, να προωθήσουμε περισσότερο το περπάτημα και το ποδήλατο για τις μεταφορές μας και ε, να ε, χρεώσουμε τους χρήστες των οδικών μεταφορών. Κατά πόσο τώρα είναι η κατάλληλη πολιτική στιγμή αυτή θα έπρεπε στα πλαίσια των σχεδίων για την ε, φοραστική μετακίνηση να έχουμε και εκστρατείες για συνειδητοποίηση. Πρέπει να βοηθήσουμε τις πόλεις να κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν και αυτό που θέλουν να κάνουν. Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις δηλαδή πρέπει να αναθερούν συνεχώς τις εθνικές τους πολιτικές προκειμένου οι πόλεις να μπορούν να συνεισφέρουν στους στόχους της Λευκής Βίβλου. Αυτό έχει να κάνει με προδιαγραφές, έχει να κάνει με χρηματοδότηση, αλλά οι εθνικές κυβερνήσεις επίσης πρέπει να μειώσουν τα φορολογικά αντικίνητρα και τα αντιπαραγωγικά ε, φορολογικά κίνητρα τα οποία ε, εφαρμόζουν και προτείνουν και να βελτιωθεί και το νομοθετικό πλαίσιο ώστε να μπορεί να υπάρχει ένα σύστημα που να πληρώνουν τα οχήματα τα οποία ρηπαίνουν περισσότερο. Οι πολιτικοί πρέπει να αναλάβουν τους κινδύνους ενός τέτοιου συστήματος. Τώρα, η γνώση είναι κάτι πολύ σημαντικό επίσης. Οι πολιτικές της πόλης είναι κάτι περίπλοκο και η γνώση μερικές φορές λείπει. Πώς δουλέψαμε εμείς στο δικό μας το πρόγραμμα Υπάρχει μια έκθεση, να Νάτι, που την έχουμε ετοιμάσει. Έφερα 10 αντίγραφα για τις αστικές μεταφορές. Υπάρχουν και στο διαδίκτυο και υπάρχουν και περιλήψεις, αν δεν έχετε χρόνο να το διαβάσετε ολόκληρο. Τι κάναμε λοιπόν. Αναπτύξαμε ένα χάρτη πορείας για το τι πρέπει να κάνει η Ευρώπη, τι πρέπει να κάνουν οι χώρες μέλη. Να, εδώ μερικά σημεία. Περιλαμβάνουμε επίσης και το τι πρέπει να κάνουν οι ίδιοι πολίτες. Είναι δηλαδή ένα πλήρες έγγραφο που ετοίμασαν οι διάφοροι φορείς με τη δικιά μας τη βοήθεια. Όσον αφορά λοιπόν τους αστικούς στόχους, μπορώ να πω ότι ο στόχος είναι εφικτός, καταρχήν, αλλά πρέπει να δράσουμε. Και όταν λέω να δράσουμε, ενώ οι χώρε μέλη. Ξέρω ότι δεν έχω περισσότερο χρόνο στη διάθεσή μου να μιλήσω για τις επορικές μεταφορές, τις ε, πιο μεγάλες. Δύο λύσεις πάντως υπάρχουν, που έχουν εντοπίσει δηλαδή οι φορείς συμπληρωματικές μεταξύ τους. Η μία είναι να δούμε τις επενδύσεις μεγάλης κλίμακας στις υποδομές, είναι προφανής, και το δεύτερο είναι να κοιτάξουμε ε, μικρές επεκτάσεις υποδομών που να εξυπηρετούν τις υπηρεσίες. Όταν λέμε ότι οι εμπορικές μεταφορές Ε, όταν είναι πάνω από 300 χιλιόμετρα πρέπει να φύγουν από τους δρόμους. Το ερώτημα που τίθεται είναι πώς θα γίνει αυτό. Έχουμε κάποιες ιδέες εμείς, δεν προλαβαίνω εδώ να σας τις παρουσιάσω όλες, αλλά το έγγραφό μας τα λέει όλα. Ευχαριστώ πολύ. Ακολουθεί ο κ. Χάινερ Μονχάιμ της ΡΑΜΚΟΜ, που είναι Ινστιτούτο για την Περιφερειακή Ανάπτυξη και την Επικοινωνία. Κυρίες και κύριοι, αγαπητέ Πρόεδρε, η δική μου προοπτική είναι αυτή των ευρωπαϊκών περιφερειών, δήμων και κοινοτήτων, δηλαδή κινητικότητα από κάτω προς τα πάνω. Το μεγάλο πεδίο είναι ε, τα διόδια που δεν το συζητούν. Τα κράτη-μέλη τα συζητούν αυτά περισσότερο με παλαιωμένο τρόπο με διάφορα σήματα κυκλοφορίας και σε πολύ τοπικό επίπεδο. Αν θέλουμε μία ευφύ στρατηγική ε, ε, διοδίων για τους Δήμους και τις κοινότητες, τότε θα έχουμε μια ευκαιρία γιατί αντιμετωπίζουν τεράστιο οικονομικό πρόβλημα στις μεταφορές οι Δήμοι και οι κοινότητες και θα λυθεί. Γιατί ε, η μεγαλύτερη μετακίνηση γίνεται στα αστικά και περιαστικά κέντρα. Τα αστικά διόδια υπάρχουν στη Σκανδιναβία και στο Λονδίνο. Κανονικά θα πρέπει να ε, δίνουν ε, ένα πλαίσιο, μάλλον να τους δοθεί ένα πλαίσιο σε όλη την Ευρώπη. Το δεύτερο φορά το Uber και το μπλα big data και FEE e κινητικότητα. Έχουμε από τη μια ένα τεράστιο δυναμικό σε αυτό το επίπεδο. Στη Γερμανία και μόνο κάθε μέρα 90 εκατομμύρια ε, και άδειες θέσεις οχημάτων κυκλοφορούν ε, στους δρόμους. Αν τα γεμίσουμε αυτά, εάν υπάρχει προσφορά ε, και συναντήσει τη ζήτηση για κινητικότητα, με τρόπο ευφύ έχουμε τεράστια ευκαιρία. Αλλά αυτό δεν μπορούμε να το αφήσουμε στην εταιρεία ε, Uber. Ε, χρειάζεται ένα πλαίσιο ε, που θα τα εξασφαλίζει όλα αυτά. Δεν θα πρέπει να είναι εμπορικά, να είναι νομικά νομοθετημένα με μια τιμολόγηση, με ασφαλιστική κάλυψη και όχι παράνομες διελεύσεις. Ένα τρίτο που ακούστηκε πολύ συχνά σήμερα είναι ο εξηλεκτρισμός της κίνησης. Ε, η κλασική ηλεκτρική κινητικότητα είναι το τραμ. Ορίστε ένα μέσο σταθερή ε, τροχιά ηλεκτρικό, χρειάζονται και αυτά μια αναγέννηση. Το τραμ να μην είναι μόνο μέσο σταθερή ε, τροχιά τοπικό για μεγάλε πόλει, αλλά έχουμε μακρά πύρα και σε μικρές πόλεις και σε μεσαίου μεγέθους πόλεις υπήρχαν τραμ. Χρειάζεται μια αναγέννηση. Και επίσης ο περιαστικός σιδηρόδρομος, προαστιακός. Ε, επειδή ε, όμως ε, αυτά τα συστήματα, τα τρόλεϊ, τα ηλεκτροκίνητα έχουν καλώδια στον αέρα, πρέπει να βρούμε ένα άλλο σύστημα με συσσωρευτές, με μπαταρίες. Το Μπορντό πρωτοτυπεί σε αυτή τη περίπτωση και πρωτοστατεί. Χρειαζόμαστε ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα έρευνας και επενδύσεων. Ένα τεράστιο πρόβλημα είναι ε, η ε, τοπική κυκλοφορία στις παραμεθόριες περιοχές. Υπάρχουν δύο ευρωπαϊκά δίκτυα, μεγάλοι διάδρομοι που μας απασχολούν, αλλά υπάρχει καθημερινή κινητικότητα των εργαζομένων που δουλεύουν 20 χιλιόμετρα δεξιά των συνόρων και ζουν 30 χιλιόμετρα δεξιά των συνόρων. Ε, χρειαζόμαστε μια στρατηγική για την τοπική κυκλοφορία. Αυτοί οι άνθρωποι περνάνε τη μέρα τους μέσα σε ε, μποτιλιαρίσματα. Υπήρχαν ε, τραμ και τοπικά τρένα ε, στις παραμεθορίους της Ευρώπης, τα οποία τα καταργήσαμε και τα ξυλώσαμε. Αυτό θα πρέπει να ανανεωθεί. Ένα άλλο θέμα ε, είναι κάτι που μπορεί να μας διδάξει πολύ η Σκανδιναβία. Οι δημόσιες συγκοινωνίες ε, παραδοσιακά ε, ήταν συνδυασμένες μεταφορές επιβατών και εμπορευματικές. Πάντα το ταχυδρομείο, είχε, ακόμα και η τραχυδρομική άμαξα μετέφερε και επιβάτες και ε, εμπορεύματα. Το έχουμε στο αεροπλάνο, επάνω επιβάτες κάτω τα εμπορεύματα. Στη Φιλανδία, στη Σουηδία, μέχρι και τα λεωφορεία μεταφέρουν και επιβάτες και εμπορεύματα. Αυτό είναι η ευκαιρία πραγματικά να τονωθούν οι συγκοινωνίες και να είναι πιο αποδοτικές στην Ήπεθρο η Φιλανδία και η Σουηδία που είναι πολύ αεροκατοικημένες έχουν ε, κάθε μισή ώρα λεωφορείο. Google Car, επόμενο θέμα από τη μια μας λένε οι κατασκευαστές των αυτοκινήτων ότι έχουν τεράστιες δυνατότητες, φανταστικές, με αυτοκίνητα αυτόματα που οδηγούν μόνα τους. Από την άλλη, οι κυβερνήσεις και οι δήμοι και οι κοινότητες είναι τελείως επιφυλακτικοί, δεν θέλουν να αξιοποιήσουν αυτή την ευκαιρία. Δεν θέλουμε μόνο έξυπνα αυτοκίνητα που να οδηγούν μόνα τους, αλλά θέλουμε και έξυπνους δρόμους για να το καταλαβαίνουν, να βγάλουμε όλα τα εμπόδια ε, και όλα τα νομοθετικά μέτρα που είναι περιτά και άχρηστα, αν είναι οι δρόμοι μας ευφυείς. Και να ρωτάμε τους πολίτες, εδώ που θα περνάει ένα αυτοκίνητο από μπροστά σου, με ποια ταχύτητα, ε, θα είναι τηλεκατευθυνόμενο, θα επιτρέπεται να βαρκάρει, όχι, και αυτό θα είναι τηλεκατευθυνόμενο. Θα πρέπει η τοπική αυτοδιοίκηση, οι δήμοι και οι κοινότητες να έχουν αυτή την ευκαιρία να αξιοποιήσουν το αυτοκίνητο της Google χρειαζόμαστε και μια επανάσταση στα συστήματα τιμολόγησης. Η Ευρώπη είναι μια ε, ζούγκλα ε, μικροτιμολογήσεων στις ε, συγκοινωνίες. Κανείς δεν τα ξέρει αυτά. Τι, υπάρχουν παραδείγματα από την Ελβετία που έχουν ένα, μια γενική κάρτα σύνδρομης ή στη Γερμανία που έχουμε ένα πάσο διάρκειας 6 μηνών. στη Γερμανία καταφέραμε να μην κυκλοφορούν με τα αυτοκίνητα οι φοιτητέ, αλλά με τα μέσα μαζικής μεταφορές γιατί έχουν ένα πάσο ε, ε, με ενιαία τιμή εισιτηρίου, flat rate και λογική. Χρειαζόμαστε ένα εισιτήριο για τον πολίτη σε όλα τα ευρωπαϊκά κράτη και νομοθετικό πλαίσιο. Θα το δώσουμε στην Ευρώπη και μετά οι εθνικές κυβερνήσεις να ε, το εφαρμόσουν. Και τελικά αυτό που χρειαζόμαστε για τις μαζικές συγκοινωνίες και μεταφορές. Ε, ξέρουμε όταν θες να φτιάξει ένα νέο τραμ, μια νέα διαδρομή χρειάζεται 10 χρόνια. Υπάρχουν ε, συστήματα ε, όμως τελεφερικ που είναι ε, ηλεκτροκίνητα. Η Λαπά στη Βολιβία μας δείχνει πώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Ε, μπορείς να έχεις και συγκοινωνία με τελεφερικ. Δεν είναι ανάγκη να είναι τραμ. Ε, υπάρχει και αστικό τελεφερικ το τελευταίο. Ε, στη δεκαετία του 80 και 90 τεράστιο πρόβλημα ήταν ε, ο, ο θόρυβος. Σήμερα ε, μιλάμε για πρόθεση του ποδηλάτου, για αυτοκίνητα που θα τα μοιραζόμαστε και συνδυασμένη κινητικότητα. Είναι πολλά τα τοπικά πειράματα και χρειάζεται μια εθνική ε, ομπρέλα ας πούμε. κάποιες χώρες έχουν προγράμματα εθνικά για το ποδήλατο είναι πραγματικά ο φτωχό συγγενή, εξαιρετικά οι πεζοί και οι με την κακώ νοούμενη έννοια τη επικουρικότητα. Σου λέει η εθνική κυβέρνηση αυτό είναι θέμα του Δήμου. Ναι, αλλά το πλαίσιο για τον ποδηλάτη και για τον πεζό ε, θα πρέπει να είναι υποχρεωτικά εθνική υπόθεση και γι' αυτό θα πρέπει η Ευρώπη να ανοίξει νέες προοπτικές. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Η Ζόνκια Χάικελ έχει τώρα το λόγο από το ΤΕΚΕΣ, το Ίδρυμα της ε, Φιλανδίας για την Καινοτομία και την Ανανέωση. Ευχαριστώ Πρόεδρε, είμαι η Σόνια Χέκελε και όντω εργάζομαι και το ΤΕΚΕ, την ε, Φιλανδική, το Φιλανδικό Ίδρυμα για την Καινοτομία. Ε, φέτος την Άνοιξη θα χρηματοδοτήσουμε καινοτόμες ιδέες που προωθούν την αποτελεσματικότητα ραντάρ στις μεταφορές με λύσεις που μπορεί να αλλάξουν την συμπεριφορά των ανθρώπων στις μεταφορές και έτσι να στηρίξουν την ε, βιωσιμότητα. Οι προκλήσεις στο σημερινό σύστημα μεταφορών είναι προφανείς. Χρειάζονται βελτιώσεις βεβαίως, πέραν αυτών που έχουν επιτευχθεί ήδη σε κάποιους τομείς, όπως η τεχνολογία των οχημάτων, αλλά δεν εξαρκούν όσο έχουν γίνει. Πρέπει να γίνουν πολύ περισσότερα. Καταρχάς, έχουμε τεράστιο ρυθμό αυτοκινήτων. Όμω αυτά τα οχήματα χρησιμοποιούνται αναποτελεσματικά. Χρησιμοποιούνται μόνο κατά 5% όπως θα έπρεπε. Τον υπόλοιπο καιρό παραμένουν σταθμευμένα. Δεύτερο μεγάλο θέμα, ε, δεύτερη μεγάλη δαπάνη των οικοκυριών είναι τα αυτοκίνητα μετά την ε, στέγαση. Είναι μεγάλη επένδυση λοιπόν τα οχήματα, αλλά δυστυχώς τα γιοταχή είναι ακόμα πολύ δημοφιλή. Γι' αυτό δεν έχουμε βρει ακόμη αρκετές εναλλακτικέ για την οδήγηση και την, την αυτοκινήτου. Βεβαίω όχι μόνο για τους χρήστες, αλλά και για τι δημόσιες επενδύσεις η κάλυψη των αναγκών των, των είναι μεγάλη δαπάνη. Η κατάσταση ακόμα είναι ε, κάπως ασταθής και δεν υπάρχει αρκετή καλή συντήρηση του οδικού δικτύου, ακόμη λιγότερο του συστήματος μεταφορών. Πρέπει λοιπόν να υπάρξει η κατάλληλη διασύνδεση, αλλά δεν υπάρχει δημόσια χρηματοδότηση της διαμετακόμισης ή η επέκτασή της. Η μόνη λύση λοιπόν για να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα του συστήματος μεταφορών είναι να βελτιώσουμε τη συνολική αποτελεσματικότητά του. Όχι μόνο τις δυνατότητες του συστήματος οι προκλήσεις στις μεταφορές είναι τόσο μεγάλες και είναι τόσο μικρές οι βελτιώσεις μας ως τώρα που πρέπει να κάνουμε κάτι πιο ριζοσπαστικό. Η κατάσταση θα μπορούσε να είναι πολύ καλύτερη αρκεί κάποιες από τις τάσεις που εμφανίζονται στην κοινωνία και επηρεάζουν τις μεταφορές να ε, αξιοποιηθούν γιατί οδηγούν ήδη στην βιωσιμότητα. Θα έπρεπε απλώς να δώσουμε στις τάσεις αυτές το περιθώριο να, ε, να ανθίσουν και να ε, πολλαπλασιαστούν, να διαδοθούν. Στους νέους λόγου χάρη υπάρχει η αντίληψη ε, ότι η διοκτησία αυτοκινήτου έχει μεγάλη επίπτωση στις μεταφορές. Προτιμούν αν έχουν εναλλακτικό τρόπο μεταφοράς να το χρησιμοποιήσουν. Η, ψηφιοποίηση έχει διαδοθεί στις περισσότερες βιομηχανίες και εταιρείε. Και συνήθως δεν υπάρχει άλλος τρόπος ε, παροχής υπηρεσιών παρά μόνο επιγραμμικός. Οι επιγραμμικές υπηρεσίες δεν θα ήταν... Μπορεί μάλλον έτσι να γίνουν δημοφιλείς και να επηρεάσουν τελικά κατά τη συμπεριφορά των ανθρώπων. Η πολλαπλή χρήση μέσων είναι ίσως ε, ο τρόπος που θα γίνει κάποια στιγμή φυσικός οι μεταφορές λοιπόν θα πρέπει να περάσουν από την ιδιοκτησία στην χρήση. Αυτή είναι η βασική αλλαγή στην συμπεριφορά και την οτροπία. Είναι πάρα πολλά τα αυτοκίνητα όπως είπα, αλλά θα ήταν διαφορετικό αν ήταν αξιοποιήσιμα και προσβατά σε όλους. Επίσης πρέπει να γίνει η βιωσιμότητα πιο ελκυστική, δηλαδή σε χαμηλές τιμές, ανταγωνιστικές και με εύκολη πρόσβαση η ευκολία της χρήσης είναι από τα σημαντικότερα όταν μιλάμε για τις μεταφορές. Το γνωρίζουμε ε, γιατί χρησιμοποιούμε μεταφορές όλοι καθημερινά. Γι' αυτό το λόγο στη Φινλανδία έχουμε προβλέψει μία λύση που, ονομάζουμε ε, ε, υπηρεσίες κινητικότητας με μεγάλη με μεγάλο δυναμικό να μετατρέψουν τον κλάδο των μεταφορών. Αυτός αυτή είναι η φιλοδοξία που τρέφουμε. Μιλάμε για υπηρεσίε κινητικότητα που αξιοποιούν όλα τα μέσα μεταφορά, όλου του τρόπου μεταφορά, με τη συμμετοχή των παραγόντων, των εταιριών μεταφορών και για του χρήστε να υπάρχει δυνατότητα ε, επιλογή τη πλέον πρακτική λύση μεταφορά στην περίπτωσή του. Έτσι, η κινητικότητα ω υπηρεσία θα αυξήσει την αποτελεσματικότητα του συστήματο μεταφορών, καθώ οι εταιρείε θα έχουν το περιθώριο να αντιμετωπίσουν σωστά το κόστος και να οργανώσουν σωστά τις υπηρεσίες μεταφορών. Όμως, για να είμαστε και πραγματιστές, οι υπηρεσίες κινητικότητας οπωσδήποτε χρειάζεται να έχουν συμμετοχή και από τον ιδιωτικό τομέα αλλά και πρωτοβουλία από τον κρατικό με την ε, διευκόλυνση και την ενδυνάμωση. Ναι, να σας ευχαριστήσω και να ανυπομονώ για τη συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ. Ακολουθεί η συζήτηση ακριβώς και οι ερωτήσει. Πρώτος ο Βιν Βανεκάμπ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δύο ερωτήσεις έχω προς τον Γιος Ντίνγκς. Πρώτα για τον καθορισμό των προδιαγραφών. Έχουμε αρκετές προδιαγραφές, τις έχουμε καθορίσει. Η λευκή δίβλος του 2011 επαρκεί, πρέπει να έχουμε πιο αυστηρές προδιαγραφές. Λέτε ότι με το ΣΥΠΙΚ δεν έχουμε. Με εκπλήσει βέβαια λίγο, γιατί πάντα είχαμε και προσπαθούσαμε να πετύχουμε τις πιο καθαρές μεταφορές. Δεύτερον, όσον αφορά τις ηλεκτρικές μεταφορές, τον εξηλεκτρισμό των μεταφορών. Από πού θα έρθει ο ηλεκτρισμός αυτός. Στην Ολλανδία ξέρουμε ότι η Γαλλία θέλει μόνο πυρηνική ενέργεια. Εσείς πώς βλέπετε αυτό το θέμα του ηλεκτρισμού, από πού θα μας έρθει. Τώρα προς τον κύριο Ρούπερ. Ρούπρεχτ. Επίσης θέλω να σας ρωτήσω από πού θα προέρθει ο ηλεκτρισμός, η ηλεκτρική ενέργεια. Τον κύριο Μούνχαιμ τώρα και την κυρία Χαϊκίλα. <laughs> Δεν προφέρω καλά το όνομά σας, εσείς το ξέρετε, με καταλάβατε. <laughs> Το μικρό σας. Σόνια. Α, ωραία. Ερώτηση λοιπόν προς τη ναι. Σόνια. Κυρίως... Α, όχι, ολλανδικά θα μιλάω. Στον κύριο Μόνχαμ λοιπόν και την κυρία Χακίλε θέλω να ρωτήσω. Και ο ιδιωτικό τομέα τι ρόλο Εγώ δεν έχω αυτοκίνητο. Ζω όμως σε μια πόλη. Πολλοί Ευρωπαίοι όμως ζουν στην Ήπεθρο. Και εντάξει, είναι πολύ ωραία τα ωραία λόγια για το να μοιραζόμαστε τα αυτοκίνητα. Ναι, τι θα κάνω εγώ αν πρέπει να βάλω τα παιδιά μου στο σχολείο. Πρέπει να χρησιμοποιήσω το αυτοκίνητό μου. Θα μου πείτε ότι είναι παλιωμοδίτικος αυτός ο τρόπος σκέψης. Ωραία, πείτε μου το δικό σας. Ο ρόλος του ιδιωτικού αυτοκινήτου, ποιος είναι, του γιοταχή δηλαδή, πώς το βλέπετε εσείς. Κλάδια Παπαντέλ. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρε, είναι αλήθεια ότι το τμήμα αυτό της Λευκής Βίβλου που έχει να κάνει με τις βιώσιμες μεταφορές και τον ε, εξηλεκτρισμό είναι πολύ καλά. Εγώ θέλω να αναφερθώ στην αρχή το ρηπαίνο πληρώνει. Πώς μπορούμε να έχουμε ολοκληρωμένα συστήματα για την πληρωμή, ώστε τα χρήματα αυτά που πληρώνουν οι ρηπαίνοντες, τα χρήματα αυτά πράγματι να χρησιμοποιούνται για την προστασία του περιβάλλοντος. Μ' άρεσε η παρουσίαση του κυρίου Μονχάιμ. Είμαι ενθουσιώδης γιατί έχω εμπειρία στην τοπική δίκηση. Ρωτώ όμως πώς μπορούμε να έχουμε ένα τέτοιο ολοκληρωμένο σύστημα μεταφορών και για τους χρήστες. Πώς μπορούμε να προσφέρουμε αυτό το ενιαίο εισιτήριο, για παράδειγμα, το οποίο στηρίζω πλήρως και το οποίο θα μπορούσε πράγματι να χρησιμοποιηθεί για όλα τα μέσα μεταφοράς, αλλά και για πάρκινγκ, για στάθμευση. Πώς μπορεί όμως να εφαρμοστεί κάτι τέτοιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς εμείς μπορούμε να στηρίξουμε τις τοπικές αρχές. Έχουμε την αρχή της επικουρικότητας και η πιο αποτελεσματική μέθοδος είναι αυτή η οποία πρέπει να εφαρμόσετε για τον καθένα. Και τελευταία μου ερώτηση είναι για τη Σόνια. Και το δικό μου το όνομα είναι περίπλοκο. Λοιπόν, δεν ξέρω αν σας κατάλαβα καλά, αλλά είπατε ότι πρόκειται για 300 ευρώ για κάθε οικογένεια το μήνα ή για κάθε άτομο και ότι με αυτή την πληρωμή των 300 ευρώ ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιεί διάφορα μέσα μεταφοράς δεν ξέρω αν σας κατάλαβα καλά. Αυτό είναι το σχέδιο. Μπορείτε να μας το εξηγήσετε παρακαλώ καλύτερα. Γιατί εδώ πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι άλλες χώρες έχουν χαμηλότερα εισοδήματα. Και δεν ξέρω αν ένας συνήθις χρήστης μπορεί να αντέξει να πληρώνει 300 ευρώ το μήνα για τέτοιου είδους υπηρεσίες μεταφοράς. Είναι πάντως μια πολύ καλή λύση, αλλά να ρωτιέμαι πώς θα μπορούσε να εφαρμοστεί σε όλες τις χώρες μέλη, δεδομένου ότι το κόστος ζωής είναι διαφορετικό από χώρα σε χώρα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, Ζήνε Μάισνερ. Ευχαριστώ. Τώρα θα το κάνω αλλιώς. Έχω πολλές ερωτήσεις που δεν είναι για ειδικό μιλήτη. Σύμφωνο με την προλαλή σας για το ενιαίο εισιτήριο. Πώς μπορούμε να μάθουμε. Υπάρχει μια πλατφόρμα για ανταλλαγή. Είναι ένα θέμα επικουρικότητας θα μου πείτε, αλλά γνωρίζω ότι στο Αμβούργο λειτουργεί θαυμάσια. Ε, δίνεις ε, την αφετηρία και τον προορισμό σου και σου δίνουν ένα δρομολόγιο. Και στο Λονδίνο το έχω δει, φαντάζομαι και σε άλλες πόλεις. Για το ενιαίο εισιτήριο για διάφορα μέσα μεταφοράς. Μπορούμε να διδαχθούμε ένας από τον άλλον. Γιατί δεν λέμε τόσα πολλά για τα ηλεκτρονικά, ηλεκτρικά ε, ποδήλατα. Δεν μιλάω για το τιμολόγιο, αλλά για την κινητικότητα στις πόλεις. Ε, μου άρεσε αυτό που αναφέρθηκε για τα τελεφερίκ, γιατί στην αρχή ε, νόμιζα ότι θα τα έλεγε ο, ο κύριος εκπροσωπεί το Ρούπρεχτ, ο κύριος Ρούπρεχτ, αλλά ο κύριος Μόνχαιμ το είπε στη συνέχεια. Ε, είναι ένα πολύ ε, νέο καινοτόμο μέσο μεταφοράς, φιλικό στο περιβάλλον, δεν είναι πανάκι, αλλά θα μπορούσε να συζητηθεί. Και πάλι για τον κύριο Μόνχαιμ, ε, έχω την ίδια αίσθηση με τον κύριο Βάντεν Κάμπ. Αν είναι όλα αυτά τόσο ρυθμισμένα και ηλεκτρονικά ε, και τηλεκατευθυνόμενα, μέχρι και για το παρκάρισμα δεν περιορίζεται η ασφάλεια, η, ελευθερία των ανθρώπων. Εντάξει, μπορεί να είναι η πόλη πιο ασφαλής, δεν έχει συμφόρηση, αλλά δεν έχει κάποιο αυτόβουλο ο κόσμος και ελεύθερα να αποφασίζει και για την κυρία Χέκαλ από την Φιλανδία. Ε, πολύ ενδιαφέρον αυτό που είπατε, το έχετε συζητήσει με άλλες χώρες, μπορεί να μεταφερθεί σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πώς το βλέπετε. Ευχαριστώ πολύ. Μαρία Κίλωνεν. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, ευχαριστώ όλους όσοι πήραν το λόγο για τις παρουσιάσεις τους. Δύο ερωτήσεις έχω. Και ο καθένας από εσά μπορεί να απαντήσει. Πρώτον, τι δυνατότητες βλέπετε σε εθνικό ή σε διεθνές επίπεδο όσον αφορά ένα ευρωπαϊκό σύστημα μεταφορών που να είναι αποτελεσματικό και ευφυές. Επίσης, τι γίνεται με τις υπηρεσίες κινητικότητας, mobility services. Πώς μπορούμε επίσης να εφαρμόσουμε ε, αυτό το νέο σύστημα και πότε, αμέσως ή σε 10 χρόνια το βλέπετε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Λέει ο κύριος Κλέτς. Πολύ καλές παρουσιάσεις κάνατε. Και μας παρουσιάσατε οράματα όσον αφορά τις μεταφορές, ιδίως η τελευταία παρουσίαση. σε όλες όμως τις εκθέσεις της Επιτροπής των Εμπειρογνώμων οι μεταφορές είναι από τους κλάδους που αγνούν κάπως τις προσπαθειές μας για μείωση του διοξιδίου του άνθρακα εν ώψη του 2020-2030. Οπότε, πώς η πολιτική μεταφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να οδηγήσει στην προστασία του περιβάλλοντος και σε χαμηλότερες εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα ώστε να πετύχουμε περισσότερα πράγματα στο κοπήκωση του Παρισιού. Η πολιτική μεταφορών είναι κάτι για τους νέους, όχι για τους πιο μεγάλους. Και σήμερα βλέπουμε ότι περισσότερες από τις προτάσεις πρέπει να ανταποκρίνονται στις επιθυμίες και τις ανάγκες των νέων. Οπότε, τι έχετε να συστήσετε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Συμβούλιο, το Κοινοβούλιο ως πρώτη προτεραιότητα για αλλαγές στην Λευκή Βίβλο. Αυτές ήταν οι ερωτήσεις, απαντήσεις. Με την ίδια σειρά, ε, την αντίστροφη δηλαδή, παρακαλώ. Ο κύριος Δίνξ. Δεν ξέρω ποιες ερωτήσεις ήταν για μένα εκτός από αυτές του κύριου Φαντεκάμπ. Διαλέγω λοιπόν για μεταφορές και κλίμα. Ναι, το COP21 φυσικά και πρέπει να το έχουμε υπόψη μας. Οι πλωτέ μεταφορές και οι αεροπορικές μεταφορές είναι αυτές που πρέπει να κοιτάξουμε περισσότερο οι εκπομπές των κλάδων αυτών λιγάκι εξαφανίζονται χωρίς να προβαίνουμε σε πραγματικές αλλαγές. Εξαφανίζονται σε μια μαύρη τρύπα δηλαδή. Ρωτάτε για προδιαγραφές. Αν δείτε την ρήπανση του αέρα από τα φορτηγά, από τα αυτοκίνητα. Δείτε ποιες είναι οι προδιαγραφές, τα παραρτήματα που όλοι σας διαπραγματευτήκατε. Βλέπουμε πολύ χαμηλά νούμερα. Θα σκεφτόταν κανείς, καλά τα πάμε. Και όμως, ακόμα διαπραγματευόμαστε το μικρό γάμα, το μικρό δέλτα και γιατί. Γιατί τα νούμερα αυτά δεν τα βλέπουμε στους δρόμους. Άρα ε, χρειάζονται διορθώσεις ώστε στην πράξη να έχουμε τα σωστά αποτελέσματα. Για την ενέργεια και το διοξίδιο του άνθρακα, που είναι μεγάλη πρόκληση για τις επόμενες δεκαετίες, δεν υπάρχουν ε, καλές προδιαγραφές, αρκετά αποτελεσματικές προδιαγραφές. Πρέπει να κάνουμε πολύ περισσότερα. Παντού και για όλα, και για τα αεροπλάνα, και για τα σκάφη, και για τις οδικές μεταφορές. Υπάρχουν μελέτες που δείχνουν ότι πριν από μερικές δεκαετίες τα πλοία ήταν εξίσου αποτελεσματικό όπως και σήμερα. Υπήρχε διαφορετικός σχεδιασμός. Άρα μένουν πολλά να γίνουν για όλα τα είδη μεταφορών. Από πού θα έρθει ο ηλεκτρισμός? Πολύ καλή ερώτηση. Ε, με πολλούς τρόπους μπορεί κανείς και μάλιστα βρώμικους τρόπους να παράγει ηλεκτρισμό που ρηπαίνουν. Αλλά το πετρέλαιο βλέπουμε ότι ρηπαίνει όλο και περισσότερο. Γιατί, γιατί πάμε στην Αρκτική, γιατί πρέπει να κάνουμε εξορίξεις από ακόμα πιο βαθιά. 70% του ηλεκτρισμού ότι να έρχεται από τις αναλλακτικές πηγές ενέργειας. Πρέπει να δούμε τι περιμένουμε στα επόμενα 20-30 χρόνια. Η πυρηνική ενέργεια γίνεται πιο καθαρή. Δεν ισχύει το ίδιο στο πετρέλαιο όμως, στα ορυκτά καύσιμα. Έτσι είναι. Τι να κάνω. Για το νέο Πολύ καλό παράδειγμα. Όντω, πολλέ πόλει το έχουν εφαρμόσει και μερικέ χώρε, αλλά χρειάζεται ρύθμιση, όντω. Και ναι, τα ηλεκτρικά ποδήλατα μπορούν να βοηθήσουν να καλύψουν το χάσμα ανάμεσα σε αυτό που κάνουν τα σημερινά ποδήλατα, τα μη ηλεκτρικά δηλαδή, και αυτά που μπορεί να κάνει ο ποδηλάτης. Νομίζω ότι το πλαίσιο υπάρχει σήμερα δεν είναι αρκετά καλό. Όταν μιλάμε για οικονομικά κίνητρα, επιδοτήσεις και τα λοιπά δεν ακούγονται αρκετά, αλλά είναι ένας στο μέσα αυτός. Ευχαριστώ. Δεν είδα το Ζος Μπαχ που ήθελε να κάνει ερώτηση. Αν κάνει μια ερώτηση προς τους υπολείπους τρεις, καλώς. Και του δίνω το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ε, το ξέρω, είμαι τόσο μικρός, όμως είναι εύκολο να μην με δείτε. Ε, όχι, έχω κάνει μια ερώτηση για το πάνελ γενικά, που μου άφησε πολύ καλή εντύπωση όλες οι τοποθετήσεις πολλές προτάσεις λύσεις που κατατέθηκαν εδώ απαιτούν αλλαγή νοοτροπίας. Και αυτή η αλλαγή νοοτροπίας, να φύγουμε από την κλασική κυκλοφορία και να πάμε σε εναλλακτικά συστήματα μετακινήσεων, θέλω να ρωτήσω το παν. Αρκεί να υπάρχει καλύτερη προσφορά για να γίνει αυτό ή χρειάζεται πολιτική επέμβαση, να πάρουμε πολιτικές αποφάσεις. Και αν ναι, <laughs> κλασικές μέθοδοι ποιες είναι. Πρώτον διόδια ή κρατικές ενισχύσεις, κίνητρα. Φόβητρο ή κίνητρο. Οι κρατικές ενισχύσεις το τελευταίο διάστημα γνώρισαν τα όρια τους γιατί είναι πάρα πολύ σφιχτοί οι προϋπολογισμοί. Πώς το βλέπετε, ή αρκεί απλώς να είναι καλύτερη προσφορά σε όλα τα συστήματα συγκοινωνιών για να τα παίρνει ο κόσμος. Ε, κύριος Ρούπριχτ. Έχω λίγο περδευτεί με τις γλώσσες. Τι να μιλήσω. Αγγλικά. That's part of the confusion. Είναι και αυτό μέρος της σύγχυσης, αλλά αφού άρχισα αγγλικά, συνεχίσω αγγλικά. Από πού προέρχεται το ηλεκτρικό ρεύμα. Να συνεχίσω από εκεί που σταμάτησε ο Γιος Ντίνγκς δεν μιλήσαμε για τη μεγαλύτερη πηγή ενέργειας. Η μεγαλύτερη πηγή ενέργειας είναι η ενέργεια που εξοικονομούμε και δεν χρησιμοποιούμε. 30% ίσως και παραπάνω μπορεί να προκύψει από εξοικονόμηση ενέργειας. Ένα δεύτερο στοιχείο που δεν αναφέρουμε είναι οι συνέργειες που θα δημιουργήσουμε για την εξοικονόμηση και πάλι ενέργειας για να μειωθεί το συνολικό κόστος παροχής, ας πούμε στις αστικές μεταφορές, μετρό, τραμ, τρόλεϊ, ε, σε κάποιες πόλεις δίνουν ε, μια ε, συνολική υποδομή ηλεκτρική. Δεν χρειάζεται να επανεφευρίσκουμε τον τροχό όταν μιλάμε για ηλεκτροκίνητα, αυτοκίνητα υπάρχει αυτή η γνώση, μπορεί να μεταφερθεί ή ακόμα και να διασυνδεθούν τα τεχνικά συστήματα. Πού είναι λοιπόν οι συνέργειες ανάμεσα στα ηλεκτροκίνητα μέσα μαζικής μεταφοράς και στα νέα ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα, τα FEE συστήματα. Αυτά θα πρέπει να τα ε, συμπεριλάβουμε και τα ηλεκτρικά ποδήλατα οπωσδήποτε. Στην πόλη είναι πραγματικά, πώς να το πω, αναπόσταστο τμήμα ε, συνδυασμένων μεταφορών. Έχετε συμβατικά ε, ποδήλατα, ηλεκτρικά ποδήλατα, αυτοκίνητα που μπορείτε να μοιράζεστε, δημόσια συγκοινωνία. Υπάρχουν πόλεις αντιβρέμοι που ε, βάζουν πολύ μεγάλη έμφαση σε αυτό και θα πρέπει να γίνει πραγματικότητα σε πολλές πόλεις. Όταν μιλάμε για συνδυασμένες μεταφορές, τι σημαίνει αυτό. στις δημόσιες συγκοινωνίες υπάρχει και στις πόλεις ανταγωνισμός για τη χρήση του χώρου. Και είναι και ένα τμήμα της νέας συμφωνίας ενός New Deal για το πώς θα κατανέμουμε το κόστος, το χώρο στην πόλη και τη χρήση. Γιατί κάποιες μη αποδοτικές συγκοινωνίες ε, να κυκλοφορούν άδειε, ενώ μπορούν τα δύο τρίτα του χώρου που μπορεί, ενώ καταλαμβάνουν μάλλον τα δύο τρίτα του χώρου που προσφέρει μία πόλη. Το θέμα του κόστους. Γιατί μακροπρόθεσμα να μην συμπεριλάβουμε και τις αστικές συγκοινωνίε σε ένα τροποποιημένο σύστημα εμπορίας εκπομπών ρήπων. Πέραν του ορυπαίνων πληρώνει υπάρχουν ιδέες για το πώς μπορούν οι ιδιωτικές επενδύσεις εκεί να ε, ενταχθούν. Για, η πρώτη μου ευχή θα ήταν να μην ξεχνάμε τις αστικές μεταφορές. Εκεί είναι τα προβλήματα και εκεί μπορούν να βρεθούν οι λύσεις. Και πρέπει. Και μια που είμαι σε αυτό το τομέα μπορεί να σας εκπλήξει. Θα πρέπει να σκεφτούμε πώς να δημιουργήσουμε μια κουλτούρα αλλαγής. Μια νοοτροπία να δανειζόμαστε τις βέλτιστες πρακτικές με, με δικτύωση, με πόλεις που να συνεργάζονται. Δεν είναι πολύ ακριβό, είναι ίσα ίσα φτηνό αυτό, και, αλλά έχει πολύ μεγάλα αποτελέσματα. Ευχαριστώ. Χάιν, ε, ε, κύριος Μονχάιμ, Ράινερ, αρχίζω από τον κύριο Βάντεν Κάπ. Πόσα αυτοκίνητα χρειάζεται η Ευρώπη. 10% του σημερινού στόλου ε, οχημάτων αρκούν για να κινείται η Ευρώπη. 10% το 1 δέκατο των όσων έχουμε. Το δεύτερο, τι γίνεται με την Ήπεθρο που ρωτήσατε. Η Ήπεθρο στη δεκαετία του 50 σε όλη την Ευρώπη ήταν ε, ε, ο χώρος ε, που ε, ο κόσμος μετακινείται με δημόσια συγκοινωνία γιατί δεν είχε αυτοκίνητο. Α, άρχισε να αγοράζει ε, αργότερα. Και μάλιστα στην δεκαετία του 50 ανθούσε και το auto stop. Στην Ελβετία παντού και στο τελευταίο χωριό υπάρχει δυνατότητα να μοιραστεί αυτοκίνητο. Δηλαδή ακόμα και το χωριό δεν χρειάζεται να είναι χωρίς καμία συγκοινωνία. Ε, η Ελβετία και πάλι έχει ένα, μια γενική συνδρομή για όλα τα μέσα μεταφορών, ό,τι έχει. Ε, αυτοκίνητα, αεροπλάνα, βαπόρια, όχι αεροπλάνα, ε, ε τρόλεϊ, τελεφερή και ε, στις λίμνες. Δεν βγάζεις κάθε μέρα ένα εισιτήριο ενιαίο, είναι τίσιο. Έχεις μια συνδρομή. Είναι τεράστια η απήχηση του κόσμου. Και να πάμε στη διπλανή χώρα, ε, στην Αυστρία, στη Βιέννη, 365 ευρώ ε, το χρόνο, ένα ευρώ το κεφάλι την ημέρα για να μπορεί να κυκλοφορεί σε όλη τη Βιέννη με όσα τα μέσα μεταφοράς. Χρειάζεται μια στρατηγική ε, που να αλλάξει. Στη Γερμανία έχουμε εξαμηνιαία συνδρομή, ένα ειστήριο για έξι μήνες. Bike sharing, ε, ποδήλατα που τα μοιράζεσαι, αυτοκίνητα που τα μοιράζεσαι. Είναι συνδυασμένες μεταφορές, όχι μόνο οι δημόσιες κοινωνίες, όλα τα μέσα μεταφορά πολυτροπικό. Ανήκει εδώ φυσικά και το ηλεκτρικό ε, ποδήλατο και ε, τα καινοτόμα συστήματα έχουν εντάξει 10% ε, των ποδηλάτων και έρχομαι στην ερώτηση να κάνει η Ευρώπη. 45 χρόνια έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου. Έχω συμμετάσχει σε διάφορα ευρωπαϊκά έργα. Και είναι πολύ κουραστικό. Τρία χρόνια κάνουμε βέλτιστες πρακτικές, μαζεύουμε 30 θαυμάσια παραδείγματα, γράφουμε έκθεση και καμία εθνική πολιτική δεν μας δίνει σημασία. Ε, κάτω ανθεί το λιβάδι της καινοτομίας και πάνω είναι όλα ε, τα ίδια. Η Γερμανία δεν έχει καταφέρει ακόμα να φτιάξει μία στάση, ένα, μία πιάτσα, εν για να μοιράζει το κόσμο σε ένα αυτοκίνητο. Είναι πάρα πολύ νοθρές και χαλαρές οι διαδικασίες. Η Ευρώπη θα πρέπει να ταράξει τα νερά, να κουνήσει λίγο τα πράγματα για να γίνει κάποια στιγμή πολιτική ιδέα του κόσμου. Αυτά έχουν να κάνουν και με τα τελεφέρικ η Ευρώπη, πολύ ωραίο παράδειγμα, έχει οδηγία ολόκληρη για τα τελεφέρικ. Σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες θα πρέπει να εφαρμόζεται. Ωραία, είναι μια οδηγία ασφαλείας, δηλαδή να μην πέσει το πράγμα και σκοτωθεί ο κόσμος, αλλά ε, ως δημόσια συγκοινωνία δεν αναφέρεται καθόλου το τελεφερίκ. Δεν τους είχε περάσει από το μυαλό για να καταλάβουμε ακριβώς ότι είναι σιδηρόδρομοι ε, είναι ένα είδος τρένου που απλώς κρέμεται από ένα σειρματόσχηνο. Χρειάζονται ευρωπαϊκά προγράμματα, πιλωτικά και μια νέα οδηγία που δεν έχει να κάνει με την ασφάλεια, αλλά να πει ότι είναι ένα κανονικό μέσο μεταφοράς, μπορεί να υπάρχει παντού, όχι μόνο εκεί που έχει χιόνια και ψηλά βουνά, και στο Αμβούργο και στην Ιταλία και όπου αλλού θέλετε φτιάξτε ένα τελεφερίκ. Είναι ένα κανονικό μέσο μεταφοράς της πόλης. για την ελευθερία. Είναι απλή η απάντηση. Όταν είναι οι δρόμοι ευφυείς μπορείτε να κάνετε εσείς κάτι άλλο, δεν χρειάζεται να οδηγείτε. Μπορείτε να φυλάτε το συνοδηγό σας, ας πούμε, ή τη συνοδηγό σας. Έχετε την ελευθερία σας. Η σημερινή κυκλοφορία είναι άρση ελευθερίας. Χρειαζόμαστε ελευθερία στην κινητικότητα, να είναι λιμένα τα χέρια μας, να μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε. είναι όλα γεμάτα κομπιούτερ τα αυτοκίνητα. Έχετε υδραυλικό ε, τιμόνι σήμερα, έχετε βοήθεια για την ανηφόρα. Αυτό τι είναι, σας αφαιρεί ελευθερία. Μπορείτε να είστε και λίγο απρόσεκτοι, δεν θα τρακάρετε. Και ρωτάτε ποιο είναι το επιχειρηματικό μοντέλο. Το επιχειρηματικό μοντέλο είναι λίγο Big Brother, είναι λίγο Big Data, το έχει καταλάβει αυτό η Apple που είναι μέγας πρωτοπόρος με όλες αυτές τις εφαρμογές. Αλλά ε, όσο δεν το χρησιμοποιούν αυτά τα δημόσια συστήματα, ε, γιατί έχουν μείνει στήλοι άλατος και δεν ε, βάζουν ένα πλαίσιο, δεν αντιδρούν, δεν δημιουργούν ένα τρόπο που να μπορεί να συνδυάζεται και με τις άλλες χώρες, θα έχουμε πάλι ζούγκλα. Ο καθένας θα έχει τις δικές του προδιαγραφές και χαιρετίσματα. Λοιπόν, πώς θα γίνουν όλα αυτά πολιτική μεταφορών τώρα. Εγώ είμαι ένθερμος υποστηρικτής της δημοτικής επικουρικότητας. Οι καλύτερες ιδέες φυτρώνουν από τα κάτω. Σας είπα ότι είναι ένα ε, λιβάδι ε, γεμάτο λουλούδια και η Δανία και η Ιταλία και η Ολλανδία. Ο κήπος είναι ανθυρός. Αλλά ε, δεν μπορεί να παραμένει σε μία πόλη, το, η Delft πριν από 40 χρόνια, η Κοπενχάγη αργότερα. Εφόσον δεν γίνει αυτό εθνική πολιτική και να έρθει η Ευρώπη να πει ότι μου είναι σημαντικό αυτό το πρόγραμμα και πρέπει να γίνει ευρωπαϊκή πολιτική γιατί αφορά θέματα του μέλλοντος ευρωπαϊκά και οι εθνικές κυβερνήσεις αντιλαμβάνονται λάθος την επικουρικότητα. Αφήνουν στη μοίρα τους τις κοινότητες που είναι όλες ε, σε αφέμαξη οικονομική. Αν δεν έχουν τη δυνατότητα να βάλουν διόδια οι πόλεις για να πάρουν λεφτά, γιατί η συμφόρηση και τα ποτηλιαρίσματα είναι πρόβλημα δημοτικό, είναι τοπικό, ε, αλλιώς δεν θα προχωρήσουμε. Και έγινε και μια ερώτηση για νέους και οι ε, πιο ηλικιωμένους. Μας λένε οι κοινωνιολόγοι ότι οι νέοι είναι πιο δυναμικοί, πιο ε, καινοτόμοι, υιοθετούν νέε ιδέε. αλλά την πολιτική δεν την κάνουν οι νέοι, την κάνουν οι γέροι. Αν δεν κουνηθούν οι γέροι, τι να το κάνω αν είναι οι νέοι ε, καινοτόμοι και ε, ανανεωτικοί. Αν τα νομοθετικά, τα οικονομικά συστήματα παραμένουν σε αγκύλωση στην πολιτική. Και τι γίνεται με την οτροπία. Εγώ είμαι απολύτως αισιόδοξο. Κοιτάξτε λίγο τις επικοινωνίες, τηλεπικοινωνίες. Ευρώπη, Αφρική, Ασία, οι πάντες αμέσως ήταν έτοιμοι να καινοτομήσουν όταν βγήκαν τα καλώδια από τα τηλέφωνα. Θυμάστε, το τηλέφωνο ήταν σταθερό, περίμενες τρεις μήνες για να πάρει σύνδεση. Σήμερα πας σε ένα μαγαζί, αγοράζεις το καφορδιστήρι σου και το έχεις ο κόσμος αντιδρά ανάλογα με τη τεχνολογία. Το ψυχολογικό μοντέλο ποιο είναι. Χρειάζεται marketing, μια καλή ιδέα και πρέπει να έχεις και λεφτά να επενδύσεις και στο marketing. Και ε, πάλι είμαστε σε λάθος δρόμο. Υπάρχει marketing για πεζούς, <laughs> για ε, ε, ποδήλατα. Με μόνο εξαιρέσεις υπάρχουν. Και πάλι πιστεύω ότι και εμείς σε ευρωπαϊκό επίπεδο χρειαζόμαστε οθήσεις, κίνητρα που είναι κάτι παραπάνω από συλλογή βελτίωση των πρακτικών που καλέσει και αυτέ, αλλά δεν φτάνει. Χρειάζεται μια ευρωπαϊκή πολιτική για την κινητικότητα. Ευχαριστώ πολύ. Η Σόνια Χέκηλετα. Ευχαριστώ. Συμφωνώ με τον κύριο Μόνχαεμ για τα τρία στοιχεία που θα μπορούσαν να μα φέρουν μεταφορέ, εάν ε, οργανωθούν καλύτερα. Οι υπηρεσίε κινητικότητα θέλουν περισσότερη ευελιξία και περισσότερε επιλογέ για του χρήστε τη μεταφορέ. Κρίμα που δεν είχαμε το χρόνο να περάσουμε στις λεπτομέρειες για ε, τις υπηρεσίες κινητικότητας, αλλά καταρχάς μιλάμε για περισσότερες επιλογές στις υπάρχουσες ε, δυνατότητες μεταφορών, για να καλυφθούν πραγματικές ανάγκες, ανάγκες των ανθρώπων, που τώρα με ένα γιοταχή, μάλλον δεν έχουν ένα γιοταχή, δεν σκέφτονται καν να αγοράσουν, γιατί ζουν σε περιοχές όπου οι δημόσιες συγκοινωνίες είναι κακές και έχουν διαφορετικές πραγματικές ανάγκες από αυτόν που είναι κάτοχος για ταχύ. Εδώ υπάρχει ένα χάσμα όπου πρέπει να έρθουμε να καλύψουμε τις ανάγκες τους με τις υπηρεσίες κινητικότητας. Έχετε δίκιο για τα αυτοκίνητα. Είναι πρακτικός τρόπος ε, ε, μεταφοράς, μετακίνησης. Θα πρέπει να οδηγούμε, εντάξει, αλλά πρέπει πάντοτε να μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει τον πρακτικότερο και αποτελεσματικότερο τρόπο. Δεύτερον, σας έδειξα μια εικόνα της μηνιαίας συνδρομής με 300 ευρώ. Αυτό σας δείχνει πόσο, οργανώνονται οι υπηρεσίες κινητικότητας. Αντί να αγοράζει όμως κανείς αυτές τις υπηρεσίες, για αυτό ή ένα άλλο ποσό χρηματικό, κάποιοι αγοράζουν ένα συγκεκριμένο επίπεδο υπηρεσιών. Δηλαδή τι θα πει αυτό, ότι με ένα ποσό οι πολιτές θα έλαβαν ένα επίπεδο ποιότητας και θα μπορούσαν να βασιστούν σε αυτές τις υπηρεσίες. Εκεί προσπαθούμε να συναγωνιστούμε τις δημόσιες κοινωνίες και την ιδιωτική ε, χρήση, ε, την ιδιωτική κατοχή αυτοκινήτου. Πολλά είναι τα γιοταχή που διαρκώ είναι σταθμένα σε γκαράζ ή δεν μετακινούνται. Οι δημόσιε συγκοινωνίε όμω πρέπει να έχουν ένα υψηλό επίπεδο ποιότητα για να είναι ανταγωνιστικέ. Και για το επιχειρηματικό δυναμικό. 300 ευρώ, ε, ένα παράδειγμα είναι αυτό, είναι κάτι που ο καθένας μας τίνει να το χρησιμοποιεί μηνιαίως ε, για τις ε, Τα περισσότερα τα διαθέτουμε για την ε, κατοχή και ταχύ. Όμως θα μπορούσαν να, σε, να κατευθύνονται σε άλλες υπηρεσίες μετακίνησης. Εκεί θα υπήρχε ένα μεγάλο επιχειρηματικό δυναμικό εμπορικό μάλλον δυναμικό. Όσο για τα συστήματα πληρωμής, οι υπηρεσίες κινητικότητας θα μπορούσε να χρησιμοποιούν ένα ενιαίο πλαίσιο και μια διαπαθή που να αξιοποιείται από το, όλους τους φορείς. Ευχαριστώ. Ολοκληρώνεται εδώ το δεύτερο πάνελ. Σας ευχαριστώ και πάλι για τις παρουσιάσεις και εκείνους που έκαναν τις ερωτήσεις και πάμε τώρα στο τρίτο πάνελ. Σας ευχαριστώ και πάλι. So, dürfte ich dann bitten... Λοιπόν, παρακαλώ. Καθίστε και πάλι για να συνεχίσουμε. Τρίτο πάνελ. Μεταφορές για τους πολίτες, προώθηση ασφάλειας, απασχόλησης και ποιότητας υπηρεσιών μεταφορών. Η Γκρατσιέλα Γιούστ ε, διευθύντρια προγράμματο από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών. Έχετε το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ για την πρόσκληση να σας μιλήσω. Ο διευθυντή μου θα έπρεπε να έρθει να σας μιλήσει, αλλά δυστυχώς τραμπούληξε τον του το πρωί, οπότε δεν μπορεί να είναι μαζί σα σήμερα, αλλά επειδή είναι τελειομανής, ήθελε να σα μιλήσω για το θέμα αυτό από πρώτο χέρι θα ερχόταν να σας μιλήσει για την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τις λογικές ε, επεμβάσεις, αλλά τέλος πάντων πλάκα κάνω ή θα να σας μιλήσω για τους 11 ε, νεκρούς που χάσαμε από τις αεροπορικές μεταφορές πέρσι, ε, που Μα θυμίζει ότι χάσαμε χίλιου ανθρώπου επίση από τι δρομικέ μεταφορέ. Αυτό είναι ένα τρένο εκτροχιασμένο στο Σαντιάγκο το 2013, όπου 32 έχασαν την ε, ζωή του. Ε, το βίντεο το είδαν ένα εκατομμύριο θεατέ στο YouTube και υπάρχουν και άλλε εκδοχέ του ίδιου βίντεο ε, με παρόμοιου αριθμού θεατών. 26.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή του από οδικές συγκρούσει συγκρούσεις αυτοκινήτων. Δηλαδή 500 θάνατοι κάθε εβδομάδα στους δρόμους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμως οι συγκρούσεις αυτές αναφέρονται ως καθημερινό φαινόμενο. Και Μόνο λίγε γραμμέ σε μια τοπική εφημερίδα θα αφιερώνονταν σε, αυτές τις, ε, στα αυτοκινητιστικά δυστυχήματα το να σώζει κανείς ζωές έχει και οικονομικό κέρδος 1,9 εκατομμύρια για μια ζωή που φόβεται Αν σκεφτείτε το 1 εκατομμύριο ζωές που αποφύγαμε από το 2010 στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτό σημαίνει ότι φτάνουμε στα 18 δις ευρώ που εξοικονομήθηκαν μεταξύ του 2011 και του 2013. Έτσι έχουμε ένα στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μειώσουμε τους θανάτους ε, από αυτοκινητιστικά κατά 50% από το 2010 στο 2020. Εκτιμούμε ότι με ένα 7% μείωση ετησίως ε, κατά μέσο όρο θα μπορέσουμε να τα καταφέρουμε. Ε, Δυστυχώ το 2014 τα προσωρινά ε, στοιχεία για την Ευρωπαϊκή Ένωση μας δίνουν μόνο 2% μείωση σε σχέση με το 2013. Πρέπει να κάνουμε περισσότερα. Καλούμε το Ευρωκοινοβούλιο να μας στηρίξει για τις συστάσεις μας. Στη δική σας έκθεση, κύριε Κάμπ, ζητούμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εγκρίνει έναν στόχο ώστε να μειωθεί ο αριθμός και των σοβαρών τραυματισμένων για να έχουμε μια ισχυρότερη στρατηγική με τα απαραίτητα μέτρα. Επίσης η οδηγία για τη διαχείριση της ασφάλειας των υποδομών να μην καλύπτει μόνο τα TNT, τα ευρωπαϊκά δίκτυα, αλλά και τι οδικέ μεταφορέ. Χρειάζονται εδώ εμπειρογνώμονε μελέτη των υψηλών κινδύνων, τα σημεία όπου χάνουν τη ζωή του οι άνθρωποι και ε, προτινόμενε λύσει. Επίση πρέπει να δούμε την αναθεώρηση του Γενικού Κανονισμού για την Ασφάλεια φέτο ω μια μοναδική ευκαιρία. Πολλά μπορούν να γίνουν τα επόμενα 5 με 10 χρόνια για να υπάρχει ε, τεχνολογική ε, παρέμβαση εντό των οχημάτων, όπως τα εξελιγμένα φρένα, τα μέσα ελέγχου τη ταχύτητα. και οι ζώνες ασφαλείας σε όλα τα καθίσματα. Αυτό θα ε, εξασφαλίσει ε, την διάσωση ζωών και στα αστικά κέντρα αλλά και εκτός. Και βεβαίω να περιορίσουμε και την εκπομπή διοξιδίου του άνθρακα. Το 95% όλων των ε, θανάτων από τι μεταφορέ συμβαίνουν στο δικό δίκτυο. Αλλά δεν υπάρχει ίδρυμα ε, ή Ινστιτούτο για την Οδική Ασφάλεια. Καλούμε το Ευρωκοινοβούλιο να απευθύνει έκκληση για την ε, επέκταση των αρμοδιοτήτων του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για του Ιδροδρόμου, ώστε να δημιουργηθεί και ένα ανάλογο οργανισμό για τι οδικέ μεταφορέ. Ευχαριστώ. Κρίστοφερ Έρβιν, αντιπρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Επιβατών. Ευχαριστώ. Η Ομοσπονδία μας είναι μια εθελοντική ομοσπονδία που αποτελείται από 30 οργανώσεις σε 20 χώρες. Υπάρχει κάτι το οποίο μας ενώνει, όπως και με σας, και αυτό είναι ότι όταν κοιτάμε τις προτάσεις, αυτό που σκεφτόμαστε είναι σε τι χρησιμεύουν για τον επιβάτη. Αυτό είναι η αρχή και το τέλος κάθε αξιολόγησης που κάνουμε. Και το λέω αυτό με θετικό πνεύμα. Το λέω στην Επιτροπή σας γιατί πιστεύω ότι με ομοφωνία πρέπει να αποφασίζετε ανάλογα με τα ωφέλη που οποιαδήποτε πρωτοβουλία πολιτικής μεταφορών προσφέρει στο χρήστη. Τα τελευταία 15 χρόνια έγιναν διάφορες πρωτοβουλίες και είδαμε μερικές που είχαν τεράστια αποτελέσματα, χαμηλότερες τιμές, ευελιξία και είδαμε φοβερά πράγματα και ωραία να συμβαίνουν. Και όχι μόνο όσον αφορά τα δικαιώματα των επιβατών, και αυτό είναι σημαντικό βέβαια, γιατί είναι απτή απόδειξη της αναγνώρισης των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων ότι οι επιβάτες αποτελούν τον πιο αδύναμο κρίκο της αλυσίδας αυτής μεταφορών. Ο κλάδος προσφέρει πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Αυτοί λοιπόν που χρησιμοποιούν τις μεταφορές, οι χρήστες, πρέπει να μπορούν να υποφεληθούν από αυτά. Παρ' όλα αυτά, εξακολουθούμε να έχουμε τεράστιες προκλήσεις μπροστά μας σε σχέση με τους στόχους της Λευκής Βίβλου του 2011. Για παράδειγμα, μείωση των εκπομπών διεξουδίου του άνθρακα κατά 60% μέχρι το 2050. Αυτή είναι μεγάλη πρόκληση και δύσκολη. Είναι οι στόχοι δύσκολοι που πρέπει να πετύχουν διαφορετικοί παράγοντες με διαφορετικές καταστάσεις. Οι επιβάτες, το πιο χαρακτηριστικό αυτή την εποχή είναι ότι αλλάζουν ε, τρόπο μεταφοράς, μέσο μεταφοράς. Η κίτρινη γραμμή είναι οι συνδρομικές μεταφορές, πηγαίνοντας προς το 2060. Και εδώ είναι το μερίδιο των οδικών μεταφορών, Βάση της Λευκής Βίβλου. Είναι τρομερό. Και είναι τρομερό γιατί μιλάμε για μια πολύ μεγάλη αύξηση του μεριδίου της αγοράς που ανήκει στις ευρωμικές μεταφορές πια, τουλάχιστον σύμφωνα με αυτή την εκτίμηση. Αυτό θα γίνει, θα το κάνει η οικονομία από μόνη της. Ή είναι το ότι οι πολίτες αισθάνονται ότι δεν έχουν άλλη επιλογή παρά μόνο αυτή. Οπότε για να αποφύγουν τις οδικές μεταφορές θα πάνε στα τρένα όσο κακά κι αν είναι αυτά γιατί δεν έχουν άλλη λύση ή μήπως θα πρόκειται για επιλογή ή μήπως θα φροντίσουμε να έχουμε καλές μεταφορές σε όλα τα είδη μεταφορών, όλα τα μέσα να έχουν ικανοποιητικά αποτελέσματα για να έχει την ελεύθερη επιλογή ο πολίτης και ο χρήστης. Ο κόσμος αντιλαμβάνεται όλο και περισσότερο ότι αποκτά όλο και μεγαλύτερη σημασία για οδική ασφάλεια. και ότι επηρεάζει πάρα πολύ κόσμο. 400.000 θάνατοι, λέει η υπηρεσία η αρμόδια, και πάρα πολλοί τραυματισμοί. Είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας αυτός που πρέπει να λάβουμε υπόψη μας. Η συμφόρηση πόσο μας κοστίζει. Δεν έχουμε καταφέρει να υπολογίσουμε τις οικονομικές επιπτώσεις των κυκλοφοριακών συμφορήσεων. Μόνο από αυτά τα δύο που ανέφερα θα έπρεπε κανείς να ξαναδεί τη Λευκή Βίβλιο και να δει τι θα κάνουμε από εδώ και πέρα. Αυτή είναι μια ωραία φράση. Πώς θα πετύχουμε υψηλούς στόχους, πώς ε, θα φτάσουμε στο φεγγάρι. Ο καθένας προσπαθεί να πετύχει τέτοιους φιλόδοξους στόχους διαφορετικά. Υπάρχει ένας φαύλος κύκλος. Βελτιώνεται η ποιότητα, ικανοποιείται ο χρήστης, αλλάζει μέσω μεταφοράς, έχει την πολιτική στήριξη, συνεπώς βρίσκεται χρηματοδότηση και άρα ξαναπάμε στην ποιότητα. Εδώ έχω ετοιμάσει αυτό το χαρτί, έχει πολλές λεπτομέρειες και συγγνώμη αν δεν καταφέρετε να τα διαβάσετε στην οθόνη. Τι λέω εδώ. Λέω μερικά πράγματα με ευθύτητα. Ποια είναι αυτά που νοιάζουν, που έχουν νόημα για τους χρήστες. Η αποτελεσματικότητα, η αξιοπιστία, η προσβασιμότητα, ε, το κόστος. Πώς θα συνδυάζουμε όλα αυτά. Όλα αυτά απαιτούν αλλαγή νοοτροπίας. Να αλλάξουμε τον τρόπο που σκεφτόμαστε για τις μαζικές μεταφορές και να λάβουμε υπόψη μας την βιωσιμότητα να αλλάξουν οι σχέσεις. Το θέμα είναι προσφορά και ζήτηση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Τόμας Αβαντζάτα τώρα, Διευθυντής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων του ε, Διεθνούς Ένωσης Δημοσίων Συγκοινωνίων. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση να σας απευθυνθώ σήμερα και να παρουσιάσω τι δικέ μας συστάσεις για την ενδιάμεση αναθεώρηση της Λευκή Βίβλου του 2011. Η EAPT είναι μια διεθνή οργάνωση ε, ενδιαφερομένων και φορέων από όλο τον κόσμο με μεγάλη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η συμβολή τώρα των δημόσιων συγκοινωνιών στους στόχους της, της Λευκής Βίβλου. Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, μεταφέρει 100 68 δις βιβάτες ε, το χρόνο και είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να μειωθούν οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, η εκτεταμένη χρήση Ο τομέας μας ε, κινείται και προς την απαλλαγή από τον άνθρακα με την ηλεκτροκίνηση ήδη από σήμερα και με, εναλλακτικά, ε, με εναλλακτικές πηγές καυσίμων. Πέραν της απαλλαγή από τον άνθρακα, η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να βελτιώσει και την, το, την ασφάλεια την ασφάλεια των δρόμων και όπως φαίνεται, ότι, ε, όπως φαίνεται οι δημόσιες συγκοινωνίες είναι οι ασφαλέστερες. Επίσης οι δημόσιες συγκοινωνίες συμβάλλουν στην καλύτερη ποιότητα των αστικών κέντρων και την φυσική κατάσταση των πολιτών και την υγεία τους. Επίσης από τη συμφόρηση και το αυξανόμενο κόστος που έχει να κάνει με την ε, συμφόρηση. Ε, σημαντικό ε, για τις δημόσιες συγκοινωνίες είναι να πούμε ότι προάγουν την οικονομική ανάπτυξη στις πόλεις, τις καλές σχέσεις μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών και μειώνει και το κόστος ε, μετακίνησης για πολλές ευρωπαϊκές εταιρείες η κάλυψη του κόστους των συγκοινωνιών είναι το σημαντικότερο παράγοντα για να σκεφτούν που θα εντοπίσουν την προσφορά των υπηρεσιών τους. Η πρόσβαση στι ε, δημόσιε συγκοινωνίες κάνει τις πόλεις ε, πιο αλκιστικές και αυξάνει και την αξία των, ε, των ε, ακινήτων. Στις Ηνωμένες Πολιτείες πρόσφατες μελέτης από τις τιμές των ακινήτων κοντά σε κέντρα δημόσιων συγκοινωνιών δείχνουν ότι είναι ανατεκτικότερε τιμές αυτές τις τιμές κρίσης. Βεβαίως οι δημόσιες συγκοινωνίε ε, προσελκύουν και τουρίστες τα αστικά κέντρα. Οι δημόσιες συγκοινωνίε και οι φορείς του είναι από τους μεγαλύτερου εργοδότες της πόλης και ε, απασχολούν πολίτες με, με, με ένα μεγάλο φάσμα δεξιοτήτων. Οι θέσεις αυτέ εργασίας δεν φεύγουν στο εξωτερικό. Τα μέλη μας επίσης ε, επιτελούν συνεχή πρόοδο για τη βελτίωση της ποιότητας και της ε, πρόσβασης των ανθρώπων και η πρόοδος που επιτελείται σε αυτό το τομέα αφαιρεί όλους τους επιβάτες με ή χωρίς την περισσότερη κινητικότητα. Για να πετύχουμε τις γοργά εξελισσόμενες προσδοκίες των επιδοτών προχωρούμε και προς την πόρτα σε πόρτα κινητικότητα καθώς και την ευφύ ε, την ε, επιβολή ε, εισιτηριών έχουμε αυτή την ευφυή συμμαχία για τα εισιτήρια με την από κάτω προς τα πάνω προσέγγιση τη διαλογικότητα των συστημάτων της Ευρώπης κάτι που ήδη γίνεται σήμερα και επίσης πιστεύουμε ότι η συνεργασία με άλλους παρόχους κινητικότητας είναι επιθυμητή, είναι καθοριστική σημασία και οι δημόσιες κοινωνίες μπορούν να γίνουν ραχοκοκαλιά τη Αστική κινητικότητα. Αυτό θα πρέπει να λειτουργήσει ω παράγοντα συντονισμού ενός ολοκληρωμένου συστήματος. Για τους λόγους που έχουν αναφερθεί ως τώρα είναι σαφές ότι η βιώσιμη ε, κινητικότητα της πόλης, που είναι φιλική και προς τους πολίτες πρέπει να βασίζεται στις δημόσιες κοινωνίες κατά τη γνώμη μας. Η Λευκή Βιβλία του 2011 βαδίζει στη σωστή κατεύθυνση προς το στόχο αυτό. Ε, όπως ξέρετε οι ευφυείς πόλεις υιοθετούν το απόφυγε μετακινήσου βελτίωσε. Ε, αυτό είναι το σύνθημα και αυτές οι βελτιώσεις πρέπει να συνεχιστούν η μετατόπιση του τρόπου ε, μετακίνησης είναι ένας στόχος που πρέπει να επιδιωχθεί περαιτέρω. Ε, είναι απολύτως αναγκαίος για να πετύχουμε τη βιώσιμη και αποτελεσματική αστική κινητικότητα. Αν κοιτάξουμε τα αριθμητικά στοιχεία, ε, το βλέπετε στη διαφάνεια τώρα, η μετακίνηση, η μετατόπιση των τρόπων μεταφοράς δεν έχει επιτευχθεί πλήρως ακόμη. Βλέπετε με το διάγραμμα ότι οι τοπικές διαδρομές στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυξάνονται, αλλά αναλόγως μόνο με την αύξηση του πληθυσμού οι δημόσιες συγκοινωνίε, τα αστικά κέντρα και οι καθημερινές διαδρομές ε, σε αυτά μειώνονται στο γαλάζιο τμήμα του διαγράμματος. Εάν συνεχίσουμε με το σημερινό σύστημα, και αυτή είναι η δεύτερη στήλη, δεν θα αυξηθούν πολύ οι καθημερινές διαδρομές. Όμως ο συνολικός αριθμός διαδρομών θα αυξηθεί μαζί με την ιδιωτική ε, ε, ηλεκτροκίνηση. Εάν όμως διπλασιάσουμε το μερίδιο των δημόσιων συγκοινωνιών, περισσότερες δυνατότητες κινητικότητας θα ε, αναδυθούν. Όπως βλέπετε, αυτό θα έχει και δραστικές επιπτώσεις στην αναχέτηση των ε, εκπομπών ε, διοξιδίου του άνθρακα. Οπότε συστήνουμε τους ε, φιλόδοξους στόχους της Λευκής Βίβλου να τους διατηρήσουμε, έχοντας κατά νου ότι οι στόχοι αυτοί ενθαρρύνουν τις πόλεις να εγκρίνουν σε τοπικό επίπεδο τις κατάλληλες πολιτικές. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να λάβει ενισχυμένα μέτρα για να επιδιώξει του στόχου της Λευκής Βίβλου. Ε, μια αποτελεσματική πολιτική μεταφορών εξαρτάται από πολλέ αποφάσεις όπως τον την αστική πολεοδομία, την ε, σωστή καταγραφή των ε, μέσων μεταφοράς ε, και ούτω καθεξής. Θα πρέπει λοιπόν σε τοπικό επίπεδο να εγκρίνει τις κατάλληλες πολιτικές η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ε, τρίτη μα σύσταση είναι να δοθεί χρηματοδοτική στήριξη για τι δημόσιε συγκοινωνίε στα αστικά κέντρα και τι υποδομέ του, λόγω χάρη μέσω στρατηγικών επενδύσεων που θα πρέπει να συμπεριλαμβάνουν ε, το Connecting Europe Facility και να προέρχονται και από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων. Η ασφάλεια τη μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση είναι η βάση για την επιτυχημένη εξέλιξη των ε, δημόσιων συγκοινωνιών. Είναι πολύ σημαντικά για τη μετατόπιση των μέσων συγκοινωνιών, για τι υπηρεσίε προ του επιβάτε και για τη χρήση τεχνολογιών που που δεν καταναλώνουν άνθρακα. Πρέπει να ενθαρρύνουμε τα κράτη-μέλη να βεβαιωθούν για τη χρηματοδότηση αυτή σε εθνικό επίπεδο. Ε, Παρομοίω, για να βελτιώσουμε τι δημόσιε συγκοινωνίε στα αστικά κέντρα, χρειάζεται περισσότερη έρευνα και καινοτομία. Όπω ε, τέτοιε βελτιώσει θα ε, εξυπηρετήσουν και τι φιλοδοξίε μα για την ε, μετατροπή των τρόπων την μετατόπιση των τρόπων μεταφοράς. Με την ανάληψη των, ε, του εξωτερικού κόστους θα μπορούσε η Ευρωπαϊκή Ένωση να πετύχει βιώσιμες και συλλογικές δημόσιες συγκοινωνίες που να έχουν στοχευτεί σωστά. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα η Σαμπίνε Τρίερ, αναπληρώτρια Γενική Γραμματέας ε, της CTF, που είναι η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Εργαζομένων στι Μεταφορέ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Καταρχάς η Ομοσπονδία μας εκπροσωπεί πάνω από 3,5 εκατομμύρια εργαζομένους μεταφορές σε όλα τα μέσα μεταφοράς. Τα προβλήματα μας πάντα είναι ότι έχουμε να πούμε πολλά για την πολιτική μεταφορών, για όλα τα μέσα μεταφορών, γιατί κάθε μέτρο πολιτικής επηρεάζει την απασχόληση, τις εργασιακές συνθήκες κτλ και ποτέ δεν έχουμε το χρόνο. Έξι λεπτά, τι να πεις έξι λεπτά μέσα. Δεν προλαβαίνουμε τίποτα. Γι' αυτό θα επικεντρωθώ στο θέμα του κοινωνικού ντάμπινγκ και την ανάγκη μιας πραγματικής κοινωνικής ατζέντα ενός θεματολογίου για τις μεταφορές. Βεβαίως για κάθε μέσο μεταφοράς θα μπορούσα να επεκταθώ σε βάθος, αλλά τώρα πρέπει να παραμείνω σε πολύ γενικά. Δεν θα πρέπει να λησμονούμε ότι χωρίς τους εργαζομένους μας τι μεταφορές δεν νοούνται μεταφορές, τουλάχιστον όχι επί των και όχι τα επόμενα 20 χρόνια θα έλεγα. Η Λευκή Βίβλος για τις μεταφορές λέει στην παράγραφο 37 ότι η διάνοιξη της αγοράς θα πρέπει να συμβαδίζει με ποιοτικέ θέσει απασχόλησης και ε, εργασιακές συνθήκες γιατί το ανθρώπινο δυναμικό και η ανθρώπινη πόρη είναι ουσιαστικό στοιχείο κρίσιμο για οποιασδήποτε μεταφορές ποιότητας. Επίσης λέγει ότι είναι ευρέως γνωστό ότι είναι μεγάλη ανησυχία στο μέλλον η έλλειψη προσόντων και η έλλειψη προσωπικού. Η Ομοσπονδία μας θεώρησε θετικό αυτό το μήνυμα, αλλά η προηγούμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή έμεινε μόνο στα λόγια σχετικά με αυτό και έκτοτε δεν έχουμε δει καμιά σοβαρή δράση που να έχει στόχο να προλαμβάνει και ή να επιλύει τις ανητικές επιπτώσεις της διάνοιξης αγοράς της ποιότητα, στην ποιότητα στις εργατικές συνθήκες ή στην ε, πρόληψη του κοινωνικού ντάμπινγκ. Μπορούμε να σας δώσουμε πλήθος παραδειγμάτων για όλα τα μέσα μεταφορών. έχουν ειδικά χαρακτηριστικά οι μεταφορές τα οποία συστηματικά παραγνωρίζονται. Πρώτα απ' όλα θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι οι μετακινούμενοι εργαζόμενοι είναι ε, μετακινούμενοι εξορισμού. Αυτό δεν έχει καμιά σχέση με την κινητικότητα των εργαζομένων. Μιλάμε για ανθρώπους που εργάζονται στο δρόμο και, και μετακινούνται. Είναι πιο ευάλωτοι και χρειάζονται ειδική προστασία για να μην καταντήσουν θύματα επιχειρησιακών μοντέλων επιχειρηματικών που χρησιμοποιούν κάθε παραθυράκι της εσωτερικής νομοθεσίας με μοναδικό στόχο το να μειωθεί στο ελάχιστο το, το κόστος. Και δεν ανησυχούν μόνο οι εργαζόμενοι, αλλά και οι εταιρείε που πληρώνουν σωστά και δίκαια ε, επηρεάζονται αρνητικά από αυτό το κοινωνικό ντάμπινγκ και τις θέμητες πρακτικές. Και αυτό απειλεί και τις εναπομείνασες ποιοτικέ ποιοτικές θέσεις εργασίας και τις εταιρείες που λειτουργούν σωστά. Δεύτερον, ε, πολλά ε, από τα επαγγέλματα των μεταφορών συνδέονται άμεσα με την ασφάλεια. Γι' αυτό χρειάζεται ένα σταθερό πλαίσιο χωρίς κούραση, χωρίς κόποση και να υπάρχουν ε, άνθρωποι καλά καταρτισμένοι με υψηλή ενθάρρυνση. Και θα πρέπει να είναι ελκυστικά αυτά τα επαγγέλματα. Χωρίς αθέμητες πρακτικές, με μακριές περιόδους μακριά από το σπίτι του καθενός, με μακρές χρόνες οδήγησης. Είναι σύγχρονη κοινωνία και οι νέοι μας, όχι μόνο οι γυναίκες αλλά και οι νέοι άντρες, ε, ενδιαφέρονται πιο πολύ ε, από ε, το συγκυρασμό της ιδιωτικής με την επαγγελματική ζωή. Και είναι δύσκολο να προσελκύσουμε νέους επαγγελματίες η Ομοσπονδία μας και τα μέλη της καθημερινά διαπιστώνουν ότι η εσωτερική αγορά των μεταφορών δημιούργησε κοινωνικά χάσματα και κενά τα οποία είναι αφόρητα πλέον και απαράδεκτα. Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Γιούνκερ και ο Επίτροπος Μπούλτς Μεταφορών έχουν δηλώσει και οι δύο ότι είναι κατά του κοινωνικού ντάμπινγκ. Ωραία. Ας ε, φέρουν λοιπόν αποτελέσματα. Η Ομοσπονδία μας φρονεί ότι η αναθεώρηση ε, λέγω, αυτό που χρειάζεται είναι ε, ε, αναδιατύπωση και όχι απλή αναθεώρηση της οδηγίας για το κοινωνικό ντάμπινγκ, για να καταπολεμηθεί με τρόπο σωστό, με κανόνες που να εξασφαλίζουν ίσους κανόνες παιχνιδιού για όλους τους φορείς και όλες τις μεταφορικές εταιρείες. Η αναδιατύπωση της Λευκής Βίβλου θα πρέπει να αντιμετωπίσει διάφορα ε, πράγματα. Εταιρείε φραγίδες, ε, ευκαιριακές ε, σημαίες σε αεροπλάνα και αλλού. Θα πρέπει να γνωρίζουμε πού εδρεύει η εταιρεία, πού έχουν εγγραφεί σε Μητρώα εργαζόμενοι και πού παρέχεται η υπηρεσία μεταφορών. Και να σπάσει και αυτό το φαινόμενο των ψευδό να μην χρησιμοποιείται ε, ενοικίαση εργαζομένων και υπεργολαβία με μόνο στόχο το κοινωνικό ντάμπινγκ. Χρειάζεται ε, να προστατεύονται οι εργαζόμενοι από αθέμητες πρακτικές σε δημόσιους διαγωνισμούς, σε όλα τα μέσα μεταφορών, σε αεροδρόμια, αυτοκινητοδρόμους κτλ. Ε, σε όλα τα μέσα μεταφοράς, όχι μόνο στις οδικές μεταφορές, θα πρέπει να γίνονται σεβαστοί χρόνοι οδήγηση και εργασίας και ε, ξεκούραση. Το σύστημα του ταχυγράφου θα πρέπει να γενικευθεί, να υπάρχει καλή ε, εκπαίδευση, ε, κατάρτιση και να μην έχουμε dumping και στα προσόντα και στις δεξιότητες. Αν είναι υψηλού επίπεδου εκπαίδευση βελτιώνεται η ασφάλεια. Κοινωνική προστασία ε, των εργαζομένων επίσης επιβάλλεται γιατί ε, οι άνθρωποι αυτοί ζουν αλλού και δουλεύουν αλλού. Θα πρέπει να υπάρχει ευρύτερος ορισμός ε, της προσωρινής έδρας στην απασχόληση ισχυρά μέτρα για δίωξη εταιριών που δεν σέβονται κοινωνικά, το κοινωνικά δικαιώματα, το εργατικό δίκαιο και άλλες υποχρεώσεις βλέπουμε ότι υπάρχει μια τάση να ε, μεταφέρει το πρόβλημα στον ευρωπαϊκό κοινωνικό και κλαδικό διάλογο. Αλλά αυτός ο διάλογος δεν μπορεί να λύσει το πρόβλημα. Χρειάζεται ο νομοθέτης ή οι νομοθέτες για να το λύσουν. Και για να επίσης κάποιες αρχές επιβολής του νόμου αυτή τη στιγμή υπάρξει αυτή η νομοθεσία. Ναι, ο κοινωνικός διάλογος θα πρέπει να συμμετέχει στη διαβούλευση και να γίνεται η φωνή του ακουστή. Και βεβαίως οι επιτροπές κοινωνικού διαλόγου υπάρχουν στους διάφορους κλάδους και είναι πρόθυμες να βοηθήσουν να βρεθεί λύση, αλλά δεν μπορούν να δώσουν από μόνες τους τη λύση. Ολοκληρώνω. Οι πρόσφατες εξελίξεις και τοπικές και ευρωπαϊκές μας ανησυχούν και περισσότερο για το κατά πόσο θα επιβιώσει ο κλάδος των μεταφορών και από οικονομική και κοινωνική άποψη. Για να υπάρχει καλός ανταγωνισμός και θεμητός χρειάζονται ίσοι κανόνες παιχνιδιού. Γι' αυτό η Ομοσπονδία μας φρονεί ότι η περαιτέρω συνέχιση της ε, φιλελεύθεροποίησης, χωρίς να λυθούν τα κοινωνικά προβλήματα, χωρίς καν να ακούγονται, θα μπορούσε ενδεχομένως να οδηγήσει σε νέα οικονομικά, κοινωνικά, ίσως και πολιτικά προβλήματα στο ιστορικό της Ένωσης. Καλούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να σταματήσουν την κοινωνική απορρίθμιση, το ξύλωμα μετά από αυτή την τυφλή εφαρμογή της απελευθέρωσης που ε, ε, πρέπει οπωσδήποτε σοβαρά να λάβει υπόψη στην κοινωνική ατζέντα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ακολουθούν ερωτήσεις ο Βίμ Βαντακάμ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Δεν θα εκπλήξει κανέναν ότι αρχίζει η κόπωση λόγω της ώρας, του προχωρημένου της ώρας. Παρ' όλα αυτά κρατάω καλά. Έχω δύο ερωτήσεις στην κυρία Γιούστ. Μπορείτε να μας πείτε κάτι για τις καλές και τις κακές χώρες. Ξέρω ότι το naming και shaming είναι επικίνδυνο αλλά παρόλα αυτά σε κάποιες χώρες βλέπω να μην τηρείται η ασφάλεια, αλλού να τηρείται. Έπειτα η Ευρώπη τι μπορεί να κάνει παραπάνω με ρυθμίσεις που και εσείς προτείνετε σε εθνικό επίπεδο για την ε, μεσοπρόθεσμη αναθεώρηση της Λευκής Βίβλου μπορείτε να μας πείτε ακριβώς τι θα μπορούσε να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Για τον κύριο Ερβουίν. Και εσείς, αλλά και το ETSC, μιλάτε για διπλασιασμό τα οχήματα, τα αυτοκίνητα όντως είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα. Οπότε σας ρωτώ, κύριε Ρουίν, τι θα μπορούσε να γίνει ώστε να προθεθούν ακόμα περισσότερο οι αστικές μεταφορές. Ήταν πολύ εντυπωσιακό αυτό που μας δείξατε με την κόκκινη γραμμή και την κίτρινη γραμμή. Προς τον κύριο Βανσάτα. Συμφωνήσαμε το 2011 στη Λευκή Βίβλο ότι θα εσωτερικεύσουμε το εξωτερικό κόστος. Πώς όμως. Και προς την κυρία Τρίρ. Αυτά που μας είπατε είναι σαφή. Αλλά είναι λίγο παλιωμοδίτικα. Μιλάτε για αλλαγέ, μιλάτε για την αξία της εργασίας, για την ευελιξία. Ναι, αλλά εσείς Πείτε μου τρία πράγματα που θα θέλετε να κάνουμε, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να κάνει κανόνες, να θεσπίσει κανόνες. Αν όμως η αγορά πάει προς την άλλη κατεύθυνση, παράδειγμα με τον ανταγωνισμό εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης στις αεροπορικές μεταφορές, τι νόημα έχει. Οπότε μπορείτε να κατονομάσετε τρεις προκλήσεις. Αντί να μας λέτε αυτή την ε, ιστορία ότι όλα είναι λάθος. Πείτε μας τρία πράγματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ όλους σας που αναφερθήκατε στην ασφάλεια και στις κοινωνικές προδιαγραφές. Εκπροσωπώ τους σοσιαλιστές. Αυτό που πιστεύω ότι είναι σημαντικό είναι η λευκή βίβλος να έρθει με βελτιώσεις και να έχει πραγματικές επιπτώσεις πάνω στις ζωές των πολιτών. Όλοι αυτοί οι παράγοντες πολύ συχνά εξαρτώνται από την επικουρικότητα, εξαρτώνται από το εθνικό επίπεδο. Πώς μπορούν να εφαρμοστούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η κοινωνική πτυχή είναι ζωτική σημασίας, η ποιότητα ε, της απασχόλησης, η κατάρτιση, η πληρωμές. Όλα αυτά είναι ζωτική σημασία στις μεταφορές βέβαια. Πώς όμως μπορεί να επιτευχθεί η εναρμόνιση. Πώς μπορούμε να συμφιλιώσουμε αυτή την ιδέα με το γεγονός ότι πρόκειται για εθνικές αρμοδιότητες. Η ασφάλεια και η προστασία είναι βέβαια πολύ σημαντικά. Φυσικά και πρέπει να μειωθεί ο αριθμός των ατυχημάτων, των νεκρών. Πώς όμως σε ευρωπαϊκό επίπεδο μπορούμε να το πετύχουμε αυτό. Πώς μπορούμε να πείσουμε τις ευρωπαϊκές χώρες για το ότι είναι θετικά αυτό το οποία κάνουμε εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Κομισιόν από τη δικιά της την πληροφορά. Ευχαριστώ και εγώ. Εξ ονόματος των φιλελευθέρων θέλω να ευχαριστήσω τους ομιλητές μας. Έχω μια ερώτηση ε, για ε, τις αστικές συγκοινωνίες. Βεβαίως χωράει μεγάλη βελτίωση, το είπε και ο προλαλής σας και οι μελέτες σας το δείχνουν, αλλά εμείς τι μπορούμε να κάνουμε το ευρωπαϊκό επίπεδο. Είναι θέμα των κρατών μελών στην επικορικότητα οι δημόσιες συγκοινωνίες οι αστικές. Δεν είναι μόνο τα λεφτά, το ξέρω, αλλά εμείς χρηματοδοτούμε ευρωπαϊκούς ε, διαδρόμους μεταφορών ε, και αυτό είναι μεταξύ κρατών μελών, δεν είναι οι αστικέ συγκοινωνίε που είναι μικρή τοπική κλίμακα. Εκεί τι λέτε, πώ θα προχωρήσουμε, τι πρέπει να κάνουμε εμεί από την Ευρώπη. Κύριε Βανζάτα, εσεί μιλήσατε για αλλαγή μέσου μεταφορά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για μια βιώσιμη και αηφόρο κινητικότητα στι πόλει. Ωραία για τι πόλει. Τι γίνεται με την Ήπεθρο, γιατί δεν υπάρχει αυτό. Θα μπορούσε κανείς να έχει περισσότερα συστήματα, ε, να μοιράζεται τις μεταφορές. Δεν χρειάζεται να χτίσει ολόκληρο τρένο. Ε, Πολλέ φορέ έχουν αποκατασταθεί κάποιε σιδηροδρομικέ διαδρομέ και συνδέσει χωρί να έχει αποτέλεσμα. Καλά, δεν θα τι ξυλώσουμε, αλλά δεν είναι οπωσδήποτε απαραίτητο αυτό. Τι, τι λέτε για την Ήπεθρο. Και μια ερώτηση προ όλου. Πώ φαντάζεστε ε, την ένταση της κυκλοφοριακής αγωγής. Ε, το ξέρω ότι αυτό είναι ένα θέμα που αφορά την τοπική κυκλοφορία. Υπάρχουν κάποια μοντέλα που ονομάζονται open space, όπου ξυλώνουν μέχρι και πινακίδες από το δρόμο. Ακούσαμε ότι αν γίνουν όλα ψηφιακά δεν θα χρειάζονται πινακίδες, γιατί όλοι ε, θα τα γνωρίζουν με τα κομπιούτερ που έχουν και θα τους τηλεκατευθύνουν, που, που θα παρκάρουν, θα παρκάρουν μόνα τους τα αυτοκίνητα αλλά πεζοί θα υπάρχουν πάντα. Και οι πεζοί πώς θα κανονίζουν την πορεία τους. Υπάρχουν και άνθρωποι με αναπηρίες που κυκλοφορούν στους δρόμους. Τι είναι το open space, πώς το βλέπετε εσείς. Με ευχαριστώ. Η Μαρία Κίλωνεν. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ευχαριστώ και τους ε, ομιλητές για τις εξαιρετικές τους παρουσιάσεις. Ήθελα να θέσω την ερώτηση μου προς την κυρία Τρίερ που εκπροσωπεί τους εργαζομένους στον τομέα των μεταφορών της Ομοσπονδία του. Είπατε ότι υπάρχουν επίγουσες δράσεις που πρέπει να αναλάβουμε για να βάλουμε ένα τέρμα στο κοινωνικό ντάμπινγκ. Ποιες δράσεις εννοούσατε. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Κέλετ. Ευχαριστώ. Είχαμε και σήμερα πολύ ωραίες παρουσιάσεις. Η πρώτη μου ερώτηση αφορά την ασφάλεια στο δικό δίκτυο. Είμαστε και πάλι μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες που πρόσφατα προέλειψαν νόμο να υπάρχει επίγουσα κλίση από το αυτοκίνητο εφόσον συμβεί κάποιο ατύχημα. Δεν υπάρχει ακόμα αυτό παντού στην αυτοκινητοβιομηχανία μας. Ποια είναι η άποψή σα. Διότι αυτό θα μπορούσε να έχει επιπτώσει, όχι μόνο ω προ τον αριθμό των θυμάτων στου δρόμου μα, αλλά και την ανταγωνιστικότητα τη ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία. Η δεύτερη ερώτηση αφορά το εξή. Σήμερα είχα μία συζήτηση με τους συναδέλφους για να βρούμε έτσι τελείως ε, πρόχειρα κάποιες ιδέες για κάποιο άλλο θέμα. Συνειδητοποιώ ότι πρέπει να μιλήσουμε για πολιτικές, αλλά πρέπει και κάποιοι να τις ακολουθούν. Και το θέμα είναι επίσης ποιος χρηματοδοτεί την πολιτική και τι επιθυμεί να πετύχει. Ποια είναι η γνώμη σας λοιπόν σήμερα Μπορεί κανείς να αγοράσει ανοιχτό εισιτήριο από ένα smartphone. Ε, την κάρτα επιβίβασης συγκεκριμένα μπορεί να τη λάβει επίσης στο smartphone. Είναι όμως αδύνατο να αγοράσει εισιτήριο για τις δημόσιες συγκοινωνίες με αυτόν τον τρόπο. Και στις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές πόλεις δεν θα έπρεπε Το πρόγραμμα επενδύσεων του Juncker να βρεθούν τα απαραίτητα ποσά να τον πείσουμε μαζί με την ομάδα του να διατηρήσει ένα μέρος των χρηματών για την εξέλιξη των δημόσιων συγκοινωνιών. Να βρεθεί μια ευρωπαϊκή λύση για, την ε, για το ευθύ συστήριο. Ευχαριστούμε κύριε Κόχ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Έχω μια ερώτηση προς την κυρία Γιώση Μιλήσατε για ε, συστήματα βοήθηση της οδήγησης. Τα δύο-τρία τελευταία χρόνια ε, υπήρξε τεράστια αλλαγή και νέα τα συστήματα και ποιοτικότερα. Εσείς περιμένετε από την πολιτική να ορίσει υποχρεωτική χρήση αυτών ή μόνο ενημερωτικές εκστρατείες και τα υπόλοιπα να τα αφήσει στην αγορά. Ευχαριστώ πολύ. Ja, jetzt habe ich mich auf die Έχω γράψει και τον εαυτό μου τώρα στον κατάλογο των ομιλητών. Ακούστηκε εξάμεινη συνδρομή. Ε, αυτό έχει και ένα διαπαιδαγωγικό χαρακτήρα γιατί οι φοιτητές είχαν συνηθίσει να έχουν ένα πάσο 5-6 χρόνια και μετά το ε, ε, συνεχίζουν μετά το τέλος των σπουδών τους. Για την θετική εμπειρία μπορούν να τη συνεχίσουν. Παίρνουν άλλο ένα πάσο για 6 μήνες. Στις περισσότερες ε, πόλεις που έχουν μεγάλα πανεπιστήμια αυτό συνεχίζεται και οι νέοι δεν χρησιμοποιούν το γιοταχή πια όπως οι μεγαλύτεροι, το ακούσαμε. στη συνέχεια. Λέτε ότι 10% το γιοταχή στην Ευρώπη θα αρκούσαν για να μπορούμε να μετακινούμεθα. Το είπε ε, ο Χάινερ Μονχάιμ. Αυτό σημαίνει 90% λιγότερα αυτοκίνητα και θα ξεσηκωθεί η αυτοκινητοβιομηχανία. Θα πει θα μου κλείσετε το σπίτι. Χάνουμε εκατομμύρια θέσει εργασία στην Ευρώπη. Ισχύει αυτό, αλλά πώ θα αντιδράσουμε. Αυτό είναι. Γιατί αν αλλάξει η συμπεριφορά του κόσμου θα πρέπει να αλλάξει και η βιομηχανία. Γι' αυτό υπάρχει ένα καλό παράδειγμα. Ας αφήσουμε το 90% λιγότερων τραυματιών και νεκρών από τροχέα. Αλλά υπάρχει ένα καλό παράδειγμα, Daimler Benz, πριν από 25 χρόνια λεγόταν Ρόιτερ ο επικεφαλής της Mercedes και είπε δεν είμαστε ε, μόνο ε, αυτοκίνητο βιομηχανία, θα πρέπει να γίνουμε κινητικότητα. Δηλαδή πριν από 25 χρόνια δεν φτιάχναν μόνο τις μεγάλες Mercedes αλλά ε, φτιάχνανε και φορτηγά μέχρι και ποδήλατα σε δηροδρόμους και αυτοκινητοδρόμους. Βέβαια ένα ποδήλατο ε, που είχε γρανάζια και δεν είχε αλυσίδα και κόστιζε 6.000 ευρώ. Όταν έφυγε ο διάδοχος τα πούλησε όλα, ε, έκοψε και τα μπόνους και σήμερα είναι 100% εξαρτημένη η Daimler-Benz από τη Mercedes, το αυτοκίνητο. Ε, εάν τους πούμε ότι δεν μπορείτε να παράγετε μόνο αυτοκίνητα γιατί θα χρεοκοπήσετε, θα αλλάξουν τακτική. Ταυτόχρονα έχουμε παγκοσμίω μια άνθηση σε αυτοκινητοδρόμους, ε, τρένα υψηλής ταχύτητας, ε, ποδήλατα και ηλεκτροκίνητα ποδήλατα. Εάν λοιπόν τώρα καταφέρνω να κάνω αυτή την αλλαγή ή τα εργοστάσια να ξεφύγουν από το αυτοκίνητο και να ε, έχουν μια συνολική αντίληψη για την κινητικότητα θα επενδύσουν αλλού. Γιατί όταν φτιάχνεις ένα σασί καροτσέρις μπορείς να είσαι και να φτιάξεις αυτοκίνητο και φορτηγό και σιδηρόδρομο για να φτιάξεις το σκελετό. Ε, χρειάζεται λοιπόν αλλαγή νοοτροπίας και θα προστατεύσουμε το κλίμα και το περιβάλλον, πρέπει να αλλάξουν και τα εργοστάσια, τακτική και νοοτροπία. Και δεν θα έχουμε τόσο τεράστιο πρόβλημα με τις θέσεις εργασίας που δεν θέλουμε να χαθούν βέβαια, αλλά πώς το βλέπετε, αυτές είναι οι ερωτήσεις μου. Και ερχόμαστε στις απαντήσεις με αυτή τη σειρά την ίδια η Γατσιέλα Γιώστ. Thank you. Ευχαριστώ. Η ερώτηση του κ. Φαντακάμπ με τις καλές καταστατικές χώρες. Καλές χώρες είναι αυτές που έχουν χαμηλό αριθμό ε, θανάτων στο σύνολο του πληθυσμού, Σουηδία, Κατοχώρες, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, και χώρε που έχουν κάνει μεγάλη πρόοδο πρόσφατα, όπω η Ιλλανδία, η Ισπανία, χώρα τη Βαλτική. Μελετήσαμε την πρόοδο αυτή και δεν έχει σχέση μόνο με την κρίση. Κάποιοι κάτι μέλη θετούν σωστά μέτρα. Το βασικό είναι η επιβολή. Η σωστή επιβολή των ορίων ταχύτητα ή ε, των νόμων για την ε, κατανάλωση αλκοόλ ή η απουσία χρήση ζώνης ασφαλείας. Η βάση τη οδική ασφάλεια είναι ο έλεγχο τη ταχύτητα. Εάν μόνο και ένα μέτρο έπρεπε να εγκριθεί, θα ήταν καλύτερα να εφαρμοστούν τα όρια ταχύτητας και οι επιτόπιοι αστυνομικοί έλεγχοι. Δεν χρειάζεται να εξηγήσουμε και πολύ γιατί το κάνουμε αυτό, για να σωθούν ζωέ. Τα αποτελέσματα τη Γαλλία και τη Ισπανία δείχνουν ότι υπάρχει όντω αποτέλεσμα. Τα υπόλοιπα μέτρα στόχουν να βελτιώσουν τι υποδομέ. Εδώ έχουμε και ένα συσχετισμό με τα όσα η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορούν να κάνουν. Το κάθε θεσμικό όργανο το δικό του ρόλο δεν μπορούν να τα κάνουν όλα μόνο του τα κράτη-μέλη, πρέπει να πιεστούν να κάνουν περισσότερα. Ανέφερα στην παρουσίασή μου ότι χρειαζόμαστε παράταση του, διεύνηση μάλλον του συστήματο διαχείριση ασφάλεια των σιδηροδρόμων στα οδικά δίκτυα. Αυτό πρέπει να το εντοπίσουμε στα κράτη-μέλη, να δουν ποια είναι τα μελανά σημεία, οι γκριζόνε ζώνε στου δρόμου του και να κάνουν του απαραίτητου ελέγχου. Όχι μόνο στου αυτοκινητοδρόμου των διευρωπαϊκών δικτύων, χρειάζεται να γίνεται σε όλου του δρόμου αυτό, επαρχιακού και μικρότερου. Και θα πρέπει να δούμε τι γίνεται και με τον αριθμό των σοβαρών τραυματιών. Πολλοί είναι αυτοί που είναι, έχουν τραυματιστεί σοβαρά. Πρέπει να ξέρουμε περισσότερα λοιπόν ε, τι μέτρα πρέπει να εγκριθούν, διότι υπάρχει μια φθήνουσα τάση για τους ε, θανάτους από αυτοκινητιστικά. όμως ο αριθμός των σοβαρών τραυματιών δεν μειώνεται το ίδιο γρήγορα. Επίση, απευθύνουμε έκκληση για Ευρωπαϊκό Οργανισμό. Δεν υπάρχει Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Οδική Ασφάλεια ακόμη. 7% των ε, θανάτων από τις μεταφορές είναι στα αυτοκινητιστικά. Πρέπει λοιπόν ο Οργανισμός για τη Συνδρομική Ασφάλεια να ασχοληθεί και με την οδική ή να δημιουργηθεί ένα εξάρτητος οργανισμός. Και τέλος η Επιτροπή σας, η Επιτροπή Μεταφορών θα πρέπει να πιέσει για την ε, υποχρεωτικό χαρακτήρα των ε, προδιαγραφών ασφάλειας στον νέο κανονισμό που αναθεωρείται φέτος. Αυτό θα γίνει φέτος. Και το ρώτησε και ο κύριος Κοχ. Πολύ πρόοδος έχει γίνει για τις τεχνολογίες για την ασφάλεια των οχημάτων. Η πρόοδος που έχουμε δει κινητοποιείται, κινείται χάρη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά τα περισσότερα συστήματα είναι εθελοντικά. Υπάρχει υπενθύμηση για τις ζώνες ασφαλείας, υπάρχει φρένο ε, έκτακτης ανάγκης, Υπάρχουν ε, δοκιμές crash test για τα αυτοκίνητα παντού, αλλά πρέπει να ωφελείται ο κάθε πολίτης. Η αγορά έχει καταγερματιστεί μεταξύ των δυτικών χώρων, όπου οι κοινοί φορείς προσφέρουν παρόμοιες προδιαγραφές ασφαλείας, και τις ανατολικές χώρες, όπου δεν μπορεί κανείς να αγοράσει καν τα οχήματα με αυτές τις προδιαγραφές ασφαλείας, διότι είναι ιδιαίτερα ακριβά. Αυτές οι τεχνολογίες λοιπόν θα πρέπει να ξέρουμε ότι θα προσφέρουν και θέσει εργασίας στην Ευρώπη και θα επιτρέψουν την καλύτερη παραγωγή με, τη, με, τα, με τις ζώνες ασφαλείας, με τα φρένα έκτατης ανάγκης, με το, τη διάσωση ζωών, πεζών και ποδηλατών πρέπει το ίδιο να γίνει και για, την, για τον ευφύ έλεγχο της ταχύτητας. Δηλαδή αντί έχουμε, πρέπει να έχουμε πολλές τεχνολογικές λύσεις πλέον στα αυτοκίνητα. Ευχαριστώ. Χριστό Thank you very much. Um, Ευχαριστώ. Όπως οι περισσότεροι από μας εδώ, πιστεύω και εγώ ότι οι μεταφορές είναι ζωτικής σημασίας για την οικονομική ανάπτυξη και για την κοινωνική συνοχή. Και αν θέλουμε να είμαστε σοβαροί επίσης για την ζωή του πλανήτη μακροπρόθεσμα. Αν λοιπόν συμφωνείτε με αυτά, για να απαντήσω κύριε Σιγητά στην ερώτησή σας, τι παραπάνω μπορεί να γίνει, θα άρχιζα από το να βάλω στο μυαλό του καθενός ότι οι μεταφορές είναι κάτι σημαντικό δεν μπορεί να αλλάξει η πολιτική μεταφορών αν δεν την παίρνουμε στα σοβαρά. Πώς είναι δυνατόν αν πιστεύουμε, αν θέλουμε οι μεταφορές να οδηγήσουν σε αξιοπρεπείς μεταφορές για το μέλλον. Πρέπει να δουλέψουμε και πολιτικά και να προσφέρουμε χρήματα για να έχουμε τις μεταφορές που θέλουμε. Αρχίζουμε λοιπόν λέγοντας ποια είναι η ζήτηση, τι θέλουν οι καταναλωτές. Θέλουν προσβασιμότητα, το ξέρουμε γιατί το λένε, θέλουν αξιοπιστία, θέλουν να έχουν μια θέση όταν τη χρειάζονται και θέλουν και να μην πληρώνουν υπερβολικά πολλά. Αν αρχίσουμε λοιπόν από αυτό το σημείο, τότε σιγά σιγά προχωράμε στις κοινωνικές πολιτικές και τις πολιτικές πολιτικές που μπορούν να βοηθήσουν να τα προσφέρουμε αυτά. Στο Ηνωμένο Βασίλειο από όπου προέρχομαι εγώ, ιδεολογικά θέλουμε το άνοιγμα της αγοράς, θεωρούμε ότι είναι κατεξοχήν αυτό για να υπάρχει φιλελεύθερη αντιμετώπιση και το κάνουμε σε ένα βαθμό εκτός ε, πόλεων, μέσα όμως στις μεγάλες πόλεις με μέτρα που έχουμε πάρει, ελέγχους, συστήματα εισιτηρίων που είναι ευέλικτα, διαπιστώνουμε ότι μπορούμε να κάνουμε την αλλαγή και να τα προσφέρουμε αυτά. Χρειάζεται όμως πολιτική βούληση, χρειάζεται δέσμευση, να μην είμαστε υποκριτές. Βραχυπρόθεσμα λοιπόν, θα έλεγα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Σταματήστε τους υποκριτές. Μην τους αφήνετε να εμποδίζουν μια πολιτική η οποία μπορεί να φέρει αποτελέσματα. Ευχαριστώ, Ευχαριστώ. Κύριε Σίγητα, τι να κάνουμε για να βελτιώσουμε τις δημόσιες συγκοινωνίες, τι μπορούμε να κάνουμε εδώ για τις αστικές δημόσιες μεταφορές, συγκοινωνίες. Πρέπει να λύσουμε το παράδοξο της αρχής της επικουρικότητας. Η δημόσια συγκοινωνία είναι ένας τομέας δραστηριότητας, ε, εξόχως τοπικός και είναι πολύ σημαντικό κάποιες αποφάσεις, κάποιες προτεραιότητες να ορίζονται σε επίπεδο τοπικό. Αυτό δεν μπορεί να ε, αλλάξει. Όμως σήμερα κατ' ανάγκη υπάρχει στις πόλεις. Το βλέπουμε ξεκάθαρα αυτό. Βλέπουμε ότι τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα διστάζουν. Διστάζουν ιδίως σε ό,τι αφορά την αλλαγή της προσέγγισης για το δημοσιονομικό επίπεδο. Αλλά και το επίπεδο της παρέμβασης που μπορούν να έχουν σε αυτό το τομέα δράσης. Επίγουσα λοιπόν ανάγκη υπάρχει στις πόλεις. Αυτές είναι οι προκλήσεις των κλιματικών αλλαγών και αυτές είναι οι προκλήσεις της ε, βελτίωσης της ποιότητας της διαβίωσης ή της ανταγωνιστικότητας. Εκεί έχουν προσδοκίες οι πολίτες, εκεί έχουν προσδοκίες οι επιβάτες. Στις πόλεις έχουμε συμφόρηση. Και στις πόλεις έχουμε την τόσο μεγάλη σημασία των δημόσιων συγκοινωνιών. Μας πάνε όλα στραβά όταν κάτι δεν πάει καλά στην πρωινή μας διαδρομή. Εδώ λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να διδραματίσει ένα ρόλο με στόχους που καθορίζονται σαφώς στη Λευκή Βίβλο αλλά που θα πρέπει να επιταχύνουμε την επιδίωξή τους. Σήμερα χρειάζεται αυτή η επιτάχυνση. Ε, πρέπει να καταλάβουμε ότι υπάρχει πραγματική ανάγκη στις πόλεις. Και Πρέπει να αναλάβουμε δράσεις σε αυτό το τομέα των αστικών δημόσιων συγκοινωνιών. Και εκεί πρέπει να αξιοποιήσουμε την τεχνογνωσία μας. Να πω ποιες είναι οι προτεραιότητες, οι τρεις που λέγαμε. Έρευνα, δημόσια συγκοινωνία στα αστικά κέντρα, αυτό δεν το ξεχνάμε στα ερευνητικά προγράμματα, που είναι ο φτωχό, για να μην πω ο άπορο συγγενής, στα προγράμματα έρευνας, επενδύσεις, το συζητάμε πολύ το πρόγραμμα Juncker, αλλά ο στόχος του, της βελτίωσης της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας δεν θα επιτευχθεί εάν μείνουμε, αν αφήσουμε εκτός της πόλης. Και στα ε, διευρωπαϊκά δίκτυα υπάρχει το θέμα των αστικών κόμπων. Είναι μια ευκαιρία εδώ να ξεπεράσουμε τα πρώτα εμβριακά στάδια και να περάσουμε στην αξιοποίηση του χρηματοδότησης από το πρόγραμμα Juncker. Και μετά συνοχή. Δεν θα βελτιώσουμε την κατάσταση με μικρές πινελιές από εδώ και από εκεί. Έστω και αν είναι χρωματιστές. Πρέπει να πάρουμε λίγη απόσταση και να δούμε τον πίνακα συνολικά. Η χωροταξία στις πόλεις επίσης είναι σημαντική. Πρέπει να σκεφτούμε το θέμα των ωραρίων, των ε, ετεροχρονισμένων ωραρίων εργασίας. Όλα αυτά πρέπει να μελετηθούν. Όπως και η ανάληψη του εξωτερικού κόστους, όπως είπατε κύριε Σίγητα. Δεν ξέρω ποιοι είναι ακριβώς οι υπεύθυνοι, αλλά σίγουρα για το θέμα αυτό απαιτείται μεγάλη τόλμη. Τόλμη που είναι δύσκολο να τη βρει κανείς όταν ε, είναι κολλημένος με τις τοπικές εκλογές. Εδώ λοιπόν χρειάζεται τόλμη, αλλά είναι μέρος της λύσης. Και μια τελευταία κουβέντα, κυρία Μάισνερ. Η δουλειά των δημόσιων συγκοινωνιών είναι να μεταφέρουν τις μεγάλες μάζες πολιτών, μεν, αλλά και άτομα, πρόσωπα, όπως το τονίσατε. Υπάρχει πραγματικά θέμα εδώ με το τι θα γίνει με τι ε, μεταφορέ ε, στην Ήπεθρο. Εδώ είναι θέμα κοινωνική συνοχή. Δεν θα είναι οι ίδιε απαντήσει, αλλά είναι κάτι που οπωσδήποτε πρέπει να σκεφτούμε. Ευχαριστώ που μου δώσατε ένα λεπτό παραπάνω. Ευχαριστώ. Η Σαμπίνε Τρία, ε, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Φαντεκάμπ, είμαι πιο εξοικειωμένη με τους σιδηροδρόμους και τις πλωτές μεταφορές και ξέρω περισσότερο τους εργαζόμενους που απασχολούνται σε αυτούς τους δύο τομείς. Το θέμα του διεθνούς ανταγωνισμού δεν έχει τόσο να κάνει με αυτό. Για τις αεροπορικές μεταφορές νομίζω ότι δεν πρέπει να κοιτάξουμε τις ε, θαλάσσιες μεταφορές. Ξέρουμε τι γίνεται με τις μέσες ευκαιρίες εδώ και τόσα χρόνια. Αν χρησιμοποιήσουμε αυτό το επιχείρημα, τότε κάποια στιγμή θα έρθουν και αεροπορικές μεταφορές στην ίδια κατάσταση. Δεν θα υπάρχουν δηλαδή τελικά Ευρωπαίοι εργαζόμενοι. Αυτό πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας και να προσπαθούμε να ακολουθήσουμε άλλα παραδείγματα καλύτερα. Τα τρία σημεία που μου ζητήσατε, ε, φυσικά είναι πολύ δύσκολο για μένα να επιλέξω ένα από τα μεγάλα προβλήματα πάντως στις μεταφορές για τους εργαζόμενους είναι η διαφάνεια των συμβάσεων, τι γίνεται με την κοινωνική ασφάλιση που πληρώνεται αυτή και να αποφεύγουμε καταστάσεις όπου έχετε εταιρείε που έχουν απλώς μια θηρίδα, δεν υπάρχουν δηλαδή καλά-καλά, που οι εργαζόμενοι δεν γνωρίζουν τι γίνεται με την κοινωνική τους ασφάλιση, που μπορούν να απευθυνθούν αν έχουν κάποια διαμαρτυρία, τι γίνεται με τα κοινωνικά του δικαιώματα κλπ. κλπ. Σας είπα, είναι το πρόβλημα των εταιριών θηρίδων, των αυτοαπασχολούμενων, αλλά και το θέμα της νομοθεσίας για το συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης. Ένα άλλο σημείο είναι βέβαια η ασφάλεια. Και αυτό έχει να κάνει με τις συνθήκες εργασίας και τον χρόνο ανάπαυσης. Είναι μεγάλη προτεραιότητα. Και όπως είπα και πριν, δεν πρόκειται μόνο για τις οδικές μεταφορές, πρόκειται για όλες τις μεταφορές. Πρέπει να κάνουμε πολύ μεγάλες προσπάθειες για να ενισχύσουμε την υπάρχουσα νομοθεσία και να χρησιμοποιήσουμε τα μέσα εκεί που δεν υπάρχουν. Και το τρίτο που θα έλεγα, που έχει να κάνει πιο πολύ με το δικό μου τομέα, είναι υποχρεωτική προστασία των εργαζομένων κάθε φορά που γίνονται διαγωνισμοί. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα ακολουθούν τα σχόλια του εισηγητού μας. Ε, του ΟΚΕ, όχι το δικό μας, είναι ο κύριος Στέφαν Μπακ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ζητήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να υποβάλει τις απόψεις της όσον αφορά την εφαρμογή της Λευκής Βίβλους για τη... Βίβλου του 2011 για τις μεταφορές, για να βοηθήσει το Κοινοβούλιο να ετοιμάσει τη δικιά του την έκθεση. Σας ευχαριστούμε πολύ λοιπόν για την ευκαιρία που μας δίνατε να συνεργαστούμε. Η γνωμοδότησή μας δεν είναι έτοιμη ακόμα, σκοπεύουμε να την υιοθετήσουμε τον Απρίλιο στην Ολομελιά μας. Αυτό που μπορώ σήμερα να σας παρουσιάσω είναι μια περίληψη του σχεδίου γνωμοδότησης μετά από τις δύο συναντήσεις που είχαμε στην ομάδα εργασίας που ασχολείται με αυτό. Όπως και εσείς, έτσι και εμείς, είχαμε μια κρόαση στις 6 Μαρτίου για να ακούσουμε τους διάφορους φορείς, τη γνώμη τους για την εφαρμογή και για το τι θα γίνει στο μέλλον όσον αφορά τη λευκή αυτή βίβλο. Σημειώσαμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ένα μεγάλο βαθμό έχει τηρήσει τις υποσχέσεις της ε, από τη Λευκή Βίβλου, γιατί ε, τα μισά τουλάχιστον θέματα έχουν προχωρήσει στην νομοθετική διαδικασία. Δεν έχει τελειώσει όμως η νομοθεσία, δυστυχώς, γιατί οι νομοθέτες σε πολλές περιπτώσεις δεν έχουν δεχτεί τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή τις έχουν αλλάξει αυτές εντελώς. Και μερικές φορές οι χώρες μέλη έχουν καθυστερήσει ή δεν έχουν προχωρήσει σε εφαρμογή. Αυτό ισχύει με το άνοιγμα της αγοράς σιδηροδρόμων, με την ολοκλήρωση των ευρωπαϊκών εθέρων, με το πακέτο αεροδρομίων, με την εσωτερική του εξωτερικού κόστους και με άλλα ζωτικά θέματα της Λευκής Βίβλου. Βέβαια, δεν πρόκειται για μια τεχνική διαδικασία και μόνο, πρόκειται για μια πολιτική διαδικασία η οποία παράγει κάτι το οποίο να είναι πολιτικά αποδεκτό. Όμως το χάσμα που υπάρχει ανάμεσα στους φιλόδοξους στόχους της Λευκής ε, Βίβλου είναι κάτι πολύ μεγάλο. Γι' αυτό ακριβώς εμείς πιστεύουμε ότι η πρόθεση της νέας Επιτροπής που είπε ότι ε, θέλει πρώτα να είναι σαφής η πολιτική κατάσταση πριν προχωρήσει σε προτάσεις που είπε ότι προτιμάει να ε, κάνει λίγες προτάσεις αλλά που να έχουν περισσότερες πιθανότητες επιτυχίες και ότι θα φροντίσει για τον έλεγχό του είναι κάτι θετικό. Ελπίζουμε να μας δείξει ότι όντως θα τα όλα αυτά. Εν πάση περιπτώσει, τα περισσότερα ζητήματα τα οποία αναφέρονται στη Λευκή Βίβλο εξακολουθούν να βρίσκονται στην εμερήσια διάταξη και θα λέγαμε ότι σχεδόν κανένα δεν έχει ολοκληρωθεί, ή δεν έχει φτάσει στο σημείο της εφαρμογής. Η γνωμοδότησή μα υπογραμμίζει λίγα μόνο ζητήματα τα οποία βλέπουμε ως στοιχεία κλειδί. Πρώτον, η χρηματοδότηση και η σχέση ανάμεσα στο συνδέοντας την Ευρώπη και το επενδυτικό πακέτο Juncker. Όντως πιστεύουμε ότι είναι πολύ σημαντικό να έχουμε επενδύσεις για τα ευρωπαϊκά δίκτυα. Το επενδυτικό πακέτο θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει περισσότερους πόρους από το συνδέοντας την Ευρώπη για θέματα τα οποία εμπορικά δεν είναι τόσο ενδιαφέροντα. Αλλά τι θα γίνει στις πιο αεροκατοικημένες περιοχές. Εμείς θέλουμε και το επενδυτικό πακέτο να βοηθήσει με προγράμματα τα οποία να είναι σημαντικά αλλά να μην μπορούν να χρηματοδοτηθούν από το συνδέοντα στην Ευρώπη. Τα ποσά τα οποία λοιπόν παίρνουμε από το συνδέοντα στην Ευρώπη για την εγγύηση στο επενδυτικό πακέτο είναι κάτι που δεν μας αρέσει. Πρέπει να ξέρουμε ότι τα χρήματα αυτά που είναι περίπου 2,7 δισεκατομμύρια θα χρησιμοποιηθούν με τέτοιο τρόπο που να είναι συμβατός με τις προτεραιότητες των διευρωπαϊκών δικτύων. Αλλιώς κινδυνεύουμε να δούμε ότι οι πόροι αυτοί θα χαθούν από εμπορικά, εμπορικού ενδιαφέροντος προγράμματα περισσότερο και όχι τόσο για τους στόχους της ε, ε, σύνδεσης στην Ευρώπη όπως θέλουμε. Δεύτερον, η χρηματοδότηση των υποδομών και η χρέωσή τους. Υπάρχουν τομείς που δεν θα λειτουργήσει ποτέ αυτό και όπου η χρέωση θα είναι απαγορευτική ή θα περιορίσει πάρα πολύ την κινητικότητα των πολιτών ή θα έχει καταστροφικές συνέπειες στον ανταγωνισμό των επιχειρήσεων. Αυτό ισχύει σε απομακρυσμένες περιοχές σε αεροκατοικημένες περιοχές και για τους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι οικονομικά δεν ε, είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Πρέπει να αποφύγουμε τέτοιες αρνητικές επιπτώσεις τη χρέωσης. Το ίδιο ισχύει και για την εσωτερική του εξωτερικού κόστου. Εμείς πιστεύουμε ότι δεν έχει νόημα σε περιοχές όπου δεν υπάρχει επιλογή, όπου μόνο δικές μεταφορές προσφέρονται και όπου δεν υπάρχει συμφόρηση. Σε τέτοιες περιπτώσεις το οριπένον πληρώνει θα αυξήσει το κόστος της κινητικότητας. Εμείς πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό να γίνει διάκριση ανάμεσα στο οριπένον πληρώνει και ο χρήστης πληρώνει. Γιατί ο στόχος της εσωτερικής του εξωτερικού κόστους είναι να χρεώνεται η συμπεριφορά. Το να χρηματοδοτήσεις δεν πρέπει να είναι σε βάρος των υποδομών. Επίσης τώρα η αλλαγή του είδους του μέσου μεταφοράς είναι ένας στόχος που αναφέρεται του στόχου του 2011 αλλά πρέπει να είναι πιο ευέλικτος. Γιατί πρέπει να γίνεται διάκριση ανάμεσα στο κέντρο και την περιφέρεια. Όλες οι μορφές μεταφορών πρέπει να είναι πιο αποτελεσματικές και βιώσιμες, η κάθε μία χωριστά και όλες μαζί. Αυτό θα ήταν μια καλύτερη επιλογή για το μέλλον. Πιστεύουμε επίσης ότι το άνοιγμα της αγοράς είναι κάτι σημαντικό για όλους τους τομείς υπέρ τη βιωσιμότητα των μεταφορών. Συγχρόνως όμως πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό οι κανόνες που ισχύουν να είναι σαφείς, να είναι εύκολο να τηρηθούν. Δυστυχώ δεν ισχύει αυτό πάντα σήμερα. Πρέπει να χρησιμοποιούμε καλά το πρόγραμμα REFIT και την πρωτοβουλία για την καλύτερη ρύθμιση. Χρειαζόμαστε μια ανοιχτή αγορά με σαφείς κανόνες. Από κάτι τέτοιο μπορούν να υποφεληθούν όλοι οι επιβάτες και να έχουν καλές μεταφορές. Το κοινωνικό ντάμπικ τώρα είναι για μας ένα σοβαρό πρόβλημα. Είναι κάτι που πρέπει να αντιμετωπιστεί. Δεν χρειάζεται όμως να το συνδέσουμε αυτό με το άνοιγμα της αγοράς. Υπάρχουν κανόνες, ε, μάλλον τρόποι, ρυθμίσεις που μπορούν να βοηθήσουν να αντιμετωπίσουμε τις αποκλήσεις που υπάρχουν ε, στους μισθούς, στους φόρους, στα επίπεδα κοινωνικής προστασίας κλπ. Πρέπει να φροντίσουμε να αντιμετωπίσουμε για παράδειγμα την αδήλωτη εργασία. Χρειάζονται επιπλέον μέτρα για καλή επικοινωνία μεταξύ των αρχών των διαφόρων χωρών μελών. Αλλά να αποφύγουμε τη δημιουργία θεραπείων οι οποίες να χειροτερεύουν το πρόβλημα. Οι λύσεις πρέπει να είναι αναλογικές και δεν πρέπει να εμποδίζουν τη δράση των περισσότερων παραγόντων της αγοράς οι οποίοι συμμορφώνονται στους κανόνες. Πιστεύουμε ότι οι αστικές συγκοινωνίες είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα για το μέλλον και για τους επιβάτες και για τα εμπορεύματα. Πιστεύουμε λοιπόν ότι θα έπρεπε να επεκταθεί η νομοθετική αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στις πόλεις, στους δήμους, για να μπορέσει να υπάρξει αναρμόνιση όσον αφορά τα συστήματα χρέωσης και τις διάφορες ρυθμίσεις. Κάτι θετικό και για το περιβάλλον και για τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Οι τεχνολογικές καινοτομίε μεταξύ άλλων αλλακτικά καύσιμα, άλλα συστήματα κινητήρων, είναι σημαντικές λύσεις για βιώσιμες μεταφορές στο μέλλον. Οι περισσότερες μεταφορές είναι κάτι που πρέπει βέβαια να μην ξεχνάμε και γι' αυτό, αυτό πρέπει να αναφέρεται και στη Λευκή Βίβλο σαφώς. Στα πλαίσια αυτά λοιπόν θέλουμε να επικεντρωθούμε και σε νέα επιχειρηματικά μοντέλα όπως είναι το Uber. Πιστεύουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να κοιτάξει και τις κοινωνικές πτυχές, τις ηθίκες εργασίας των εργαζομένων, την κατάσταση των επιβατών ως καταναλωτές που είναι και το καταμερισμό των ευθυνών στην περίπτωση που υπάρξουν ματυχήματα ε, ή άλλα συμβάντα. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε που μας δώσατε την ευκαιρία να σας παρουσιάσουμε τις θέσεις μας. Ευχαριστούμε. Έχουμε δύο μιλητές ακόμα. Κανονικά ο χρόνος έχει τελειώσει. Θα ήθελα να παρακαλέσω τους διερμηνείς να ακούσουμε δύο μιλητές ακόμα γίνεται και παρακαλώ να είστε σύντομοι. Πέντε λεπτά όπου συμφωνήσαμε έκαστος η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ρολφ Äh, Ευχαριστώ. Εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα ήθελα να πω πόσο χαιρετίζουμε και καλωσορίζουμε ε, την πρωτοβουλία του Κοινοβουλίου για κατάρτιση έκθεσης ε, πρωτοβουλίας που θα μας βοηθήσει πάρα πολύ στην καταγραφή της ε, κατάστασης για τη Λευκή Βίβλο όπως και η ακρόαση σήμερα πολύ χρήσιμη απεδειχθεί από την ποιότητα των παρεμβάσεων και είναι και πάρα πολύ επίκαιρη. Έχουμε αρχίσει ήδη. Ε, οι περισσότεροι από εσά, αν όχι όλοι, θα έχετε δει. Αν όχι, σα λέω ότι έχει αρχίσει δημόσια διαβούλευση στις 10 Μαρτίου για συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων. Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και για λόγους χρονικούς αλλά και για άλλους, γιατί θα επανέλθουμε εν ευθέτω χρόνο με τις ουσιαστικέ προτάσεις, δεν θα μιλήσω τόσο πολύ για την ουσία, δύο λόγια μόνο για τη διαδικασία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει αποφασίσει ακόμα το νομικό καθεστώς του τελικού προϊόντος. Είναι θεώρηση του 2011 της Λευκής Βίβλου είναι μια καταγραφή της κατάστασης, μια φωτογράφηση. Τι έχει ε, υλοποιηθεί, με ποιο τρόπο, να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε για ποιο λόγο ενδεχομένως να μην είναι ικανοποιητική υλοποίηση. Βεβαίως, ακούσαμε πολλά από τη σημερινή ακρόαση. Το 2015 ο κόσμος, ακόμα και αν έχουν περάσει μόλις τέσσερα χρόνια, δεν είναι καθόλου ο ίδιος με το 2011 αρκεί να φέρουμε τις, την οικονομική κρίση, τις τιμές του πετρελαίου και την εξέλιξή τους, αλλά και ιδιαίτερα στις μεταφορές, νέα επιχειρηματικά μοντέλα, νέες τεχνολογίες κτλ. Επανεστιάζουμε σε κοινωνικά ζητήματα, ε, στις υπηρεσίες κτλ. κτλ. Δηλαδή ποιοτικά θα εκτιμήσουμε που βρισκόμαστε το 2015 με τη Λευκή Βίβλο του 2011. Θα υπάρξει μια εφαρμοστική έκθεση που θα δημοσιευθεί με κάποιο τρόπο μέχρι τα τέλη του έτους. Απομένει να δούμε πόσο μεγάλη θα είναι η πολιτική όρεξη, για να το πω έτσι, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και πώς θα μεταξελιχθεί σε πλήρη πολιτική αξιολόγηση αρχές του επομένου έτους. Αυτό είναι το παρόν πλαίσιο και η διαδικασία έτσι όπως την έχουμε στο μυαλό μας. θα υπάρξει ιεράρχηση προτεραιοτήτων ανευθέτω χρόνο πάντα με βάση τη δική μας ανάλυση. Και ένα τελευταίο. Βεβαίως η Λευκή Βίβλος δεν είναι η μόνη δραστηριότητα ε, που προωθούμε στις μεταφορές. Υπάρχει Ενεργειακή Ένωση και το στρατηγικό πλαίσιο δράσης και πρόγραμμα που ε, είναι και πολλές οι πρωτοβουλίες που έχουν να κάνουν με τις μεταφορές, θα ακολουθήσει το ψηφιακό θεματολόγιο για την ψηφιακή αγορά. Όλα αυτά εντάσσονται και στην αναθεώρηση της Λευκής Βίβλου. Ευχαριστώ τελευταίος, αλλά όχι έσχατος, ο εισηγητής μας για τη Λευκή Βίβλο, κύριος Βιν Βαντεκάμπ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Τώρα θα μπορούσα να μπω στον πειρασμό να πω ότι θα συνοψίσω μισή ώρα χωρίς διερμηνία για όλα αυτά που ακούσαμε σήμερα. Αλλά δεν θα το κάνω, παρόλο που είναι μεγάλος ο πειρασμός. Και αυτή τη στιγμή στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα υπάρχει εσωτερική συζήτηση και διαβούλευση για το ΕΦΣΥ, για το Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων και θα πρέπει να πάω εκεί για να προστατεύσω τα χρήματα των μεταφορών. Αλλά ε, πραγματικά ήταν πολύτιμη ημέρα, ακούσαμε πάρα πολύ κόσμο και θέλω να ευχαριστήσω πολλούς και τη γραμματεία που ακούν και σημειώνουν. Εγώ έχω σημειώσει κάποιες προτεραιότητες, κάποια μοντέλα ε, κοινωνική κινητικότητα, αστικές κοινωνίες, ε, αυτοκίνητα κοινόχρηστα ε, και θέλω να ευχαριστήσω για όλες τις προτάσεις Συμφωνώ με τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έχουμε ακούσει πολλά σήμερα, συνδυάσαμε. Νομίζω στις 14 Απριλίου θα ε, δημοσιευθεί η έκθεση και θα σας τηρώ ενήμερους ε, και παρακαλώ να συνεισφέρετε. Θέλω να ευχαριστήσω όλους ιδιαίτερως τα μέλη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής που έδειξαν προθυμία να κοιτάξουν ε, στην έκθεση τους και αυτό το θέμα ε, σας εύχομαι καλό βράδυ σε όλους. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Έτσι, τα πολλά λόγια είναι φτώχεια, λέει μια παροιμία. Ευχαριστώ. Να σας πω τώρα τα διαδικαστικά. 13-14 Απριλίου θα έρθει η πρώτη έκθεση, προθεσμία για τις τροπολογίες 20 Απριλίου και ε, η Επιτροπή Μεταφορών θα αποφασίσει 28 Μαΐου ιδέα ολομέλεια τον Ιούλιο του 2015 Θέλω να σας ευχαριστήσω και το τελευταίο πάνελ ε, και τους ομιλητές και τους συμμετέχοντες, τη γραμματεία φυσικά που ε, βοήθησε και τους και τις διερμηνείς για την υπέρβαση ωραρίου. Ευχαριστώ και πάλι. Καλό σας βράδυ. Νομίζω ότι ήταν καλή η συζήτηση, εντατική, πάρα πολύ έντονη. Ακούσαμε όλα τα θέματα που απτύνονται της Λευκής Βίβλου. Καλό σας βράδυ και πάλι και ένα μεγάλο ευχαριστώ.